Μόλις είδαμε το σχέδιο νομοθετικής πρότασης για τα προσπέκτους και μετά είχαμε την εγγύηση καταθέσεων και βεβαίως το σχέδιο δράσης για την Ένωση και τη παράξης κατεξιοδότηση για την φερεγγιότητα. Προχωράμε σιγά σιγά λοιπόν προς την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης και βεβαίως το σχέδιο δράσης έχει ορίσει κάποια φιλόδοξα βήματα. Είναι λοιπόν επίκαιρη η συζήτησή μας και ε, έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ που με ξαναδεχτήκατε στην Επιτροπή σας. Έχουν περάσει έξι μήνες νομίζω από την τελευταία φορά και όπως είπε ο Ρομπέρτο μου πρόξενε εντύπωση το πόσα έχουν συμβεί. Όχι μόνο όσον αφορά την συνέχιση της υφιστάμενης νομοθεσίας αλλά και μια νέα ατζέντα για, τις, ε, για την Ένωση Χρηματαγορών και την Τραπεζική Ένωση. Και στο πλαίσιο όλων αυτών προσπάθησα να βρω μια ισορροπία μεταξύ ανάπτυξης και δημοσιονομικής σταθερότητας και πάντα έχω κατά νου μια ανησυχία για την έλλειψη θέσεων εργασίας και ανάπτυξης και την επιθυμία να στηρίξουμε τις μικρομεσαίες της Ευρώπης. Για να είμαι λοιπόν αναλογικός σε αυτά τα οποία κάνω. Προσπαθούμε να δώσουμε κάποια ρυθμιστική βεβαιότητα στις επιχειρήσεις και να έχουμε πάντα κατά νου τα συμφέροντα των καταναλωτών. Θα ήθελα να αναφέρω τώρα κάποια από τα τελευταία βασικά σημεία των τελευταίων μηνών, αλλά γνωρίζω βεβαίως την δύσκολη και τεχνική δουλειά που κάνουν τα μέλη της Επιτροπής σας κάθε μέρα, δουλειά η οποία βεβαίως δεν ε, δημιουργεί πάντα τίτλους στα ΜΜΕ αλλά εξηγεί το γιατί έχετε τέτοια φήμη στο Κοινοβούλιο και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την στήριξή σας και για τις προκλήσεις βεβαίως πάντα που παρουσιάζεται για εμένα. Λοιπόν, το προηγούμενο μήνα είχαμε μια καλή συζήτηση για το σχέδιο δράσης για την Ένωση των Κεφαλαίων Αγορών. Όπως ξέρετε, στόχος της είναι να συνδέσει πιο αποτελεσματικά τις αποταμιεύσεις με την ανάπτυξη παρουσιάζει μια σειρά μέτρων που είναι ευρύτατα και φιλόδοξα θα έλεγα όπως υποσχέθηκα δεν χάσαμε καθόλου χρόνο ξεκινήσαμε αμέσως την προηγούμενη φορά που συναντηθήκαμε εγώ αποκόμισα την εντύπωση πως είστε ανυπόμονοι και το ίδιο συμβαίνει και με μένα. Για να αυξηθεί λοιπόν ο δανεισμός στην ευρύτερη οικονομία καταθέσαμε ένα πακέτο μέτρων για να καταλήξουμε σε μια απλή και διάφανη διαδικασία τίτλοποίησης. Ο μηχανισμός του Λουξεμβούργου συμφωνήθηκε ότι θα αποτελέσει μια γενική προσέγγιση μέχρι τα Χριστούγεννα. Αυτό το ρυθμό χρειαζόμαστε και είμαι σίγουρος πως στην Επιτροπή σας θα αναλάβετε και εσείς την σκητάλη για να κινηθούμε γρήγορα προτείναμε μια τροποποίηση της νομοθεσίας για την φερεγγιότητα 2 για να μειωθεί ακριβώς ε, κατά το 1 τρίτο ο λόγος του δεσμευμένου κεφαλαίου καθώς το θεωρήσαμε ε, ότι αποτελεί πλέον ένα κομμάτι του ενεργητικού και έτσι θα μπορέσει να διοικηθεί ένα 3 εκατομμύριο ευρώ στις επενδύσεις αυτές. Επίσης, σύμφωνα με τα όσα ζήτησαν τα μέλη τη Επιτροπής σα και συγκεκριμένα ο κύριο Μπάλτς, ζητήσαμε να μα δοθούν στοιχεία για τους κανόνες για την σορευτική επίδραση που έχουν αυτοί οι κανόνες ε, και βεβαίως οι κανονισμοί τους οποίους έπρεπε να δημιουργήσουμε γρήγορα κατά τη διάρκεια της κρίσης θα μπορούσαν πράγματι να δημιουργήσουν κάποιες ε, ακούσιες συνέπειες και αυτό θα θέλαμε να εξετάσουμε. Χωρίς βέβαια να θίξουμε το συνολικό πλαίσιο. Σήμερα το πρωί ξεκινήσαμε μια νέα πρόταση για μια οδηγία για τα προσπέκτους, ένα καθεστώς πιο φτηνό, πιο απλό, τα προσπέκτους θα γίνουν πιο χρήσιμα και έτσι οι χώρες θα μπορέσουν να αποκτήσουν την επένδυση που χρειάζονται. Αυξάνουμε λοιπόν το ποσό που μπορεί να αντλήσει κανείς από τις αγορές της Ένωσης χωρίς προσπέξεις από 100.000 σε 500.000 ευρώ. Δημιουργείται ένα ειδικό καθεστώς για τις μικρότερες επιχειρήσεις που θα τους επιτρέψει να δημιουργήσουν απλούστερα προσπέκτους. Απλοποιείται η διαδικασία για επιχειρήσεις που αντλούν κεφάλαια για δεύτερη, τρίτη, τέταρτη φορά και εγκρίνουμε την διαδικασία για μεγάλες εταιρείες που πάνε συχνά στις αγορές δημιουργώντας ένα καθεστώς ε, ανάλογο για αυτές τις εταιρείες. Ελπίζω λοιπόν να μπορέσουμε να στηρίξουμε αυτές τις επιχειρήσεις που δίνουν όθηση στην ανάπτυξη στην Ευρώπη. Κατόπιν θα έχουμε μια πράσινη βιβλιογιά της οι υπηρεσίες Λιανικής ε, θα το δημοσιεύσουμε πριν τα Χριστούγεννα και εδώ πέρα όπως ξέρετε πραγματικά θέλω να δω τα πράγματα από τη σκοπιά του καταναλωτή, πώς θα έχουμε κάποια πιο απτά αποτελέσματα από την ανιαία αγορά. Βεβαίως οι επενδυτές Λιανικής είναι βασικό κομμάτι των όσων θέλουμε με την Ένωση των Κεφαλαίων Αγορών και θέλουμε να υπάρχει διαφάνεια, ανταγωνισμός, επιλογή και να χρησιμοποιήσουμε πλήρως την ψηφιακή τεχνολογία και ελπίζω η πράσινη βίβλος ε, να δώσει νέα όθηση σε αυτή τη συζήτηση. Παράλληλα, συνεχίσαμε με τις προσπάθειες μας να ενισχύσουμε την Τραπεζική Ένωση και να δούμε τι γίνεται με τον κίνδυνο. Εξακολουθούμε να ασκούμε πίεση σε όλα τα κρατημέλη για να εφαρμόσουν την συμφωνημένη νομοθεσία, να μεταφέρουν στο Εθνικό Δίκαιο την οδηγία περί λύσης ε, των τραπεζών και να κυρώσουν την ε, διακυβερνητική συμφωνία που καθορίζει τις συνεισφορές στο ενιαίο ταμείο διάσωσης ε, και για το τελευταίο αυτό σημείο μπορώ να πω πως ένας επαρκής αριθμός κρατών έχει κυρώσει την συμφωνία αυτή και έτσι μπορεί το Ταμείο αυτό να ξεκινήσει την λειτουργία του εγκαίρως όπως είχαν προβλέψει δηλαδή από πρώτης πρώτου. Την προηγούμενη εβδομάδα καταθέσαμε μία πρόταση για να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό σύστημα ασφάλισης ε, εγγύησης καταθέσεων. Ένα κομμάτι βεβαίως το οποίο πάντα θεωρούσαμε πως θα πρέπει να συνοδεύει την Τραπεζική Ένωση μαζί με τις ενιαίες εποπτικές αρχές. Είναι κομμάτι μιας ευρύτερης σειράς μέτρων που προανήγγειλε ο πρόεδρος Γιούνκερ για να εμβαθυνθεί η Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Η πρόταση είναι να φύγουμε από το τωρινό σύστημα εθνικών εγγυήσεων των καταθέσεων σε ένα σύστημα το οποίο θα εγγυάται τις καταθέσεις σε όλη την Τραπεζική Ένωση. Οι καταθέσεις είναι ήδη εγγυημένες μέχρι τα 100.000 ευρώ εάν χρεοκοπήσει μια τράπεζα και το πανευρωπαϊκό σύστημα που προτείνουμε σημαίνει πως οι τράπεζες θα προστατεύονται καλύτερα ε, από κάποια τοπικά σοκ. Έχουμε λοιπόν μια σταδιακή προσέγγιση σε κάθε βήμα της οποίας ε, οι καταθέτες θα έχουν τις ίδιες εγγυήσεις με τώρα. Προτείνουμε τώρα να εισαχθεί ένα, να εισαχθεί ένα σύστημα αντασφάλισης το 2017 για τρία χρόνια και μετά σταδιακά να αυξηθεί το κοντιλευτό με βάση την ε, συνασφάλιση μέχρι να υπάρξει μια πλήρης αμοιβιοποίηση μέχρι το 2024. Θέλουμε αυτό να μην κοστίσει στον τραπεζικό τομέα, οπότε οι συνεισφορές θα αφαιρούνται από τα όσα ούτως ή άλλως οφείλουν να πληρώσουν στα εθνικά συστήματα εγγύησεων οι τράπεζες. Έχουμε επίσης ε, φροντίσει να μην υπάρχει ο λεγόμενος ηθικός κίνδυνος. Παραδείγματο χάρη από το ταμείο αυτό δεν θα μπορεί κανείς να αντλεί κονδύλια εκτός αν έχει συνεισφέρει πλήρω το εθνικό σύστημα εγγύησης ε, καταθέσεων και κατά την πρώτη φάση δεν ε, θα μπορεί κανείς να αντλήσει κονδύλιο μέχρι να έχουν εκταμιευθεί όλα τα κονδύλια που υπάρχουν στο Εθνικό Σύστημα Καταθέσεων. Οπότε προσφέρει κάτι το οποίο δεν είναι δωρεάν και κανείς βεβαίω δεν παριστάνει πως η διαδικασία αυτή θα είναι εύκολη, αλλά θεωρώ πως ο μόνος τρόπος για να σημειώσουμε πρόοδο είναι να δοκιμάσουμε ε, ταυτόχρονα την μείωση και του κινδύνου και ταυτόχρονα να τον επομιστούμε τον κίνδυνο από κοινό. Ταυτόχρονα με αυτή την ε, πρόταση χάρηκα ιδιαίτερα για το ότι κατέληξαν οι διαπραγματεύσεις ε, για τα μέτρα εκείνα τα συγκριτικά καθώς ε, θα πρέπει όσοι κάνουν συγκριτικές αξιολογήσεις να έχουν μία άδεια και να υφίστανται κάποιαν αξιολόγηση. Έτσι θα αυξηθεί η εμπιστοσύνη στις ε, χρηματαγορές και θα ήθελα πάλι να ευχαριστήσω την Κόρα Φανίβεν Χόζεν και τους και για τη δουλειά που έκαναν. Τον προηγούμενο μήνα συμφωνήσαμε τον ε, κανονισμό για την ε, τυλοποίηση των δημοσιονομικών συνταγών για να αυξηθεί η διαφάνεια και η ασφάλεια στον σκιώδη τραπεζικό τομέα Κατόπιν είναι και σε συμφωνία με τα όσα έχουμε πει με τους G20. Και εδώ πέρα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Σόρου. Βεβαίω, δεν έχουμε ξεχάσει την προστασία των ε, καταναλωτών που έχει μεγάλη σημασία και είχαμε βέβαια και δύο θέματα τα οποία, στα οποία καταλήξαμε συμφωνία. Είχαμε το θέμα των ασφαλιών που εγκρίθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, την έκθεση Λάγκη και θα φροντίσουμε όσοι πουλάνε ασφάλεια να αντιλαμβάνονται τα προϊόντα που πουλάνε και όσοι αγοράζουν ασφάλεια ασφαλιστικά προϊόντα να έχουν τις πληροφορίες που χρειάζονται για να λάβουν μια απόφαση. Μετά έχουμε την οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών, η αναθεωρημένη, ε, που έχει ξεκινήσει επί κυρίου Ταγιάννη μας οδηγεί στις ψηφιακές ε, πληρωμές ε, και το τι γίνεται σε περίπτωση απώλειας μιας ε, κάρτας πληρωμών καθώς και κάποιες προδιαγραφές ασφαλεία που πρέπει να πληρούν όλοι οι πάροχοι τέτοιων υπηρεσιών. Αυτά βεβαίως τα σημαντικά δεν μας εμπόδισαν να λάβουμε και μια σειρά μέτρων, μια ομοβροντία θα έλεγα, μέτρων επίπεδου 2 Έχουμε εγκρίνει 32 μέχρι στιγμή και σκοπεύουμε να εγκρίνουμε άλλα 3 μέχρι το τέλος του έτους. Αυτά έτσι ως μια γενική εικόνα της δουλειάς ε, του δικού μου χαρτοφυλακίου. Θα έλεγα πως ε, κινούμαστε γρήγορα και είμαστε αρκετά φιλόδοξοι και πιστεύω πως έχουμε βρει μια καλή ισορροπία μεταξύ της ε, χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και στήριξης Τη ανάπτυξη και των θέσεων εργασία στην Ευρώπη. Όσο για μένα, εγώ θέλω να επιταχύνω το ρυθμό για να έχουμε απτά αποτελέσματα για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις ε, της Ευρώπης. Και αναμένω τώρα τη συζήτηση που θα έχουμε τώρα και στους επόμενους μήνες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you very... Σας ευχαριστώ πολύ. Jonathan. Και τώρα θα ξεκινήσουμε με τους ομιλητές μας. Πρώτος είναι ο κύριος Μπάλτσα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Χαίρομαι για τη σημερινή συζήτηση. Θα ήθελα να αφαιρθώ σε κάποια γενικότερα ζητήματα τα οποία έχουν νομίζω κάποια ιδιαίτερη σημασία. Η Κομισιόν είναι ο θεματοφύλακας των συνθήκων ε, και της ποιότητας της ε, νομοθεσίας και βεβαίως πρέπει να τηρεί και τις διαδικασίες. Και θα ήθελα να, μάνω, θα ήθελα να μάθω πώς υπάρχουν κράτη-μέλη τα οποία δεν έχουν ακόμα κυρώσει την οδηγία για την διάσωση των τραπεζών από το 2010. Πώς είναι δυνατόν κράτη-μέλη το, κύρωσαν την διακυβερνητική συμφωνία για το σχετικό ταμείο σήμερα, τελευταία στιγμή, ή να μην την έχουν κυρώσει ακόμα. Δεν θα έπρεπε η προτεραιότητα της Κομισιόν να είναι η εφαρμογή των υφισταμένων πριν προχωρήσετε στις περαιτέρω προτάσεις τις οποίες ε, ανακοινώσατε. Και δεν θα έπρεπε η θέληση των ε, συνομοθετών να παίξει έναν πιο σημαντικό ρόλο και να τηρούνται έτσι οι ημερομηνίε που έχουμε ορίσει για την αναθεώρηση της νομοθεσίας. Η Κομισιόν λέει πως ε, θα πρέπει να σπάσει ο κρίκος που συνδέει τραπεζικό και κρατικό κίνδυνο. Τώρα, αυτό το οποίο κάνετε μάλλον ε, αντικαθιστά τον ε, εθνικό φορολογούμενο με τον ευρωπαίο φορολογούμενο. Ή πώς θα επιτύχετε μια πραγματική μείωση του κινδύνου στον ε, τραπεζικό τομέα που δεν θα δώσει λανθασμένα κίνητρα στα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να σκεφτείτε τον πραγματικό κινδύνο να υπάρξει ένα ποσοτικό ελάχιστο στάνταρ για το έμπρε παραδείγματο χάρη. Θα ήθελα να μου πείτε την άποψή σας για αυτά. Ευχαριστώ. Well, thank you first of all for that. Σας ευχαριστώ πολύ καταρχήν για τα σχόλιά σας. Εγώ κατανοώ την απογοήτευσή σας για το χρόνο που χρειάστηκε ώστε να επικυρωθεί η νομοθεσία και ε, για το τι δεσμεύσεις τελικά ανέλαβαν τα κράτη. Ε, γι' αυτό και πέρυσι κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να μπορέσουμε να έχουμε διμερή επαφή με τα κρατημέλη, με τα κοφίν, με το Eurogroup, να τονίσουμε τακτικά δηλαδή την ανάγκη εφαρμογής σε σύγκριση με το που βρισκόμασταν ε, στις αρχές του έτους ε, για να μπορέσουμε να δούμε κατά πόσο όταν θα έχει ολοκληρωθεί η αυτή η μακρά πορεία, ε, αν ο κόσμος θα μπορούσε όντως να τα θέσει όλα αυτά σε εφαρμογή. Γι' αυτό το λόγο και... Γι' αυτό και... Ξεκινήσαμε διαδικασία κατά παράβαση και θα χρησιμοποιήσω σίγουρα κάθε εργαλείο που έχω στη διάθεσή μου για να συνεχίσω να πιέζω για αυτό το θέμα. Ε, το ποσοστό αυτό έχει τεθεί σε εφαρμογή μέχρι τη σημερινή προθεσμία, από τη σημερινή μάλλον προθεσμία, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να ασκείται πίεση μέχρι τελευταία στιγμή. Τώρα, για τις ευρύτερες σας παρατηρήσεις, για τη μείωση του κινδύνου και την θεμελιώδη σας ερώτηση που αφορά το κατά πόσο θα έπρεπε να έχουμε όλα αυτά τα μέτρα ολοκληρωμένα, εφαρμοσμένα πριν προτείνουμε οποιαδήποτε άλλα μέτρα. Καταρχήν, ναι, πιστεύω πως θα έχουμε το DRT και το DGST πλήρως εφαρμοσμένα πριν να υποβάλουμε νέες προτάσεις. Και σίγουρα πρέπει να αρχίσουν να ισχύουν νέα μέτρα, γιατί θα μας φάρουν και τα νέα μέτρα άλλο τόσο χρόνο. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να δομηθεί αυτή η πρόταση με αυτόν τον τρόπο που το κάναμε, δηλαδή ε, να ε, έχουμε μέτρα μείωσης του κινδύνου ταυτόχρονα με τα μέτρα της ε, αμοιβιοποίησης και πιστεύω πως ούτως ή άλλως θα προχωρήσουμε. Πιστεύω πως όλοι συμφωνούν πως χρειάζεται πρόοδος. Ο κόσμος έχει ερωτήσεις για το, τις φάσεις που θα περάσει. Αλλά νομίζω πως ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες που εσείς αναφέρατε είναι να προχωρήσουμε από κενού. Να εξασφαλίσουμε δηλαδή όλα τα μέτρα ώστε αυτά να προχωρήσουν μαζί τα παράλληλα με το πρόγραμμα για την εγγύηση των καταθέσεων. Ευχαριστώ, είναι Ναγκίλ. Ε, ευχαριστώ, καλώς ορίσατε, Επίτροπε η CMU φαίνεται η πιο φιλόδοξη χρηματοπιστωτική πρωτοβουλία από την ε, ΟΝΕ που ξεκίνησε το 1999, που θα μπορούσε να βοηθήσει στη χρηματοδότηση τη οικονομία. Πιστεύω λοιπόν πω θα μπορούσαμε να έχουμε συνολική υποστήριξη για αυτό το πακέτο, αλλά δεν είμαι βεβαία κατά πόσο αυτό θα συμβεί για το Συμβούλιο, για, τα πλευρά Συμβουλίου, γιατί αυτό έχει δείξει έλλειψη ευρωπαϊκή προσέγγιση από την αρχή των ε, μηνών, των τελευταίων μηνών και αυτό όχι επειδή εμποδίστηκαν τα κράτη-μέλη να κινηθούν. Μέχρι ότου λοιπόν δούμε ο πραγματικό αντίκτυπο δεν θα έχουμε πολλέ δυνατότητε να αντιμετωπίσουμε άλλε αναγκαίε μεταρρυθμίσει έτσι ώστε να επιτύχει η CMU. Είτε είναι το EDIS που είναι ε, ήδη επίμαχο, είτε είναι μεταρρυθμίσεις για την αφεργειότητα και κάτι ακόμα σε σχέση με αυτό που είπε ο Μπάλτς. Εσείς τι θα κάνετε ως Επιτροπή, ως ε, θεματοφύλακα των συνθήκων στους επόμενους μήνες ώστε να εξασφαλίσετε ότι οι τομείς όπως το CMU και άλλα θα γίνουν πραγματικότητα. Και η δεύτερη μου παρατήρηση αφορά το ότι το FTT ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι η τυπλοποίηση κάποιων ε, ε, ενυπόθηκων δανείων θα ξεκινούσε φέτο, ε, αυτή τη βδομάδα στη ΣΥΠΑ. Έχω λοιπόν την εντύπωση ότι δεν πήραμε κανένα δίδαγμα, ο μάλλον ο χρηματοπιστωτικό τομέα όσον αφορά τοξικά, προ... τοξικά προϊόντα. Και ναι, η τιτλοποίηση ίσως να είναι χρήσιμο δυνητικά εργαλείο για να προωθηθεί η οικονομία, αλλά αυτή είναι ανησυχητική εξέλιξη και ξέρω πως η πρόθεσή σας είναι να εξασφαλίσετε πως δεν θα συμβεί αυτό στην Ένωση. Αλλά υπάρχουν διάφορα σημεία που θέλω να μου διευκρινίσετε. Έχουμε περίπου 826 εκατομμύρια ευρώ σε τοξικά δάνεια από τα οποία βρίσκονται σε ευρωπαϊκές τράπεζες. Πώς θα εξασφαλίσουμε ότι όλα αυτά δεν θα τυπλοποιηθούν. Ε, και η πρότασή σας για ένα σύστημα εντοπισμού ε, ε, περιέχει κάποιους κινδύνους. Πώς θα εξασφαλίσουμε ότι οι επενδυτές θα μπορούν να βασίζονται στην σήμανση STS και ορισμένοι λένε ότι η δυσλοποίηση θα είναι επιτυχής μόνο εφόσον υπάρχει ισότιμο πεδίο για τα καλυμμένα ομόλογα που είναι αυτή τη στιγμή πολύ πιο ενδιαφέρουσα επιλογή για τις τράπεζες από ότι η τιτλοποίηση. Πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό που έχετε κάτι ετοιμάσει. Ευχαριστώ και ευχαριστώ για τη γενική υποστήριξη για την CMU. Για την ευρύτερη σας παρατήρηση για το Συμβούλιο και τη CMU, θεωρώ, θα έλεγα μάλλον, ότι ήταν καλή, αρκετή στήριξη για την CMU από το Συμβούλιο. Έχουν γεννηθεί πολύ γρήγορα για το τομέα της τυπλοποίησης, τον οποίο θα έχουν ολοκληρώσει σε μια-δυο εβδομάδες έδωσαν ισχυρή υποστήριξη και τα 28 κράτη-μέλη στην γενική προσέγγιση που ακολουθήσαμε και στην ε, καταβήμα προσέγγιση και καταστήσαμε σαφές ε, ποια ήταν τα στοιχεία αυτής ε, της προσέγγισης και εγώ τους είπα ότι θα είναι δική μου δουλειά να προχωρήσω έτσι και για, τις, ε, για το PDP κατά κάτι την απογοήτευσή σα. Δεν μπορέσαμε να προχωρήσουμε περισσότερο στη διάρκεια της Προεδρίας του Λουξεμβούργου, όπως γνωρίζετε. Ε, ήθελα εγώ, ξέρετε, να προχωρήσουμε και ελπίζω πως με την ε, ε, Ολλανδική Προεδρία θα τα καταφέρουμε κιόλας Πρέπει να μπορέσουμε να προοδεύσουμε και υπάρχουν στοιχεία που θα μας βοηθήσουν. Για τη τυπλοποίηση πιο σύντομα. Υπάρχουν συγκεκριμένες ανησυχίες και βέβαια αυτά θα λυθούν καθώς θα μελετούμε τις λεπτομέρειες του των προτάσεων στο Κοινοβούλιο για την ε, αυτοπιστοποίηση. Εγώ ήθελα να υπάρξει ένα σύστημα όπου οι εκδότες ε, τίτλων να αναλαμβάνουν και την ευθύνη για αυτό που κάνουν. Γιατί είδαμε τι έγινε με τις, ε, τους οργανισμούς ε, αξιολόγησης ε, της ικανότητα, ικανότητας, γιατί εκεί ανάλαβαν κινδύνους εταιρείε, οργανισμοί και μπόρεσαν να, να χρησιμοποιήσουν τρίτο μέρος για να δίνει αυτού του είδους την εξασφάλιση. Τώρα για τα εγγυημένα ομόλογα, covered bonds, ε, θα ξεκινήσουμε την επόμενη εβδομάδα ε, για να μπορέσουμε να εξηγήσουμε και ε, να εξετάσουμε ορισμένες από αυτές τις συσχετήσεις που εσείς αναφέρατε. Ευχαριστώ. Μπέρτ Λούκε. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε Λόρδε Χιλ. Έχω μια απλή ερώτηση για την Τραπεζική Ένωση για τον τρίτον πυλώνα και την εγγύηση των καταθέσεων. Θα συμφωνούσατε πως οι κίνδυνοι που υπάρχουν στον τραπεζικό τομέα της Ένωσης είναι ασύμετροι όσον αφορά την κατανομή τους και οπωσδήποτε το βάρος βρίσκεται στις χώρες του Νότου που βρίσκονται σε κρίση όσον αφορά και την εξάρτηση από κρατικό χρέος αλλά και από μη εξυπηρετούμενα δάνεια σε ιδιώτες. Βεβαίω κανείς δεν ξέρει το τι θα φέρει το μέλλον αλλά υποθέτουμε πως οι μελλοντικές πληρωμές σε, σε ένα τέτοιο σύστημα από γερμανική σκοπιά θα είναι μια καθαρή εισφορά προς όφελος ε, νότιο-ευρωπαϊκών κρατών. I think where ε, κοιτάξτε, εγώ θα έλεγα πως ε, πρώτα απ' όλα ο στόχος όλων αυτών των μεταρρυθμίσεων που υπάρχουν είναι να μειωθεί η πιθανότητα αποτυχίας πρώτα απ' όλα και άρα του να χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί το σύστημα εγγύησης καταθέσεων. Δεύτερον, έχετε δίκιο όταν τονίζετε το ότι υπάρχουν ε, διαφορετικά επίπεδα κινδύνου στις ευρωπαϊκές τράπεζες και αυτό το οποίο θέλουμε να αντιμετωπίσουμε μέσω μια σειρά μέτρων μεταξύ των οποίων και μέτρα μείωση του κινδύνου είναι να δούμε αυτά τα ζητήματα και να βρούμε κάποιους τρόπους μείωσης του κινδύνου και αντιμετώπισης αυτών των ζητημάτων. Και αυτά αναφέρονται στην ανακοίνωση που δημοσιεύσαμε μαζί με την νομοθετική πρόταση. Γεγονός είναι επίσης πως έτσι όπως έχουμε δημιουργήσει αυτό το σύστημα καθώς πηγαίνουμε από την αντασφάλιση στην συνασφάλιση μετά από τρία χρόνια είναι τότε το χρονικό σημείο στο οποίο θα υπάρχει κοινός κίνδυνος δηλαδή θα υπολογίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο ο κίνδυνος και όχι σε εθνικό και κατ' ουσίαν ο σταθμισμένος κίνδυνος για πιο ασφαλείς τράπεζες σημαίνει ότι θα πληρώνουν λιγότερο, ενώ οι πιο επισφαλείς τράπεζες θα πληρώνουν περισσότερο. Και έχουμε άρα άλλο ένα παράδειγμα του πώς είναι δυνατόν να αντιμετωπίσουμε κάποιες ανησυχίες που υπάρχουν, αλλά και να επιτύχουμε κάποια πρόοδο στον τρίτο πυλώνα της Τραπεζικής Ένωσης που πάντα υπήρχε. Έχουμε εποπτεία σε ευρωπαϊκή βάση, μια διάσωση σε ευρωπαϊκή βάση και βεβαίως πάντα θέλαμε να κάνουμε και εγγύηση καταθέσεων ευρωπαϊκή αλλά βεβαίω πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για να μας ακολουθήσει και η κοινή γνώμη γι' αυτό ακριβώς νομίζω πως έχουμε ένα ισορροπημένο πακέτο με διάφορες φάσεις ε, για να υπάρχει ακριβώς αυτή η διασφάλιση του κοινού πριν περάσουμε στην επόμενη φάση. Νομίζω πως έχω ακόμα χρόνο, ναι. Α, ε, ναι, αλλά γρήγορα άμα θέλετε απάντηση. Να θέσω το ερώτημα που δεν απαντήσετε. Πράγματι προσπαθείτε να μειώσετε τον κίνδυνο, αλλά προφανώς πιστεύετε ότι υπάρχουν κίνδυνοι, αλλιώς δεν θα χρειαζόταν ένα τέτοιο σύστημα. Το ερώτημά μου είναι, ήταν δεν αναμένεται μια καθαρή εισφορά από το γερμανικό τραπεζικό σύστημα, τραπεζικό σύστημα άλλων χωρών. Κοιτάξτε, μα, ο στόχος εδώ πέρα είναι να γίνει το όλο σύστημα πιο ασφαλές. Οπότε δεν είναι σωστό να λέμε πως ο στόχος ε, εδώ πέρα η συνέπεια θα είναι να δημιουργηθεί μία ένωση η οποία θα σημαίνει μεταφόρα κονδυλίων, το οποίο ξέρω πως ανησυχεί πολύ κόσμο. Νομίζω πως μπορούμε να αποφύγουμε τις ανησυχίες που έχετε εσείς ε, και άλλοι και νομίζω πως με την προσέγγιση που έχουμε θα το αποφύγουμε. Σας ευχαριστώ. Πολύ σκόπιμο θα είναι να κάνουμε ένα ίδιο αριθμό κρατών μελών από το βορρά και τον νότο για να μην λέει κανείς ότι κάνουμε διακρίσεις. Ο κύριος Τόρμπας, ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ Επίτροπε που είστε και πάλι εδώ. Η Ένωση των Κεφαλαιογορών είναι κάτι που σε μεγάλο βαθμό καλωσορίζουμε και που θέλουμε να ε, ε, γίνει. Ωστόσο έχουμε μια πολύ μεγάλη ανησυχία και γιατί υπάρχει μια τάση που μπορούμε να δούμε σε όλα τα κράτη-μέλη. Στα πιο μεγάλα και τα πιο, με τη μεγαλύτερη επιρροή έχουμε ε, κάποιους ε, ε, ε ε, συγκεκριμένου όρου και συνθήκε που ισχύουν που δεν λαμβάνουν πάντοτε υπόψη την κατάσταση στην περιφέρεια. Μπορεί δηλαδή να υπάρχει ο κίνδυνος ασυμμετρικών σοκ ή κυμάτων όπως λέγονται σε αυτό το πλαίσιο. Το διαβάζω την πρόταση για την Ένωση των Κεφαλαγορών. Φοβούμαι μήπως ε, διαπράξουμε τέτοιου είδους φάλματα άλλη μια φορά Δεν είναι μυστικό ότι έχουμε δύο διαφορετικά κέντρα, Φραγκφούρτη και Λονδίνο. Με τη βοήθεια κάποιων φίλων σας στο που μπορεί να ξεφορτωθούμε το Λονδίνο και έτσι να απλοποιηθεί το πρόβλημα αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι εύκολο να ακολουθήσει κανείς να φτιάξει νομοθεσία για να προσαρμόσει ε, μόνο τους όρους στις ανάγκες αυτών των οικονομικών κέντρων. Εσείς μπορείτε να με καθησυχάσετε ότι κάνετε το σωστό παρά το ότι έχετε φίλους και γνωστούς από συγκεκριμένο χώρο. Ελπίζω ότι μπορώ να σας καθησυχάσω. Βασικά με λόγια αλλά και κυρίως με πράξεις. Η αλήθεια είναι ότι θα γνωρίζετε πως ε, θα πρέπει κανείς να κρίνει από το πώς προσεγγίζει τα πράγματα. Όσον αφορά τα όσα είπατε, ξεκινώ με το σημείο σας ότι θα πρέπει πάντοτε να προσπαθήσει κανείς να έχει μια προσέγγιση που να είναι όσο γίνεται πιο αντίστοιχη, πιο, πιο αναλογική με την εκάστοτε περίπτωση και να αποφεύγει τις ομοιόμορφες λύσεις, όχι μόνο στον τομέα της ε, Ένωσης των Κεφαλαγορών ή των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Αν δούμε δηλαδή την αναθεώρηση της CRR, δηλαδή των ε, κεφαλαικών απαιτήσεων, την οδηγία των κεφαλαικών απαιτήσεων. Ένα από τους λόγου και την υποχρέωση επανεξέταση αυτή είναι ε, ότι ε, όντω προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε την επιρροή αυτής της οδηγίας στο δανεισμό και κυρίω δανεισμό προς τι ΜΜΕ. τι μικρομεσαίε δηλαδή. Θα ήταν ένα στοιχείο αναλογικότητας ε, όσον αφορά ολόκληρη την προσέγγιση προς την Ένωση των Κεφαλαγορών θα έπρεπε ίσως να το κάνουμε ξεκινώντας με μια γνήσια διαβούλευση. Δεν ξεκίνησα λοιπόν με ένα πλάνο το οποίο θα, ήθελα, θα προσπαθήσω να επιβάλλω εγώ στους άλλους, αλλά ρώτησα πολλούς να μου πούν τι θεωρούν ότι είναι εμπόδιο και να μου υποβάλουν προτάσεις. Ε, για το πώς να προχωρήσουμε. Και για τα εγκείμενα ομόλογα γνωρίζω πάρα πολύ καλά πόσο σημαντικά είναι αυτά τα, τα, τα ομόλογα σε κάποιες αγορές ενώ σε άλλες όχι. Για μένα λοιπόν το θέμα δεν είναι πώς μπορώ να επιβάλλω κάποιο εναρμονισμένο σχέδιο και να διαταράξω τις αγορές που λειτουργούν σωστά. Το πρόγραμμά μου είναι το να κάνω, να δω τι λειτουργεί καλά, αν μπορώ από εκεί να αποκομίσω κάποια διδάγματα, αν μπορούμε να τα μοιραστούμε ευρύτερα στην υπόλοιπη Ευρώπη, ώστε και άλλοι να ωφεληθούν με τον ίδιο τρόπο. Αυτά ε, θέλω να προσπαθήσω να κάνω και εν μέρη γι' αυτό και έχουμε κάνει έκκληση για ε, μαρτυρίες, για αποδείξεις, ώστε να δούμε πόσο αποτελεσματικά είναι αυτό που κάνουμε και να προσπαθήσουμε να, δούμε, να είμαστε μάλλον όσο γίνεται πιο ισορροπημένοι και ευέλικτοι. γιατί πρόκειται για ένα project για τους 28, ε, ένα project κλασικό για την ενιαία ώρα, ε, η κεφαλαία και, και ώρα. Και γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό να έχουμε αυτές τις χώρες που δεν έχουν τόσο αναπτυγμένη κεφαλαγορά υπόψη και να επεκτείνουμε τα ωφέλη αυτού του συστήματος σε όλους όσο γίνεται. Ευχαριστώ. Καλώ ήρθατε κύριε Επίτροπε. Κανονικά σας ρωτάω πάντα για την Ένωση των Χρηματαγορών αλλά σήμερα θα το έβρισκα κάπως βάρωτο, οπότε θα ξεκινήσω με τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στις ε, τράπεζες. Γνωρίζουμε πως η σχετική τράπεζα είναι στο κοινοβούλιο, γιατί βεβαίως ε, το πρόβλημα είναι ότι οι μεγάλες ε, ομάδες αυτή τη στιγμή είναι σε ένα κονκλάβιο και περιμένουμε να βγει καπνός δεν ξέρω, μπορεί αυτό να ήταν και η μυρωδιά που μυρίσαμε όταν μπήκαμε στην αίθουσα. Λοιπόν, είπατε όμως πως ε, ίσως αποσυρθεί η πρόταση αν δεν υπάρξει συμφωνία. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι μέχρι πότε θα περιμένετε. Εγώ δεν θα ήθελα να αποσυρθεί η πρότασή σας, ήταν πάρα πολύ καλή και καλό θα ήταν να μην εξευτελιστούμε εδώ πέρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να μην γίνει τελικά αυτή η μεταρρύθμιση. δεύτερο για την εγγύηση των καταθέσεων. Εμένα είναι αυτονόητο ότι χρειαζόμαστε κάτι τέτοιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίω συμφωνώ με κάποιες επιφυλάξεις ε, προλαλισσάντων ότι θα πρέπει να υπάρξει μια διασπορά του κινδύνου αλλά αυτό το οποίο με εξέπληξε ήταν ότι ο κύριος Γιούνκερ ανακοίνωσε πως θα εξαιρέσει τις, ε, τα συνεταιριστικά ταμιευτήρια και μετά είπε ότι δεν θα το κάνει κάτι τέτοιο. Ε, τι συμβαίνει, υπάρχει πρόβλημα επικοινωνίας εντός της ε, Κομισιόν, πώς εξηγούνται αυτά τα φαινόμενα. Τέλος, ένα ερώτημα που ίσως σας φαίνεται κάπως εξωτικό αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί Βεβαίως έχουμε τα γεγονότα στο Παρίσι. Εγώ ρώτησα Κομισιόν Κοινοβούλιο, Συμβούλιο και Κομισιόν για το εάν σκοπεύουν, αν έχουν εφαρμοστεί τα μέτρα προτείνει ο ΙΕ, πάγωμα λογαριασμών και τα λοιπά. Το Συμβούλιο μου ότι δεν μπορεί να απαντήσει και η Κομισιόν μου είπε ότι επίσης δεν μπορεί να απαντήσει και δεν είναι αρμόδια. Ναι, ναι, ικανοποιείται και σε αυτές οι απαντήσεις. Θα ήθελα λοιπόν, εάν μπορείτε, να μου πληροφορήσετε εσείς για το τι γίνεται. Μακρηγορήσατε, συνάδελφε, λέει ο πρόεδρος. Ε, Κύριο Χίλ, ευχαριστώ. Τρεις ερωτήσεις ε, μου υποβάλλατε σε ό,τι αφορά ε, τις ε, μεταρρυθμίσεις στις τράπεζες. Νομίζω ότι επί αναφέρω τη θέση μας ως Επιτροπή ότι δηλαδή θεωρούμε ότι για τις τράπεζες ε, too big to fail είναι ένα ζήτημα που καλό θα ήταν να αντιμετωπίσουμε μέσω της ε, προτάσεις μας ε, PSR. Το Συμβούλιο έχει συμφωνήσει με τη γενική προσέγγιση. Οπότε θεωρώ ότι αυτό αποτελεί μια βάση για να προχωρήσει αυτή η πρόταση. ανέκαθεν ναι, έλπιζα, δεν είναι εύκολο και το γνωρίζω. Να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Κοινοβούλιο για να μπορέσει να προχωρήσει η πρόταση. Για αυτό το σχέδιο εγγύσεων να επαναλάβω αυτό που ήδη έχω πει. Θεωρώ ότι πρόκειται και για τα δύο. Δεν μπορώ να δεχθώ δηλαδή ένα αξίωμα που λέει ότι η πρόταση αυτή ουσιαστικά έχει να κάνει με επιμερισμό κινδύνων απλά και όχι με τριασμό αυτών, διότι σκοπίμως διατυπώσαμε μια πρόταση που στόχο έχει το μετριασμό και τον επιμερισμό βέβαια των κινδύνων. Αυτή νομίζω είναι η ορθή προσέγγιση και η προσωπική μου άποψη είναι ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα μετριασμού των κινδύνων. Και το τρίτο σας σημείο για τις τοπικές ε, τράπεζες, ε, τις αποταμιστικές παρκάς. Νομίζω ότι και ο Πρόεδρος και οι υπόλοιποι επίτροποι έχουμε ε, ξεκαθαρίσει ότι θα πρέπει αυτό το ταμείο, μάλλον αυτό το σχέδιο στο να καταθέσω να καλύπτει όλες τις τράπεζες, λαμβάνοντα υπόψη τις ιδιαιτερότητε των διαφόρων ε, τραπεζικών μοντέλων, ιδίω ε, για τι ε, Sparkassen στη Γερμανία και άλλε αντίστοιχε περιπτώσει σε άλλε χώρε. Όλα αυτά θα τα μελετήσουμε όσο θα διατυπώνουμε τι συγκεκριμένε μα προτάσει. Για το τελευταίο που με ρωτήσατε, αδυνατό να σας δώσω μια συγκεκριμένη απάντηση, αλλά μπορώ να πω το εξής. Με τα χρηματοοικονομικά προϊόντα, εν γέννη, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να αποφύγουμε τα παραθυράκια που υπάρχουν ε, ε, και έτσι μπορούν να τα εκμεταλλεύονται αυτοί που θέλουν να μας κάνουν κακό να εκμεταλλεύονται και να ασφάλειας και να χρηματοδοτούν την τρομοκρατία. Αυτά τα ζητήματα πρέπει να μας απασχολήσουν πολύ προσεκτικά, αλλά πρέπει να υιοθετήσουμε μια ισορροπημένη άποψη για να μπορέσουμε να κάνουμε το σύστημα λίγο πιο στεγανό όσο μπορούμε. Ο πρόεδρος, δύο λεπτά θα δίνω πλέον ε, στον κάθε συνάδελφο Σβέν Γκίγκολτ. Καλώς ήρθατε. Καλώ ήρθατε κύριε Επιτροπέ. Ενώ καθόμαστε εμείς εδώ πέρα στο Παρίσι έχουμε διαπραγματεύσει για το κλίμα. Πρέπει λοιπόν και η οικονομία να συνεισφέρει στο πρασίνισμα. Αναφερθήκατε στην Ένωση Κεφαλαίου Αγορών στο γεγονό αυτό και έχω δύο ερωτήσεις. Πρώτον, στην ΠΡΙΠΣ συμφωνήσαμε πως οι βιώσιμες επενδύσεις και εφόρες επενδύσεις ε, θα είναι αντικείμενο πληροφόρησης των πολιτών αλλά οι υπηρεσίες σας δεν έχουν ακόμα δώσει την ε, αναγκαία εντολή για τις τεχνικές ε, προδιαγραφές Επί τη ευκαιρία λοιπόν της διάσκεψης για το κλίμα μπορείτε να μας διαβεβαιώσετε ότι θα εφαρμόσετε τους κανόνες που έχουμε συμφωνήσει και να δώσετε την ανάλογη εντολή στην ΕΣΜΑ για να υπάρχουν πληροφορίες για φόρες επενδύσεις στους πολίτες. Δεύτερον, για το θέμα της εγγύησης των καταθέσεων πρέπει πρώτα απ' όλα να πω πως συμφωνούμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα κοινό σύστημα που θα δημιουργεί την ίδια εμπιστοσύνη παντού. Οπότε υποστηρίζουμε την αρχή ενός συστήματος αντασφάλιση. Αυτό το οποίο δεν μπορούμε να στηρίξουμε είναι το τελευταίο κομμάτι της πρότασή σα να υπάρχει ένα κοινό ταμείο. Γιατί με ένα κοινό ταμείο θα καταστραφεί θα καταστραφούν τα συστήματα εκείνα τα οποία απαιτούνται σε κάποια κρατημέλη και στη Γερμανία για να στραφεί ο τραπεζικός τομέας στην πραγματική οικονομία. Και η γεγονό είναι πως ο πρόεδρος Γιούνκερ μας διαβεβαίωσε στις 8 Οκτωβρίου πως τα συστήματα αυτά δεν θα τα αγγίξουμε, έτσι είπε. Ε, τι γίνεται λοιπόν όταν ο πρόεδρος λέει ότι δεν θα τα αγγίξουμε και εσείς τώρα προτείνετε κάτι το οποίο είναι ένα ενιαίο ταμείο. Υπάρχει πως σας είναι νοησία εντός um, Για το πρώτο σημείο. Βιωσιμότητα, τρίψ. Πρώτα απ' όλα να σας πω ευρύτερα μιλώντας ότι με την Ένωση Κεφαλαίου Αγορών είναι πολύ σημαντικό να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε ένα μακροπρόθεσμο πλαίσιο. Και φυσικά γίνονται διάφορες συζητήσεις, φαντάζομαι ότι γνωρίζετε πιο πολλά από ότι εγώ, για το τι συζητείτε και στο ESRB και στο EFSB και σε εθνικό επίπεδο για όλα αυτά τα ζητήματα που άπτονται της βιωσιμότητας και των χρηματοοικονομικών κανονισμών. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να τα παρακολουθούμε και να τα προσέχουμε όλα αυτά και στο πλαίσιο της Ένωσης Κεφαλαίου Αγορών έχουμε τα πράσινα ομόλογα, green bonds, ένα θέμα που το έχουμε θέσει και το ε, εξετάζουμε. Τα το πρέπει. Ε, το ενδιαφέρον σας το γνωρίζω για το θέμα. Το έχω συζητήσει και με τις υπηρεσίες μου και θα σκεφτώ αυτά που είπατε και ευχαρίστως να το ξανασυζητήσουμε ακόμη περιττέρω για να ε, πάρουμε τώρα τη συμβουλή της ΕΣΜΑ, νομίζω ότι είναι δυνατόν αυτό. Θα συνεχίσω τις συζητήσει μου και τις επαφές μου και σύντομα θα σας ενημερώσω για το πώς θα προχωρήσουμε. Σε ό,τι αφορά τώρα την εγγύηση των καταθέσεων, εγώ σας εξέθεσα τη θέση του Σώματος των Επιτρόπων και της Προέδρου τη Επιτροπής. Νομίζω ότι και ελπίζω να αντιλαμβάνεστε και εσείς και οι υπόλοιποι ότι αυτό το οποίο πιστεύουμε είναι όλες οι τράπεζες καταρχήν να καλύπτονται, αλλά όπως είπε ο Πρόεδρος, έχουμε επίγνωση, πλήρη επίγνωση του συγκεκριμένου μοντέλου αυτών των ε, μηχανισμών ε, προστασίας επενδυτών. Το έχω συζητήσει και με αυτά τα ταμιευτήρια και με άλλες εντρικές τράπεζες και νομίζω είπε και ο πρόεδρος τη Ευρωπαϊκή πρέπει να εργαστούμε κατά τρόπον ώστε να σεβόμαστε τα μοντέλα αυτά, αλλά και να κάνουμε πρόοδο στο μέτωπο τη της των καταθέσεων. Ευχαριστώ, πρόεδρος. Τον Στίβεν Ουλφ δεν τον βλέπω. Επομένω. ο κύριος Άνεμαντς Ευχαριστώ. Άρα 10 λεπτά εγώ έχω. Eh, Θέλω να σα κάνω κάποιε ερωτήσει σε σχέση με το σύστημα εγγύηση ε, καταθέσεων. λοιπόν, Οπότε φαίνεται πως έτσι όπως έχουν τα πράγματα στην Νότια Ευρώπη η εγγύηση θα είναι κάτι το σχετικό. Υπάρχει λοιπόν αυτή η ωραία αρχή της εγγύησης, της ευρωπαϊκής, στην οποία βεβαίως έρχονται τώρα δύο άνθρωποι οι οποίοι μάλλον θα πλήξουν την όλη διαδικασία. Ο κ. Κάμερον απέστειλε μία επιστολή στον κύριο Τούσκο που υπάρχει μία παράγραφος που μιλάει για το ότι υπάρχει πάνω από ένα νόμισμα και πρέπει ανάλογα να κινηθεί και η διακυβέρνηση και δεν πρέπει να υπάρχει διακριτική μεταχείριση ε, των χωρών που είναι εκτός της ζώνης του ευρώ ότι θα πρέπει οι εισφορές τους να είναι εθελοντικές και δεν θα είναι δυνατόν να είναι υπεύθυνοι οι δικοί του φορολογούμενοι για τη σταθερότητα της Ευρωζώνης. Πώς συμβάζεται αυτό το οποίο μας είπατε με τις αρχές που ανέπτυξε ο κύριος Κάμερον, ο πρωθυπουργός σας. Και βεβαίως ο δεύτερος από την άλλη πλευρά είναι ο κύριος Σόιμπλε ο οποίος φοβάται, όπως και ο κύριος Λούκε, φοβάται πως θα έχουμε μία ένωση μεταφορών δημοσιονομικών διαβιβάσεων. Ναι, νομίζω προφανές ότι θα συμβεί αυτό. Πώς ε, συμβιβάζονται αυτά με τα όσα ωραία μας είπατε. Well, I think I Να αρχίσω πιο ευγενικά, γιατί προέρχομαι από μια βόρεια χώρα και να πω ότι και οι χώρες του Βορρά έχουν προβλήματα με τράπεζες που ε, καταραίουν ή αντιμετωπίζουν προβλήματα. Δεν είναι ένα φαινόμενο που το βιώνει μόνο ένα κομμάτι ε, χωρών. Απλά είχετε ένα τόνο στις ε, παρατηρήσεις σας ε, σαν να φαίνεται ότι είναι ένα πρόβλημα μοναδικό αλλά το έχω δει εγώ από πρώτο χέρι στη χώρα μου τα προβλήματα που προκύπτουν όταν τα βρίσκουν σκούρα οι τράπεζες. Και φαντάζομαι ότι μπορούμε να βρούμε ανάλογα παραδείγματα σε όλες τις χώρες μέλη. <clears throat> και μιλάω και για τράπεζες που λειτουργούν με βάση το συντεριστικό μοντέλο. Σε ό,τι αφορά το σχόλιο σας, Δεν ξέρω αν κατενόσα πλήρω τι εννοούσατε με την σχέση, τη διασύνδεση, τη συσχέτιση μάλλον που κάνετε μεταξύ Τραπεζικής Ένωσης και την επιστολή του κυρίου Κάμερον στον πρόεδρο Τούσκ. Δεν ξέρω τι θέλετε να, πού θέλετε να καταλήξετε. Ευρώπη πολλών νομισμάτων κτλ. Σε ό,τι αφορά την Τραπεζική Ένωση, Είναι σαφέ ότι πρόκειται για κάτι που αφορά τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης. Αλλά είναι και ανοιχτή για οποιοδήποτε άλλο κράτος θέλει να προσχωρήσει. Είναι μια απόφαση που θα πρέπει να αντιλάβει οποιοδήποτε κράτος που δεν ανήκει στην Ευρωζώνη υπό το φως όλων των ε, περιστάσεων και σε ό,τι αφορά το, το πρόγραμμα εγγύησης καταθέσεων να μην επανέλθω σε αυτά που είπα πριν δηλαδή ότι θέλουμε να έχουμε ένα σύστημα που θα δυναμώνει τις τράπεζες όλη την Ευρώπη γιατί αυτό είναι το λογικό Γιατί από σοκ μικρά ή μεγάλα ή μικρών ή μεγάλων τραπεζών όλοι θα υποφέρουμε. Ενώ με αυτό το σύστημα θα θωρακίσουμε καλύτερα τα κράτη-μέλη στα οποία ενδεχομένως συμβούν αυτά τα σοκ. Thank you. Σας ευχαριστώ. Ο Μάρκος Φέρμπερ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Δύο σύντομα ερωτήματα. Πρώτον, πριν από κάνα χρόνο στην ακρόασή σας ένα συνάδελφος σας ρώτησε αν θα κάνετε προτάσεις ε, για αλλαγή του συστήματος εγγύησης καταθέσεων. Τότε μας είπατε ότι όπως προβλέπετε στην οδηγία θα υποβάλλετε το 2019 μία έκθεση για την εφαρμογή του συστήματος. Τι σας παρακίνησε μέσα σε ένα χρόνο να αλλάξετε τελείως ε, στάση και να προτείνετε ένα πανευρωπαϊκό τέτοιο σύστημα. Δεύτερον, όσο και αν ε, αγαπάμε την ε, Ένωση των χρηματαγορών οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα εξαρτώνται πάντα από πιστώσεις. Και βλέπουμε παραδείγμα του χάρη πως εδώ πέρα η Κομισιόν ε, θα πρέπει να λάβει υπόψη της αρχής της αναλογικότητας στο πλαίσιο της οδηγίας για την ε, φερεγγιότητα, το ίδιο και στο usage και τα MIFID 2. Και θα ήθελα λοιπόν να μου απαντήσετε στο ερώτημα. Τι θα κάνουν ειδικά τα μικρότερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όσον αφορά την διασφάλιση της χρηματοδότησης. Ευχαριστώ. Well, first of all, on the, um... Λοιπόν, για το πρώτο σημείο που είπατε. Υπάρχουν ε, δύο βασικά, δύο πράγματα που θα έλεγα Πρώτον, η έκθεση των πέντε προέδρων δεν είχε τότε δημοσιευτεί. Ήμουν εδώ μαζί σας ε, μόλις πριν από ένα χρόνο. Μοιάζει να έχει περάσει μεγαλύτερο διάστημα. Οπότε, το ένα στοιχείο είναι αυτό. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο έχει αλλάξει και νομίζω πως ταιριάζει με τη γενικότερη προσέγγιση που προσπαθώ να έχω και γενικότερα προσέγγιση προσπαθώ να έχω. Δηλαδή, αν είναι να επιτευχθεί η πρόοδος σε κάποια ζητήματα, πρέπει να δούμε το ζήτημα τη εμπιστοσύνη, η οποία νομίζω έχει διαραγεί με διάφορους τρόπους μεταξύ διαφόρων κρατών μελών. Και για να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη θα πρέπει να κινούμαστε σταδιακά να μην γίνουν όλα με τιμία να δώσουμε κατευθύνσεις αλλά να μην προχωρήσουμε μέχρι να σημειωθεί η πρόοδος. Αυτό έγινε με την Ένωση των Χρηματαγορών και το σύστημα εγγύησης των καταθέσεων. Διαφορετική πρόταση οπωσδήποτε από αυτή η οποία έγινε το 2012 όταν πηγαίναμε κατευθείαν σε αμοιβιοποίηση οπωσδήποτε ε, προσπαθούμε να προχωρήσουμε σταδιακά να δούμε κάποιες από τις ανησυχίες που υπάρχουν και να υπάρξει κάποιο περιθώριο για την οικοδόμηση αυτής της εμπιστοσύνης για το άλλο σημαντικό θέμα για τα δάνεια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πώς θα τις ενθαρρύνουμε. Η απάντηση νομίζω είναι μέσω μιας σειράς μέτρων. Συμφωνώ με αυτό το οποίο είπατε πως η απάντηση δεν είναι μόνο η ένωση των κεφαλαίων και θα πρέπει πράγματι να υπάρχουν διαφορετικές ε, επιλογές με τις διάφορες πληροφορίες ε, για την πίστη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το θέμα λοιπόν του πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τις ε, τράπεζες, το παραδοσιακό μοντέλο και πάλι νομίζω πως μπορουμε να βοηθησουμε τις τραπεζες στο παραδοσιακο μοντελο και παλι νομιζω πως Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Μία μπορεί να είναι παραδείγματο χάρη η πρόταση για την τιτλοποίηση, οπότε μπορούν να ελαφρύνουν του ισολογισμού του οι τράπεζε και να δανείσουν απευθεία, ε, κάτι το οποίο στηρίζουν πολλέ χώρε ε, και η Γερμανία. Αλλά επίση συμφωνώ πω το να προσπαθούμε να βάλουμε το θέμα της αναλογικότητας ε, στις κεφαλαϊκές απαιτήσει, ε, να περιμένουμε επίσης ε, και την διαβούλευση την οποία έχουμε ξεκινήσει. Και να δούμε εάν πραγματικά αυτά τα οποία κάνουμε, η νομοθεσία μας έχει το αποτέλεσμα που θέλουμε για τον δανεισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ευχαριστώ, Ρενάτο Σόρου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα να ξέρω την γνώμη του Λόρδου για το σημείο που θα συζητήσουμε τις επόμενες ώρες αυτήν την Επιτροπή, δηλαδή την εισαγωγή του παράγοντα κινδύνου, risk factor, στις, ε, στις ε, κρατικές επιδοτήσεις και στους ε, τραπεζικούς ισολογισμούς. Από τη μια πλευρά οι μεσογειακές χώρες έχουν υποφέρει από μια λαθασμένη πολιτική υπερβολικής λιτότητας μέχρι την πρόσφατη άνοιγμα της ευελιξίας Ε, βέβαια θα έπρεπε να οδηγηθούμε σε, μια κατάσταση κανονικά μεγαλύτερη σταθερότητας. Ε, ε, τώρα, εάν εισαχθεί μια, ένα ακόμα, ένα ακόμα Λίθος, σε μια ακόμα απόσπαση των πόρων από τις μεμονωμένες χώρες που έχουν ανάγκη από μεγαλύτερη ανάπτυξη προς μια διαδικασία σύγκλησης, διαδικασία ίσως προς άλλες χώρες που έχουν, χώρες μάλλον που έχουν λιγότερες ανάγκες ή μήπω κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε πολύ σοβαρή οικονομική αστάθεια την οποία σίγουρα ε, δεν έχουμε αξιολογήσει υπαρκώ. Εγώ θεωρώ πω είναι επικίνδυνες αυτές οι προτάσεις που, που και που προκύπτουν στα διάφορα ντοσιέ και που τελικά στοχεύουν στο να δυναμετήσουν τη σύγκληση των οικονομικών και τους ισολογισμούς των χρηματοπιστωτικών συστημάτων των διαφόρων χωρών. Ευχαριστώ. Um, I think first of all that the... Πιστεύω καταρχήν ότι η παρατήρησή σας για το γεγονός ότι χρειάζεται να είμαστε ευαίσθητοι στην κινδύνου οικονομικής σταθερότητας και μήπως ε, μετακινηθούμε πάρα πολύ γρήγορα χωρίς ε, να το έχουμε αρκετά κουράσει και σκεφτεί. Νομίζω πως αυτό έχετε δίκιο. Και γι' αυτό το λόγο οι ευρύτερες διεθνείς συζητήσεις που γίνονται ε, είναι λογικό για μας να μας κάνουν να το σκεφτούμε και να το σκεφτούμε και σε ευρύτερο διεθνές πλαίσιο, όχι δηλαδή μόνο εντός Ένωσης αλλά και εντός Ένωσης και άλλων δικαιοδοσιών, διότι αν κάποιος ε, κάνει λάθος, οι συνέπειες με τον τρόπο που εσείς εκθέσατε, οι συνέπειες ενός τέτοιου λάθους θα ήταν τεράστιες. Τούτου τελευταίου νομίζω πως αυτό που είπαμε και με κάπως ισορροπημένο τρόπο είναι ότι το ε, βήμα της κάλυψης του κινδύνου και είπαμε στην ανακοίνωση που δημοσιεύσαμε μαζί με το σχέδιο εγγύησης καταθέσεων, το, το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Εγγύησης Καταθέσεων, ότι θα μπορούσαμε να εξετάσουμε, θα έπρεπε μάλλον να εξετάσουμε την έκθεση που έχουν οι διάφορες τράπεζες απέναντι στον κρατικό κίνδυνο, στην ίδια του τη χώρα δηλαδή. Είναι ένα τομέα όπου πρέπει νομίζω να δουλέψουμε περισσότερο, διότι υπάρχει ένα θέμα εκεί ε, για το οποίο θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Με τρόπο όμως ώστε να μην απειληθεί η οικονομική σταθερότητα. Και αυτό και πρόκειται να κάνουμε στην επόμενη ακριβώ περίοδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Σκύρτος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο ερωτήσεις. Η Τραπεζική Ένωση προχωρά σύμφωνα με το σχέδιο και η Κομισιόν συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση με πολύ θετικό τρόπο. Πολλοί όμως επαγγελματίε στο τραπεζικό τομέα πιστεύουν ότι οι νέοι κανονισμοί ε, ε, ε, τελικά θα υποχρεώσουν τις μεγάλες τράπεζες της Ευρώπης να μειώσουν το μεγέθη τους και θα καταστήσουν έτσι πιο δύσκολο τον ανταγωνισμό με τις αμερικανικές τράπεζες σε παγκόσμιο επίπεδο. Πώς απαντάτε σε τέτοιου είδους ε, επικρίσεις. Ε, υπάρχει κίνδυνος υπερβολικά πολλών ε, κανονισμών και περιορισμών που θα έχουν αντίστροφε επιπτώσεις στην απόδοση των μεγάλων ευρωπαϊκών τραπεζών και μια ερώτηση που αφορά την ελληνική κατάσταση. Τέσσερις ε, ε, ελληνικές συστημικές τράπεζες θα ολοκληρώσουν την τρίτη τους ανακεφαλαιοποίηση σε πολύ αντίξιες οικονομικές συνθήκες. Πιστεύετε πως ο ελληνικός τραπεζικός τομέας θα μπορέσει να ακολουθήσει την τάση προς την Τραπεζική Ένωση σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που εσείς έχετε παρουσιάσει ή πιστεύετε ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι ειδική περίπτωση ε, που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αντιμετωπιστεί με βάση εξαιρέσεις στους κανόνες. Ευχαριστώ. On um, first point. Ε, Για το πρώτο. Νομίζω πως το ερώτημα είναι κατ' ουσίαν αν υπάρχουν ε, υπερβολικοί κανονισμοί. Εν μέρη αυτό είναι ε, αυτό το οποίο μας ε, απασχολεί όλους. Νομίζω πως υπάρχει η αίσθηση παντού στο Συμβούλιο Συστημικής Σταθερότητας ε, ότι κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουμε να δούμε το, αν τα έχουμε κάνει σωστά τα πράγματα ειδικά όσον αφορά την ανάπτυξη και τις δουλειές. Αυτή είναι η απάντησή μου το γενικό ερώτημά σας όσον αφορά τώρα τα περαιτέρω πιθανά αριθμιστικά μέτρα που θα έρθουν ξέρουμε πως υπάρχει η Τίλα το Έμρε που έρχεται και άλλες συζητήσεις που γίνονται σε άλλα φόρα στη Βασιλεία η προσέγγιση που πρέπει να ακολουθήσουμε είναι να προσπαθήσουμε να λειτουργήσουμε εντός ενός ε, διεθνούς ε, ρυθμιστικού πλαισίου. Αυτό κάνουμε με το ΤΗΛΕΚ. Αλλά ταυτόχρονα όταν λέμε πως ναι, αυτές οι συστάσεις ε, προέρχονται από διάφορες επιτροπές, πρέπει να αναρωτηθούμε εάν αυτά είναι πάντα σωστά για το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα το οποίο έχει μια διαφορετική ιστορία και διαμόρφωση από το αμερικανικό σύστημα και δεν θεωρώ ότι πρέπει απλά να εισάγουμε όλα τα χαρακτηριστικά που μπορεί να ταιριάζουν στο αμερικανικό μοντέλο και να τα εφαρμόζουμε έτσι απλά στο ευρωπαϊκό. Χρειαζόμαστε λοιπόν ε, ισχυρό τραπεζικό τομέα, τράπεζες οι οποίες θα συνεχίσουν να επιτελούν τον ρόλο τους όσον αφορά τη δημιουργία αγοράς, θα μπορούν να δανείζουν και να ανταγωνίζονται. Όσον αφορά τώρα τις ελληνικές τράπεζες και την νομοθεσία BRRD παραδείγματος χάρη, πρέπει να συνεχίσουμε με την νομοθεσία αυτή να την εφαρμόσουμε οριζόντια σε όλα τα κράτη-μέλη. Νομίζω πως είναι ενθαρρυντικά τα νέα όσον αφορά την θέση των ελληνικών τραπεζών, όσον αφορά την ανάγκη ανακεφαλαιοποίησης και την πρόοδο που σημείωσαν κάποιες όσον αφορά το κεφάλαιο που άντλησαν από ιδιώτες το οποίο οπωσδήποτε είναι ενθαρρυντικό, αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε πως οι μεταρρυθμίσεις αυτές ε, έγιναν για κάποιο λόγο και όλοι μας ε, πρέπει να συνεχίσουμε αυτή τη ε, μεταρρυθμιστική διαδικασία. Ευχαριστώ. Πέτερ Τσιμέρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στην διάσκεψη τύπου την προηγούμενη Τρίτη είπατε Λόρδε Χίλ πως ένα εθνικό σύστημα εγγύησης καταθέσεων θα μπορεί να προσφύγει στο ευρωπαϊκό αν το κράτος μέλος δεν έχει εφαρμοσει μόνο την παλαιά οδηγία αλλά και τον κανονισμό SRM και την οδηγία BRRD αν την έχει μεταφέρει πλήρως στο εθνικό δικαίωμα. Το ερώτημά μου ισχύει αυτό. Αν δει κανείς το άρθρο 41.1 μιλάει πως προϋπόθεση είναι η μεταφορά των άρθρων 4, 6, 9 και 10. Για SRM και BRD δεν βλέπω τίποτα ως προϋπόθεση. Οπότε το ερώτημά μου είναι η πλήρης εφαρμογή της BRD και του SRM είναι προϋπόθεση για να υπάρχει πρόσβαση στο ταμείο το οποίο θέλετε πρώτα απ' όλα για μια αντασφάλιση και μετά για μια κοινή εγγύηση των καταθέσεων. Το δεύτερο μου ερώτημα αφορά τα ταμεία που ήδη υπάρχουν. Δεν βλέπουμε ακριβώς πώς θα μεταφερθούν τα εθνικά αυτά ταμεία ε, σε ένα κοινό Γιατί είναι σημαντικό αυτό, γιατί μιλήσατε ε, ρητός παραδείγματος χάρη για τα ταμιευτήρια και τις συνεταιριστικές τράπεζες και το ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη η μορφή του κινδύνου τους. Σημαντικό είναι λοιπόν τα συστήματα αυτά να μπορούν να λειτουργήσουν και να έχουν ένα ταμείο στη διάθεσή τους όπως είχαν μέχρι τώρα γιατί χωρίς ένα τέτοιο ταμείο βεβαίως δεν μπορούν να επιτελέσουν το ρόλο τους πώς διασφαλίζεται ότι κατά τη μεταφορά των εθνικών ταμείων που δημιούργησαν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε εθνικό επίπεδο θα συνεχίσει να υπάρχει η ίδια διασφάλιση και ότι θα υπάρχουν επαρκή κονδύλια για να καλύπτονται πλήρως οι λειτουργίες τους. Well, I think on the... Λοιπόν, για το πρώτο θέμα το οποίο θίξατε. Υπάρχει μια απλή πρακτική απάντηση όσον αφορά την εφαρμογή της BRRD γιατί σύμφωνα με τις τελευταίες δικές μου πληροφορίες ε, το BRD θα μεταφερθεί πλήρως ε, μέχρι το τέλος του έτους σε 27 τη μελη και το τελευταίο μέχρι τον Ιανουάριο. Οπότε, μέχρι να καταλήξουμε σε αυτήν την πρόταση θα έχει εφαρμοστεί πλήρως. Για το δεύτερο αυτό σημείο, οπωσδήποτε ισχύει το ότι θέλουμε να σχεδιάσουμε ένα σύστημα το, στο οποίο οι εισφορές θα βασίζονται στον κίνδυνο κατά τρόπον ώστε οι τράπεζες οι οποίες θα είναι πιο ασφαλείς να συνεισφέρουν λιγότερο. Στο... Και με βάση αυτό ακριβώς ε, προχωράμε την πρότασή μας. Προφανώς ε, εξετάζουμε το ποιο θα είναι αυτό το σύστημα, θα είναι μέρος της νομοθετικής ε, διαδικασίας. Νομίζω πως ε, θα είναι το Συμβούλιο Συστημικής Σταθερότητας μάλλον, αυτό το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή. Οπότε νομίζω πως έτσι θα έχουμε ένα σύστημα εύρωστο για να χρηματοδοτήσουμε το σύστημα εγγύησης καταθέσεων. Ε, Βεβαίω ε, σωστά αυτά τα οποία λέτε, τα αντιλαμβάνομαι και πραγματικά σας είμαι ευγνώμων για αυτές τις συζητήσεις. Αντιλαμβάνομαι πως ε, και τους επόμενους μήνες θα πρέπει να απαντήσουμε αυτές τις ε, ερωτήσεις ακριβώς για να ικανοποιήσουμε εσάς και τους άλλους για ε, να σας πείσουμε ότι το έχουμε σκεφτεί σωστά. Μία σύντομη ερώτηση. Ακριβώς, αυτή, η, ακριβώς για αυτή τη δουλειά των επόμενων μηνών. Μιλήσατε για το πώς θα γίνει η επιμέτρηση του κινδύνου που θα πάει στο επίπεδο 2. Όμως το να πηγαίνει στο level 2 ε, είναι τελείως διαφορετική εκτίμηση εντός της ε, Κομισιόν από ότι εκτίμηση που κάνει το Κοινοβούλιο από δεξιά μέχρι αριστερά. Πώς ε, θεωρείτε ότι υπάρχει κάποιος τρόπος να συζητήσουμε ακριβώ αυτό το επίπεδο κινδύνου μεταξύ ημών και του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Κοιτάξτε, νομίζω πως ο ακριβής ε, τρόπος με τον οποίο θα αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα ακόμα δεν έχει καθοριστεί, αλλά οπωσδήποτε έχουν την εντύπωση πως ε, δεν θα σημειωθεί πρόοδος ε, εκτός εάν συμφωνήσουμε να γίνει. Και οπωσδήποτε είμαι στη διάθεσή σας και σας και των συναδέλφων για τη συζήτηση Ευχαριστώ, Brian Case. Σας ευχαριστώ, Επίτροπε. Καταρχήν είμαι ευτυχής που το διευκρινίσατε και νωρίτερα πως οι ιστορικές καταρρεύσεις τραπεζών δεν περιορίζονται μόνο στην Νότια Ευρώπη. Χαρακτηριστικό και θεαματικό παράδειγμα είναι η δική μου χώρα τελευταία δεκαετία περίπου και είναι σημαντικό να το αναγνωρίσουμε αυτό. Δύο ερωτήσεις για τον Επίτροπο Χιλ. Καταρχήν για το TTIP Είδαμε την κατάρρευση του Lehman Brothers το 2008 και πόσο συνδέονται οι χρηματοπιστωτικές αγορές στην Αμερική και στην Ένωση. Ξέρουμε το επίπεδο των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών ανάμεσα στα δυο μας συστήματα και το γεγονός ότι έχουμε δύο διαφορετικά σύνολα κανόνων για τις ίδιες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Εσείς πιστεύετε πως υπάρχει δυνατότητα για ένα χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο για το τίτλο εφόσον γίνεται τώρα αυτός ο επόμενος γύρος συζητήσεων και διαπραγματεύσεων και κατά τη γνώμη σας θα ήταν, δεν θα ήταν συστημική αποτυχία εάν δεν συμφωνήσουμε για την αναγκαιότητα ενός χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου ως κομμάτι ενός γύρου TTIP. Και δεύτερη μου ερώτηση για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Μπορείτε να μας πείτε πότε θα κάνετε ένα πράσινο βιβλίο για αυτό το θέμα. Στο παρελθόν ξέρω ότι το έχετε αναφέρει. Πάντως είναι γεγονός ότι λιγότερο από το 3% των Ευρωπαίων καταναλωτών ε, χρησιμοποιούν ε, ε, πιστοτικές κάρτες νηπόθηκων δανείων, ασφαλιστικά πλάνα για, σε άλλες χώρες δεδομένου ότι υπάρχουν τόσο διαφορετικές τιμές στα ενυπόθηκα δανείο, στα ανυπόθηκα δάνεια, σε, μένα, σε εμάς πούμε στη χώρα μας είμαστε στο 4% ε, επιτόκιο, ενώ σε άλλες χώρες έχει φτάσει στο 2%. Τι σκοπεύετε να κάνετε λοιπόν για να μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε χρήματα σε βασικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και για τις δύο ερωτήσεις, λέει ο Επίτροπο. Για τη δεύτερη, τις ελληνικέ χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Εγώ ε, σκοπεύω να δημοσιεύσω ένα πράσινο βιβλίο την επόμενη εβδομα... Ε, τον επόμενο μήνα, συγγνώμη, το Δεκέμβριο. Στις αρχές δηλαδή, σε μια-δύο εβδομάδες. Και Τώρα, αυτό στόχο θα έχει, όπως κάναμε και με την Ένωση Κεφαλαιοχωρών και το σχετικό πράσινο βιβλίο, είναι να ξεκινήσουμε μια συζήτηση που έχω προσπαθήσει, θέλω να και βέβαια ακόμα πρέπει να περάσει από το Συμβούλιο των Επιτρόπων. Πάντως θέλω να ξεκινήσουμε τη συζήτηση ακριβώς όπως είπατε και εσείς από, ε, από την οπτική του καταναλωτή. Δηλαδή αντί να ακολουθήσουμε μια πιο παραδοσιακή προσέγγιση θεσμικού τύπου, να σκεφτούμε τις σηματοπιστωτικές υπηρεσίες από την άποψη των συμπολιτών μας που τις χρησιμοποιούν. Είτε πρόκειται για αυτοκινητική ασφάλιση, είτε πρόκειται για ενυπόθηκο δάνειο, είτε είναι για ασφάλεια ζωής. Ιδιαίτερα στην ενοικίαση αυτοκινήτων όπου νομίζω πολλά μπορούν να γίνουν για να βελτιωθεί η διαφάνεια σε, αυτή, σε αυτό το τομέα. Όλοι είχαμε εμπειρίες με την ενοικίαση αυτοκινήτων στις διακοπές μας. Αλλά να έχουμε και μια πρακτική προσέγγιση και να βρούμε τρόπους για να γίνουν βελτιώσεις. Λόγο για αυτές τις διαφορές στον οποίο οφείλονται αυτέ τι διαφορέ είναι διαφορετική ιστορικά η φύση των αγορών, νομοθεσία κτλ. Πάντω δεν είναι και τόσο απλό. Αλλά νομίζω πω όλα τα θέματα που αναφέρετε θα έπρεπε να βρίσκονται εδώ και αυτό θέλω και να εξετάσουν και τα, να εξετάσει το πράσινο βιβλίο και να βρούμε προτάσει για να προχωρήσουμε. Για το TTIP. Συμφωνώ εντόνως μαζί σας για το πρέπει να έχουμε ένα σύστημα καλύτερο για να ορίσουμε τους χρηματοπιστωτικούς κανονικούς, γιατί ελέγχεται η πρόσβαση στην αγορά για να... Και αν δεν λειτουργούν σωστά και με τον ίδιο τρόπο οι αγορές, η αμερικανική με την ευρωπαϊκή, δεν είναι και πολύ έξυπνο. Είναι δύο διαφορετικά συστήματα που παράλληλα λειτουργούν. Εγώ πιστεύω πως είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να το ζητάμε αυτό στο TTIP. Τώρα, τι θα καταλήξουμε δεν ξέρω ακριβώς, διότι, όπως γνωρίζετε, υπάρχουν και ένα ολόκληρο σύνολο στο οποίο στοχεύουμε. Πάντως, το προχωράμε και επιμένουμε ακριβώς για τους λόγους που αναφέρατε να βρούμε ένα δηλαδή τρόπο για να έχουμε καλύτερη συνεργασία για τον δημοσιονομικό κανονισμό και γι' αυτό και πρέπει να συνεχίσουμε τις ε, συνομιλίες. Ο Γιάκο Φαμβαϊστέκερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε έχω δύο ερωτήσει Η πρώτη βέβαια αφορά τις ε, διαφορετικές μεταρρυθμίσεις στις τράπεζες ε, Χαιρετίζω το ενδιαφέρον που δείχνετε για αυτό το φάκελο, το εκφράσετε και απόψε. Και σε μια πρόσφατη ανακοίνωση ε, ε, ε, δεν αναφέρεται καν εκεί το, το θέμα αυτό των διαθετικών ταπεισικών μεταρρυθμίσεων. Μήπως θα πρέπει να τη διαβάσουμε και να την θεωρήσουμε εκχώρηση αρμοδιοτήτων Ο προκάτοχός σας αυτό θεωρούσε ότι είναι ο τέταρτος πυλώνας ε, της ε, Τραπεζικής Ένωσης και έχει γίνει ρεζέρβα. Ε, δηλαδή έχει υποβαθμιστεί η σημασία. Τελικά αυτός ο τέταρτος πυλώνας τι έχει γίνει. έχει γίνει η ρεζέρβα στις τέσσερις τροχούς, άρα κάτι άχρηστο. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την ε, το έντισε εγγύηση των καταθέσεων. Οι οικονομολόγοι αντιλαμβάνονται το ζήτημα της ασφάλειας αυτής ε, ως ένα θέμα που λειτουργεί καλά όταν υπάρχει άγνοια. Δεν ξέρουμε τι θα γίνεται μετά από 15-20 χρόνια. Αν δούμε ε, το 2024, το 2024 που το σύστημα θα είναι πλήρως σε λειτουργία στα δικά σας σχέδια, μπορεί το πέπλο αυτό της άγνοιας ε, να μην είναι εντελώς ε, ε, διαφανές. Εσείς μας λέτε στις προτάσεις σας ε, κάποιες ημερομηνίε. Αυτό είναι πιο σημαντικό ή η ολοκλήρωση των προαπαιτούμενων. Που φαίνεται και αυτό να σας ενδιαφέρει. Αυτό είναι το δεύτερο ερώτημά μου. Για το δεύτερο ερώτημα. για την ημερομηνία. Θέλαμε να ευθυγραμμίσουμε το χρονοδιάγραμμα αυτό με την ημερομηνία έναρξη ισχύω ε, του Ταμείου για την εξηγία στον Τραπεζών. Αλλά επειδή υπάρχει ένα άλλο ανθάνων ερώτημα στην ερώτηση που μου κάνατε και έχω υποδιαιρέσει ε, το χρονοδιάγραμμα σε διάφορες φάσεις. Γιατί το έκανα αυτό, γιατί νομίζω και ελπίζω ότι θα μπορέσω να κάνω βαθμιδόν πρόοδο, γιατί μόνο με αυτή τη σταδιακή πρόοδο πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να φτάσουμε και που πιστεύω και ελπίζω ότι μπορούμε να φτάσουμε μέχρι το 2024. Άρα η ημερομηνία δεν νομίζω ότι είναι μια διαδική επιλογή. Αλλά θα μας βοηθήσει αυτή η προσέγγιση να πετύχουμε αυτό το χρονοδιάγραμμα που είναι λογικό χρονοδιάγραμμα. Νομίζω γιατί επαναλαμβάνω ευθυγραμμίστε και με άλλα αντίστοιχα χρονοδιάγραμματα. Σε αυτό το πρώτο σας ερώτημα και το PSR. Νομίζω ότι ουσιαστικά αυτό που είπατε στην αρχή έχει νόημα. Δηλαδή, η πρόοδος στις τραπεζικές διαδοτικές μεταρρυθμίσεις είναι κάτι το οποίο ήδη έχει καθυστερήσει, έχει πάρει πολύ περισσότερο χρόνο από όσα θα θέλαμε όλοι και εσείς και εγώ. Και εγώ πάντοτε έλεγα ότι η δική μου προσέγγιση κατά βάση είναι καλύτερα λιγότερη νομοθεσία όταν όμως κάποιος νομοθετεί να εφαρμόζεται αυτό που νομοθετεί ταχύτερα. Γιατί πολλές φορές κάθονται οι φάκελοι για χρόνο, πολύ. Και αυτό δεν είναι καλό και για την πολιτική συζήτηση. Και άπαξε έχει λοιπόν θεσμοθετηθεί μια νομοθεσία, θα πρέπει να εφαρμόζεται σωστά. Αυτή είναι η απόψη μου γενικά για την νομοθεσία. Τα μέτρα λοιπόν αυτά που αναφέρονται στην ανακοίνωση ήταν νέα μέτρα, ήταν βήματα που δεν έχουν γίνει ακόμη δεν έχουμε ξεκινήσει τη σχετική νομοθεσία, τη κτλ. Και το PSR, σας είπα, ε, το εξήγησα, το πώς μπορούμε να επιτύχουμε πρόοδο και πιστεύω ότι αυτό θα κάνει και πιο ισχυρό το τραπεζικό μας σύστημα. Ναι, αλλά δεν μας είπατε ποιος είναι ο ρόλος. Το PSR. Δυστυχώ κόβεται το μικρόφωνο του μιλητή. Ναι, μάλιστα. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο, τον Τζόναθαν Χιλ και όλου του συναδέλφου, γιατί πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ανταλλαγή απόψεων. Και τώρα περάσουμε στην νομοθετική διαδικασία αυτή καθεαυτή. Έχουμε και νέα ζητήματα, νέου φακέλου. Ήδη έχουμε αναθέσει την εξέταση των φακέλων θα σας πω ποιοι είναι οι συγητές. Αυτής αμέσως. Θα ξεκινήσει λοιπόν η νομοθετική διαδικασία και ίσως κάποιες παρεμβάσεις και κάποια ζητήματα που έθισαν οι συνάδελφοι να επιληθούν δια της κανονικής νομοθετικής διαδικασίας. Σας ευχαριστούμε πολύ, Τζόναθαν. <laughs> Αγαπητοί συνάδελφοι, περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Έχω να κάνω μια ανακοίνωση. Πρώτα απ' όλα, για την αυριανή κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Απασχόλησης θα ξαναφτιαχτεί η αίθουσα στο μεσημεριανό διάλειμμα από πάρτε τα χαρτιά μαζί σας. Λοιπόν, ενημέρωση για τους διαλόγους. Στις 20 Νοεμβρίου είχαμε τον τελευταίο και έβδομο γύρο διαλόγου και καταλήξαμε σε μια συμφωνία στις 25 του μηνός, νωρίς το πρωί και συμπεριλήφθησαν τα εξή σημεία. Ένα καθεστώς αναλογικότητας όπου η συγκριτική αξιολόγηση μπορεί να θεωρηθεί κρίσιμη, σημαντική και μη σημαντική. Κατόπιν υπάρχουν πολλές κατηγορίες συγκριτικής αξιολόγησης, ε, μεταξύ των οποίων το επιτόκιο και κάποια αξιολόγηση τρίτων χωρών, ένα καθιστός de minimis ε, και βεβαίως όσον αφορά την ισοδυναμία τρίτων χωρών αυτό μπορεί να γίνει είτε μέσω αναγνώρισης είτε μέσω ισοδυναμίας ε, και η ΕΣΜΑ και οι άλλες ρυθμιστικές αρχές ε, θα εξοδοτηθούν για την έγκριση. Οι τεχνικές εργασίες συνεχίζονται και αναμένουμε η ψηφοφορία του τελικού κειμένου να γίνει μόλις φτάσει επιστολή από την Κορεπέρ. Η Κορεπέρ έχει προγραμματιστεί για την 9η Δεκεμβρίου, οπότε συγχαίρω τον κύριο Νιουενχόιζεν και τη διαπραγματευτική ομάδα. Κατόπιν άλλος ένας διάλογος ε, για τα στατιστικά στοιχεία ισοζυγίου, εμπορικού ισοζυγίου και αυτό στις 23 Νοεμβρίου συζητήσαμε τα βασικά ζητήματα και θα έχουμε το δεύτερο γύρο στα μέσα Δεκεμβρίου. Τέλος, δύο γύρι διαλόγου για ένα αρμονισμένο δίκτυ τιμών καταναλωτή Κατά βάση φτάσαμε σε μια πολιτική συμφωνία. Υπάρχει ένα στοιχείο ακόμα που πρέπει ε, να ξεκαθαρίσει μεταξύ Κομισιών και Συμβουλίου όσον αφορά το Κοινοβούλιο. Εμεί ε, θεωρούμε ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και πραγματικά ενθαρρύνω Συμβούλιο και Κομισιό να καταλήξουν σε μια συμφωνία. Για ένα σημείο σημαντικό αλλά όχι τόσο κρίσιμο τελικά. Τώρα, να αναφέρω τι συστάσεις και αποφάσεις της τελευταίας συνεδρίασης των συντονιστών. Τώρα, λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την νέα διαδικασία την οποία θα αναλάβει ο Ρίτσαρτ Σούλικ από το ECR σύμφωνα με το άρθρο 46 εδαφείο 2 του κανονισμού. Πρόκειται για μια διαδικασία νομοθετική και αφορά ένα σύστημα καθορισμού κοινή αξίας για τη φορολογητή αήλη και σύμφωνα με αυτή τη διαδικασία αν το δεχτεί αυτό η Επιτροπή, ο κάθε βουλευτής μπορεί να συλλέγει υπογραφές και αν μαζέψει την ε, πλειοψηφία, την... τις υπογραφές της πλειοψηφίας των μελών ε, του Κοινοβουλίου θα πρέπει η διάσκεψη των Προέδρων να δώσει άδεια για μια έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας κάτι το οποίο οπωσδήποτε θεωρούμε πως είναι θετικό και χρήσιμο τα κράτη-μέλη να ξεκινούν τα... οι βουλευτές με να ξεκινούν από μόνο τους ε, την διαδικασία έκθεσης ίδιας ε, πρωτοβουλίας. Ένα ενδιαφέρον πείραμα, ελπίζω να αποδειχθεί επιτυχές. Τέλος επιπρόσθετες κεφαλαιακές απαιτήσεις ε, για εταιρείε ε, ασφαλιστικές που αριστεριοποιούνται σε όλους τους κλάδους ασφαλιών για εννέα τέτοιες ε, εταιρείε. Οι πληροφορίες αυτές θα σας διαβαστούν εν το χρόνο. Τέλος έχουμε ανάθεση φακέλων. Κοινοί κανόνες για κεφαλαιοποίηση, σοσιαλδημοκράτε, ε, προληπτικέ ε, απαιτήσει ε, για την τηλεοποίηση το ΕΛΚ, αναθεώρηση τη οδηγία για τα προσπέκτου στην ΑΛΔΕ, Ευρωπαϊκό Σύστημα Αντασφάλισης Καταθέσεων ΕΛΚ, προπολογισμό για την Ευρωζώνη σοσιαλδημοκράτες και συμφωνήσαμε πως η μελλοντική νομοθετική πρόταση για την ε, λύση τραπεζών θα πάει στην ομάδα του ECR. Τέλος, σύμφωνα με τη σύσταση της 26 Νοεμβρίου, το Κοινοβούλιο θα δώσει την δική του άποψη με ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στην ε, έκθεση για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο που θα υιοθετηθεί το Φεβρουάριο του 2016 προθεσμία για τροπολογής έχει πάει 8 Ιανουαρίου του 2016 και 18 Φεβρουαρίου ψηφοφορία στην Επιτροπή αυτά με τις ανακοινώσεις και τώρα περνάμε στο σημείο 5 της ημερησίας διάταξης και έχω τον λόγο ως το θέμα είναι Τραπεζική Ένωση Ετήσια Έκθεση 2015. Και θα μιλήσω και Ιταλικά και θα αλλάξει και η δουλειά μου. Ε, Ευχαριστώ συνάδελφοι. Πρόκειται για την πρώτη έκθεση, για την έκθεση περί της Τραπεζικής Ένωσης με την οποία η Επιτροπή μας στόχο έχει να αναλάβει και ε, το λεπτό έργο της συμπλήρωσης ε, του έργου του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου όσον αφορά την πρόοδο της Τραπεζικής Ένωσης καθώς και των συνιστοσών του. Άρα λοιπόν αποδίδω όχι μόνο επειδή είμαι εισηγητής αλλά λόγω της μεγάλης σημασίας της λειτουργίας του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου που δίδω σημασία σε αυτό την έκθεση που θα είναι η πρώτη μια σειρά ετησίων εκθέσεων ε, μέσω των οποίων ακριβώς θα κληθούμε να μιλήσουμε όχι μόνο για την Τραπεζική Ένωση αλλά και ε, κυρίως θα ήθελα και να πω για την συγκεκριμένη αξιολόγηση των διαφορών πυλώνων ε, για να δούμε ακριβώς και πώς ε, λειτουργούν όλα αυτά. Έχουμε μία έκθεση λοιπόν σε τρία μέρη. Δεν χρειάζεται να σα αναφέρω τι αξιολογήσει όσον αφορά τη σημασία τη λειτουργία τη Τραπεζική Ένωση, πράγμα το οποίο είναι γνωστό. Και τα τρία τμήματα τη έκθεση είναι βέβαια η ενιαία εποπτεία, η ενιαία εξυγίαση και το τρίτο συστατικό, ο πυλώνα τη σύσταση. Βεβαίω, ε, έχουμε μία ιδιαίτερη προσοχή στον πρώτο πυλώνα καθώς την επαύριο του εορτασμού της, ε, του επαιτίου της ενιαίας εποπτείας, Ξέρουμε πως δεν είναι καθόλου εύκολο, αλλά είναι απαραίτητο να μπούμε στις λεπτομέρειες και να δούμε τι λειτουργήσε, τι μπορεί περαιτέρω να βελτιωθεί σε αυτή την πρώτη χρονιά ενιαίας εποπτείας. Η εξολόγηση που εγώ ε, διατυπώνω στην έκθεση είναι συνθετική είναι σύντομη ε, και λέει ότι ε, θα πρέπει να θεωρηθεί επιτυχής ε, αυτή η προσπάθεια και λόγω της ποιότητας της εποχής, αν και φυσικά είναι λογικό και απαναπόφευκτο να υπάρχουν και κάποια στοιχεία πιο δύσκολα τα οποία προσπαθούμε να εντοπίσουμε και περιθώριο βελτίωσης βέβαια. Πρώτη πτυχή και αναλύω την λειτουργική ανάλυση, όπου δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι πολύ θετική αξιολόγηση, ίσως να μην είναι έχει ληφθεί ε, παρκώς υπόψη η ανάγκη αυτής της πρόκλησης της οικοδόμησης μιας ενιαίας εποπτείας. Εδώ λοιπόν αναλύουμε και κάποιες ειδικέ πτυχές προς τις οποίες είναι πολύ θετική η κρίση, δηλαδή η διαδικασία ομοδοποίησης, ε, η κατασκευή του εγχειριδίου εποπτείας, ε, η πληροφορική δημιουργία ε, ομάδων κοινής εποπτείας, η διαδικασία υλοποίησης και εφαρμογής των κοινών διαδικασιών και ένα στοιχείο που προέκυψε από την ε, δράση εποπτείας φέτος είναι ότι ακριβώς υπάρχουν διάφορες διοικητικές διαδικασίες και άρα η αξιολόγηση που λέει ότι εμείς είμαστε έτοιμοι να αξιολογήσουμε προτάσεις και μάλλον και να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα, να μειώσουμε δηλαδή το φόρτο στις υποδομές σε όλα τα επίπεδα μέσω μηχανισμών Ανάθεση ορισμένων διοικητικών λειτουργιών. Φυσικά θα πρέπει να διευκρινιστεί περισσότερο επί τη βάση των προσανατολισμών. Όσον αφορά τι μεικτέ ομάδε εποπτεία, και εδώ είναι πολύ θετική η κρίση μα, αν και φυσικά και εδώ θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο την ποιότητα της συμμετοχή των εθνικών αρμόδιων αρχών. Κάτι πιο κρίσιμο το οποίο προέκυψε είναι ε, ο ανεπαρκής προγραμματισμός της δράσης της εποπτείας επί του οποίου φαίνεται να υπάρχουν κάποια μικροπροβληματάκια και περιθώρια βελτίωσης. Φυσικά υπογραμμίζουμε την ανάγκη να μιλήσουμε για την λογοδοσία, την αποφυγή της διπλής κάλυψης, για την αποφυγή επιπλέον διοικητικού κόστους και αχρίας του περιττού διοικητικού κόστους. Άρα λοιπόν ίσως αν είναι σκόπιμο να ενισχυθεί η συνεργασία ανάμεσα στις τρεις γενικές διευθύνσεις ε, εποπτεία, ε, μακρο τη μακροπροληπτική ε, εποπτεία αλλά και ε, μια γενική κοινή προσέγγιση εποπτείας. Όσον αφορά τώρα τις πολιτικές εποπτείες, είναι μια αξιολόγηση πολύ θετική όσον αφορά την γενική αξιολόγηση, όπως είπα, μπορούμε να επαναλάβουμε ότι η γενική όθηση όσον αφορά την ποσότητα και την ποιότητα του τραπεζικού κεφαλαίου δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως ε, αντίφαση με τη δράση στήριξης της οικονομίας. Οι τράπεζα θα πρέπει να είναι καλά κεφαλοποιημένες ώστε να λειτουργούν σωστά και φυσικά θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και την συγκυρία. Οπότε, ένα στοιχείο πιο αποτελεσματικού συντονισμού ανάμεσα στις προληπτικές και μακροπροληπτικές πολιτικές υπογραμμίζεται ως ανάγκη για να υπάρξει μια γενικότερη σταθεροποίηση των περιουσιακών στοιχείων ώστε να εισαχθούν και στοιχεία ε, σταθερότητας. Όσον αφορά το ΣΕΡΕΠ έχουμε νέα ευρωπαϊκή μεθοδολογία αν και πιθανότατα αυτή η μεθοδολογία θα μπορούσε αργότερα να αλλάξει γιατί οριστικοποιήθηκε στην πορεία. Έχουμε δε και το κατόφλι για την κατανομή των πληρωμών γιατί πιστεύω πως η προσέγγιση η οποία επελέγει δεν είναι η μοναδική και ίσως ένα περαιτέρω στοιχείο, μια μεγαλύτερη ευηλιξία που μπορεί να έχει προκύψει ανάμεσα στο δεύτερο πυλώνα και το κατόφλι του NBA, θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη. Τώρα, για την εποπτεία. Δεν μπορέσαμε να αναλύσουμε στη διατύπωση της ε, έκθεσης τη πρόταση και τις επιλογές όσον αφορά την εθνική διακριτική ευχέρεια θα είναι αυτό αντικείμενο εις βάθος ανάλυσης. Εν γέννη πάντως νομίζω είναι θετική η στάση, ίσως θα πρέπει κάπως να εμβαθύνουμε σε κάποιες πτυχές όπως ας πούμε για τη Δανέζικη συμβιβαστική αν η επιλογή που έγινε για τις δύο διαφορετικές νομικές βάσεις δηλαδή εξασφαλίζει ένα ισότιμο πεδίο, level playing field όπως λέμε. Υπογραμμίζεται επίση η προσπάθεια που έχει γίνει όσον αφορά τις σταθμισμένε δραστηριότητε ε, για την εκτίμηση του κινδύνου και εδώ ίσως όμως να μην είναι δυνατόν να μετρήσουμε με όλες τις μορφέ τραπεζικού κινδύνου πέρα από τον πιστοτικό κίνδυνο και αυτό εδώ προέκυψε από την συνολική αξιολόγηση ιδιαίτερα για τι δραστηριότητε επίπεδου ρία. Για λόγους χρόνου τώρα θα πρέπει να αφήσω κατά μέρος τις άλλες πτυχές. Πρέπει να υπογραμμίσω ότι η αξιολόγηση είναι θετική και βεβαίως θα περιμένω και τις δικές σας παρατηρήσεις. Στο δεύτερο κεφάλαιο είναι η, μια ενιαία λύση για να δούμε ακριβώ την εργασία που έχει γίνει ε, και τελευταίο το κομμάτι είναι αυτό το οποίο είναι αφιερωμένο στο δεύτερο πυλώνα και το, το, το, το συζητήσαμε με τον Λόρδο Χίλ, δηλαδή bridge financing και backstop όπου βέβαια υποστηρίζουμε τη σημασία της πλήρους αποδοχής και μεταγραφής της οδηγίας BRRD για την ανάκαμψη και την εξυγίαση και εκείνο στο οποίο εργαζόμαστε, το Bridge Financing, για το κατά πόσο δηλαδή αυτό είναι κάτι σκόπιμο Γι' αυτό και η έκφραση, η έκφραση μάλλον της δυνατότητας λειτουργίας ε, χρήσης του ESM ε ε, για αυτό το σκοπό. Σημαντικές παρατηρήσεις που εγώ προσωπικά συμφωνώ με αυτές. Τέλος έχουμε το backstop, έχουμε το bridge financing, αλλά έχουμε και το backstop για ενδεχόμενες περαιτέρω απαιτήσει πέρα από το maximum κατόφλι. Τρίτο πυλώνα, δεν έχω να πω πολλά. Τώρα πήραμε την νομοθετική πρόταση. Ήδη, όπως είχαμε φανταστεί, έχει προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά από αυτού η έκθεση δεν λέει πολλά. Θα μείνει στο ελεύθερο κοινοβουλευτικό παιχνίδι την κανονική τακτική νομοθετική διαδικασία για να μπορέσει το Κοινοβούλιο να συμφωνήσει σε αυτό το τομέα. Μια τελευταία έκκληση για τους συναδέλφους. Είναι δύσκολη αυτή η έκθεση και ελπίζω πως θα οριστούν έτσι κάποια φόρμα για την Τραπεζική Ένωση και θα ήθελα να εστιάσω την προσοχή στην αξιολόγηση της συγκεκριμένης δράσης για την ενιαία εποπτεία κτλ. Παρά να κάνω μια έκθεση για όλη την Τραπεζική έπτωση, διαστατική σε συγκεκριμένε νομοθετικέ δηλαδή διαδικασίε. Για αυτά όλα έχουμε άλλα μέσα. Συχνά Αυτά διέπουν την τακτική νομοθετική διαδικασία. Γι' αυτό και θα ήθελα να διατηρήσουμε τη φύση αυτή τη έκθεση, αν συμφωνείτε κι εσεί, έτσι ώστε να συμβάλλει στη διαδικασία ε, ε, του SSM και του SRM. Um, Πρώτος ομιλητής εκ μέρους του ΕΛΚ, Burkhard Balz. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την έκθεση που παρουσιάσατε αγαπητέ Ρομπέρτο. Να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Θεωρώ πως Πρέπει να δούμε συνολικά το θέμα των σχέσεων τραπεζών και κρατών. Δεν είναι δυνατόν και ο εθνικός ε, φορολογούμενος να αντικατασταθεί απλά από τον ε, Ευρωπαίο. Θα πρέπει λοιπόν ε, συνολικά να μιλήσουμε για περαιτέρω μέτρα μείωσης του κινδύνου, κάτι το οποίο για μένα είναι σημείο κλειδί. Μετά, δεν θεωρώ πως ε, η αξιοπιστία της ε, Τραπεζικής Ένωσης ε, θα ενισχυθεί μέσω ενός κοινού backstop. Εγώ θεωρώ πως το bail-in μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά και εδώ πέρα θα βοηθήσουν δεσμευτικά και αρκετά υψηλά περιθώρια απολειών γύρω στο 8% θα έλεγα μετά, θεωρώ πως θα πρέπει να υπάρξει ένας επαρκής μηχανισμός χρηματοδότησης ε, γέφυρας ε, με τα απαραίτητα κίντρα. Άρα πρέπει ο τραπεζικός τομέας ε, να είναι τελικά υπεύθυνος για την πληρωμή και έτσι δεν θα χρειάζεται ένα κοινό backstop, ένα τέτοιο μηχανισμός. Και τελευταία σύντομη παρατήρηση, θεωρώ πως μια πιο αποτελεσματική προστασία των καταθέσεων δεν θα είναι μια κοινή προστασία των καταθέσεων, αλλά μια μείωση των κινδύνων που αναλαμβάνουν οι τράπεζες και επ' αυτού πρέπει να εργαστούμε τα επόμενα χρόνια. Αυτά και ευχαριστώ. Thank you. Σας ευχαριστώ. Πρέπει να πρέπει να έκανα ένα λάθος. Δεν είστε ο σκιώδης του ΕΛΚΑ. Σας έδωσα το λόγο, αλλά κανονικά πρέπει να τον είχα δώσει στην Εύα Παούνοβα. Λάθος μου. βαρός. σας έδωσα το λόγο. Τέλος πάντων, να το πούμε έτσι. Κυρία Πάουνοβα, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εσάς ως πρώτο και ως εισηγητή της έκθεσης η οποία αναφέρεται σε πολύ σημαντικά σημεία. Να αναφέρω και εγώ κάποια στοιχεία που θέλω να τονίσω. Θα ακολουθήσω την ίδια σειρά, αλλά θα είμαι πιο σύντομη. Σίγουρα πρέπει να αναπτυχθούν οι τρεις επιλώνες ε, της Τραπεζικής Ένωσης, SSM, SRM, δύο μηχανισμοί που θα πρέπει να ε, συμπληρώνονται και από το σύστημα εγγύης καταθέσεων. Αν θέλουμε τώρα ε, το SSM να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη που χάθηκε τα τελευταία χρόνια και να αποκαταστήσει την αντοχή του Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Συστήματος, θα πρέπει να ε, την χάνει τη σωστή διαχείρισης. και να δούμε τι θα γίνει και με τις δικαστικές, διαδικασίες. Και το Ταμείο πρέπει να εφαρμοστεί γρήγορα ε, και να βρεθεί ένας μηχανισμός ε, της ενδιάμεσης χρηματοδότησης που θα δίνει ε, στο Ταμείο επαρκή κονδύλια μέχρι ότου ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες. Ό,τι αφορά τώρα την εποπτική στρατηγική, θα πρέπει ε, η πολυμορφία των τραπεζικών μοντέλων να διατηρηθεί. Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα εγγύης καταθέσεων, λέτε ότι πρέπει να έχουμε ένα μηχανισμό εγγύησης που είναι σημαντικό αν θέλουμε να ενισχύσουμε τη χρηματοοικονομική σταθερότητα και να αποδυναμώσουμε τη σύνδεση τραπεζών ε, και εθνικής κυριαρχίας. Um, a little bit more to... Κάποια άλλα σημαντικά στοιχεία της έκθεσης. Μια προεξάρχουσα στρατηγική ευρωπαϊκό πλαίσιο υπηρεσιών. Πρέπει να εγκριθούν στο πλαίσιο αυτό σημαντικά ζητήματα που αφορούν τον κανονισμό για τα χρεόγραφα, καθώς επίσης και τις κεφαλακές απαιτήσει και το σχέδιο δράσης για την Ένωση Κεφαλαίου Αγορών. Πολύ σημαντικό είναι να καταλήξουμε σε μια ευρεία συμφωνία για τις πολυπληθείς αυτές μεταρρυθμίσεις για να υπάρχει λογοδοσία, έλεγχος και βέβαια διαφάνεια. Και βέβαια απαιτείται αποφασιστικότητα και πολιτική βούληση. Γιατί αυτό είναι καλό και για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Υπάρχουν πολλοί φάκελοι νομοθετικοί, δεν θα πρέπει όμως ε, ε, να μας διαφεύγει ότι είναι πολύ σημαντικό η υλοποίηση όλων αυτών των ε, μέσων και η παρακολούθηση της υλοποίησης. Βέβαια, πολλές φορές παραβλέπουμε κάποια σημαντικά αισθήματα όπως πώς μπορούμε τους πόρους μας εδώ στο Κοινοβούλιο να τους ε, αξιοποιήσουμε κατά το βέλτιστο δυνατό τρόπο ώστε να έχουμε πραγματικά παρακολούθηση αυτών των σημαντικών και πολυάριθμων νομοθετημάτων. Νομίζω ότι είναι σημαντικό για το προσωπικό μας και στο ευρύτερο θεσμικό επίπεδο, σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να έχει τη δυνατότητα να χειριστεί ως αυτούς τους φακέλους. Τούτων λεχθέντων θα συνεργαστώ μαζί σας και με τις υπηρεσίες σας επόμενες εβδομάδες για να ξεργαστούμε ακόμη περισσότερο την έκθεση. Σας ευχαριστώ πρώτα η Μπεατρίξ ε, Φον Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε τώρα την πρώτη ετήσια έκθεση για την ε, Τραπεζική Ένωση και σας ευχαριστώ που μας δώσατε την ευκαιρία να υποβάλουμε προτάσεις. Διαβάζοντας διαπιστώνω πως ε, οπωσδήποτε θα κάνουμε προτάσεις, δεν θα σας προξένει σε έκπληξη αυτό. Πρώτο κομμάτι, πρώτος πυλώνας, αναφέρατε ήδη πως ε, στην έκθεση αξιολογείται ε, πάρα πολύ θετικά την δυνατότητα εποπτείας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Δεν νομίζω να ισχύει κάτι τέτοιο. Πρόκειται για ένα έργο πραγματικά τιτάνιο και Ήδη βεβαίως ε, εσείς ε, αναφέρατε πως υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί, αλλά αμφιβάλλω αν ισχύουν και αυτά τα οποία λέτε. Κοιτάξτε, οι Γερμανοί ίσως να μην είναι γνωστοί για το χιούμορ τους ε, και τον καλό καιρό, αλλά οπωσδήποτε όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της διοίκησής μας, κάτι κάνουμε. Και στη Γερμανία χρειάστηκαν 10 χρόνια για να μπορέσει να πει η εποπτική αρχή ότι πραγματικά έχει τον έλεγχο και δεν είχαμε και τα προβλήματα που υπάρχουν τώρα με διαφορετικές κουλτούρες και διαφορετικές γλώσσες που πρέπει να συμβιβαστούν για να υπάρξει αποτελεσματική εποπτεία. Αν γίνει αυτό εντός της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα είναι πραγματικά ο πύργος της Βαβέλ. Και φοβάμαι και θα δούμε στην επόμενη τραπεζική κρίση κατά πόσο ήταν αποτελεσματική εποπτεία. Για το δεύτερο πυλώνα η έκθεση ζητάει να υπάρξει ένα backstop το οποίο θα πηγαίνει πέρα από τα 550 δισεκατομμύρια ευρώ και ταυτόχρονα προειδοποιεί για τις ε, περαιτέρω κεφαλαϊκές απαιτήσεις από τις τράπεζες. Αυτά δεν ε, συμβιβάζονται ή το ένα ή το άλλο αν το ταμείο είναι πολύ μικρό για την διασφάλιση, πώς είναι δυνατόν να μην χρειάζονται περαιτέρω κεφαλιακές ε, απαιτήσεις. Και μετά η έκθεση προτείνει το backstop να χρηματοδοτηθεί με τα λεφτά του ESM, δηλαδή πάλι με διασώσει τραπεζών μέσω του εθνικού φορολογούμενου. Φοβάμαι ότι δεν έχουμε αντλήσει τα σωστά διδάγματα. Θα πρέπει να είναι δυνατόν να χρεοκοπούν ε, τράπεζες χωρίς ε, χρηματοδότηση του φορολογούμενου. Και δεν ανάγκη να υπάρχει κάποια κρατική ασφάλιση για μεγάλες επιχειρήσεις. Για άλλες επιχειρήσεις δεν υπάρχει αυτό. Και μετά, τρίτον, για το τρίτο πυλώνα, Νομίζω φάνηκε και στις ερωτήσεις που έγιναν στον Λόρδο Χιλ, ειδικά από τους Γερμανούς ε, συναδέλφους, ε, το θέμα της εγγύησης των καταθέσεων. Και με αυτήν είμαστε αντίθετοι, δεν χρειαζόμαστε περαιτέρω κοινωνικοποίηση των κινδύνων, το αντίθετο χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε δημοσιοποίηση των ε, κινδύνων, πρέπει να είναι σαφής οι κίνδυνοι, ποιο τους ανέλαβε και βεβαίω ε, αυτός να αναλάβει και τι ευθύνε του. Το να μετατεθούν ε, οι εθνικοί κίνδυνοι σε άλλα κράτη-μέλη ανταμείβει τα κράτη-μέλη που άσκησαν ε, χειρότερη οικονομική πολιτική ή τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εκείνα τα οποία κινήθηκαν α, λάθος. Και δεν είναι δύσκολο να προφητεύσει κανείς που οδηγεί αυτό το σύστημα. Οπωσδήποτε από γερμανική σκοπιά η κοινο... και κοινοτικοποίηση αυτού του κινδύνου δεν ε, είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική. Σας ευχαριστώ η κυρία Συνδίγουλα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την έκθεσή σας την οποία θεωρώ άρτια, ισορροπημένη. Θα δούμε πώς μπορούμε να επεξεργαστούμε καλύτερα το κείμενο με τροπολογίε. Να επιμείνω σε τρία σημεία και χρονολογικά θα τα πιάσω, δηλαδή όπως τα ε, περιέγραψαν οι προηγούμενοι. Ε, για την Ευρωζώνη, το ευρώ και ότι ίσως πρέπει να έχουμε εργαλεία, να δημιουργήσουμε ίσως και θεσμούς πιο ισχυρούς από αυτούς που υπήρχαν στα κρατημέλη. Όλα αυτά με εκπλήσουν, αλλά το να έχουμε ε, νόμισμα, αστερική αγορά χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, αλλά να μην έχουμε ευρωπαϊκό θεσμό για αυτά, είναι λίγο small economy mindset, αν θέλετε, λίγο περιορισμένη κοντόθωρη νοοτροπία. Και υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Ε, πολλές φορές ε, τα μεμονωμένα άτομα και οι ε, εθνικές αρχές μπορεί να αναπτύσσουν κάποιες σχέσεις συνενοχής και με αυτή την ε, έκθεση και με αυτή την ε, αρχή, την ευρωπαϊκή, νομίζω θα βελτιωθούν αυτά τα πράγματα. Με το level playing field ε, θα πρέπει να βλέπουμε στο σύνολο τα πράγματα, να μην κατακαιρματίσουμε την Ευρωζώνη και την αγορά των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε επίπεδο 28. Αυτό είναι το πρώτο σημείο. να μπορούσαμε να επιμείνουμε λίγο παραπάνω στην έκθεση αυτό. Εάν ο λόγο ύπαρξη ε, του νέου μηχανισμού είναι αυτό, ε, μάλλον κάποιοι δεν το έχουν καταλάβει. Το δεύτερο, διακριτική ευχέρεια. Ε, για την εξουσία του SSM. Ε, πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι αυτό που θέλαμε ε, ήταν οι Ευρωπαίοι επόπτες να έχουν και κάποια μεγαλύτερα περιθώρια εκτίμησης. Θα ήταν καλύτερο αυτό και όχι να καθορίσουμε πάρα πολλούς κανόνες αυτές εξ αρχής οι οποίοι κάποια στιγμή δεν θα έχουν λόγο ύπαρξης. Η χρηματοπιστωτική σταθερότητα, η προληπτική εποπτεία, όλα αυτά είναι σημαντικά θέματα. Μέχρι στιγμής πάντως αυτή η διακριτική ευχέρεια ε, φαίνεται να χρησιμοποιείται σωστά. Τρίτο σημείο για την έκθεση πρωτοβουλίας που έχω και εγώ αναλάβει. Ίσως θα μπορούσατε να πείτε λίγο περισσότερα πράγματα για τη σχέση μεταξύ αυτών που αποφασίζονται σε παγκόσμιο, σε διεθνέ επίπεδο, TILAC για παράδειγμα, η FSB, οι εξουσίε που έχει και να πούμε ότι για μα αυτό ο ενιαίο μηχανισμό είναι η εποπτική αρχή που με τον ένα τον άλλο τρόπο θα πρέπει να έχει μια παρουσία σε παγκόσμιο επίπεδο για να υπάρχει μια μεγαλύτερη συνέπεια και συνεκτικότητα μεταξύ παγκόσμιου και ευρωπαϊκού επίπεδου. Να πούμε λίγο, περισσότερα πάνω σε αυτό. Νομίζω πάντως κύριε Πρόεδρε ότι το πλαίσιο της έκθεσης και των προσεχών εκθέσεων το έχετε καθορίσει με ικανοποιητικό τρόπο και με τα χαράς θα συνεργαστούμε μαζί σας για να βελτιωθεί το κείμενο ακόμη περισσότερο αν βέβαια αυτό είναι δυνατόν. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ ο Τεμάση. Äh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αντικαθιστώ την αρμόδια εισηγήτρια της ομάδας μου. Πρώτα απ' όλα ευχαριστούμε για την έκθεση. Για εμάς έχει μεγάλη σημασία οι τράπεζες να μπορούν να χρεοκοπούν χωρίς ε, κίνδυνο για την ε, χρηματοπιστωτική σταθερότητα και χωρίς να πληρώνουν οι φορολογούμενοι. Το έχουμε πει πολλές φορές. Αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να υπάρξει μια επιτυχής ολοκλήρωση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων των τραπεζών, κατά το οποίο θα θέλαμε να φαίνεται περισσότερο στην έκθεση. Και ίσως θα πρέπει να το τονίσει αυτό το κοινοβούλιο. Όσον αφορά την εποπτεία των τραπεζών υπάρχουν δύο σημεία, το 24 και 25 στα γερμανικά, όπου λέγεται μεταξύ άλλων ότι στο σημείο 25 να υπάρξει διαχωρισμός μεταξύ ρυθμιστικού ρόλου και εποπτείας της αγοράς. Εδώ πέρα είμαστε επιφυλακτικοί όσον αφορά τον εποπτικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, γιατί ως δανειστής τελευταίας καταφυγής έχει αντικρουόμενα συμφέροντα. Και βεβαίως υπάρχουν ούτω ή άλλω και συγκρούσει εντό τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από ό,τι αντιλαμβανόμαστε. Και θα χαιρόμαστε ε, να αναφερθεί αυτό και στην έκθεση. Στο σημείο 24 λέτε πως μέχρι στιγμής η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δίνει επαρκώς λογαριασμό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχουμε διαπιστώσει πως υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά τα έγγραφα τα οποία μπορούμε να τα δούμε μόνο σε κάτι αίθουσες ε, ανάγνωσης και δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για το τι γίνεται παραδείγματος χάρη με συγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Το λέτε αυτό εδώ πέρα κάπως διπλωματικά όταν λέτε πως οι δυνατότητες του Κοινοβουλίου για αξιολόγηση ε, του SSM θα μπορούσαν να βελτιωθούν. Μπορούμε να πούμε πως δεν είμαστε ικανοποιημένοι με την πρόσβαση σε έγγραφα. Επιπλέον θεωρούμε πως είναι σημαντικό πριν μιλήσουμε για αύξηση του, των κεφαλαιακών αποθεμάτων, να δούμε το τι μπορεί να γίνει στην, ε, στον περιορισμό της ε, πληρωμής των μερισμάτων. Τέλος, όταν δίνονται λεφτά του φορολογούμενου, θα πρέπει, ε, κάτι το οποίο βέβαια θέλουμε να αποφεύγουμε, να υπάρχει και ανάλογος κρατικός έλεγχος, είτε με κάποια χρυσή μετοχή ή κάτι τέτοιο. Δεν είναι δυνατόν ο φορολογούμενος ε, μόνο να πληρώνει, αλλά να μην έχει την δυνατότητα να ελέγχει το δημόσιο. Αυτό θα θέλαμε να το δούμε στην έκθεση. Ευχαριστώ. Thank you. Σας ευχαριστώ πολύ, ο Σβέν Γκίγκολτ. Πρώτα απ' όλα, θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή και συμμερίζομαι τις φιλοδοξίες σας με την έκθεση αυτή. Και τι εννοώ με αυτό αντί να ανοίγουμε το παράθυρο για να ακούσουμε διάφορες γνώμες και απόψεις για τη ρύθμιση των τραπεζών και να ξανακάνουμε όλες αυτές τις συζητήσεις ε, τις πολιτικές που είχαμε σε άλλα βήματα συζήτησης και να αποφύγουμε ακόμα χειρότερα γενικότητες για τον ε, ευρώ, νέος και τα λοιπά. Το θέμα είναι πώς ε, θα υπηρετήσουμε τον πολίτη και θα τον υπηρετήσουμε σωστά εάν πραγματικά ελέγχουμε και καθιστούμε υπόλογες τις δομές που έχουμε δημιουργήσει. Αυτός είναι ο στόχος, κατά με. Και νομίζω ότι οι ισχυώδεις εισηγητές μπορούμε να συμφωνήσουμε μεταξύ μα ε, για το τι είναι πολιτική συζήτηση και το τι θα πει ευθύνη, λογοδοσία και απολογισμό ε, του τι έχει γίνει στο προηγούμενο έτο, ε, για παράδειγμα. Συμφωνώ λοιπόν απόλυτα ότι καταρχά πρέπει να πούμε ότι πρόκειται περί επιτεύγματος Πράγματι, ό,τι έχει γίνει αυτό το πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Γνωρίζουμε τους περιορισμούς. Ορισμένοι συνάδελφοι ακροαφηγώς τα ανέφεραν τα σχετικά. Τώρα να δούμε και τα προβλήματα του πραγματικού κόσμου. Σε αυτή την περίοδο, και ίσως εκεί είναι ένα σημείο που πρέπει να το αναπτύξετε λίγο περισσότερο στην έκθεσή σας, έχουμε το ρόλο του επόπτη και τον ειδικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την Ελλάδα συγκεκριμένα. Υπήρχαν πολλά άρθρα στα οποία οι δύο ρόλοι ουσιαστικά συγχέονται. Η ΕΚΤ δηλαδή εντάχθηκε κατά κάποιο τρόπο στους θεσμούς όπως λέγονται και απ' την άλλη ε, δόθηκαν κάποια μηνύματα από τους επόπτες προς τις ελληνικές τράπεζες. Ε, το θεμητό ερώτημα που προκύπτει είναι χρηματοδότηση συνεχίστηκε παρά το ότι εν λόγω τράπεζες ήταν αφαιρέγγες ή σχεδόν αφαιρέγγες. Και πάλι λοιπόν θα πρέπει να μας απασχολήσει ε, και το θέμα της νομισματικής πολιτικής και η σύγκρουση συμφερόντων, η δυνητική σύγκρουση συμφερόντων ε, που ε, αναφέρθηκε σε αυτήν ο Φάμπιο πριν από λίγο. Δεύτερο μείζον ζήτημα, αναλογικότητα. Θα ήθελα να είμαστε πιο ξεκάθαροι. Μέχρι στιγμή τουλάχιστον η Τραπεζική Ένωση στερείται μια σαφούς καθοδήγησης, ενός σαφούς προσανατολισμού. Έχουμε τις αρχές, αλλά όταν φτάνουμε πλέον στον νόμο ε, δεν υπάρχουν τα απαιτούμενα καθεστώτα. Ξεκινάμε με ένα καθεστώς και προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τις μικρές τράπεζες με, το, με τις μεγάλες τράπεζες σαν να είναι το ίδιο ε, μοντέλο. Δεν ισχύει αυτό όμως. Και έπειτα έχουμε τα λογιστικά πρότυπα, τα παγκοσμιολογιστικά πρότυπα. Όταν συγγράψαμε τα, την νομοθεσία για την ΕΚΤΑ, είχαμε μιλήσει ακριβώς για τα ε, πρότυπα αυτά, Ξέραμε ότι έχουν ελλείψεις, αλλά τα χρησιμοποιεί τα πρότυπα αυτά στις ε, πρακτικές ε, πληροφόρησης της ΕΚΤΑ. Αντίστοιχα, θα εφαρμόσουν σύντομα ένα ε, κάπως ε, βαρύ, φορτωμένο ε, σύστημα, το Anacredit, και γιατί θα πρέπει να συλλέγουν πάνω από 100 σημεία δεδομένων για κάθε πίστοση πάνω από 25.000 ευρώ. Δεν ξέρω, ή μήπως εγώ δεν καταλαβαίνω. Δεν έχω καταλάβει πάντως από ό,τι μου εξηγούν γιατί γίνεται αυτό. Γιατί λαμβάνει τέτοια απόφαση η ΕΚΤ και μάλιστα πριν τα συζητήσουμε με την κυρία Σλέγκερ. Όταν λοιπόν λαμβάνουν αποφάσεις πρέπει να έχει προηγηθεί συζήτηση, σοβαρή συζήτηση και στην ομάδα εργασία στην Τραπεζική Ένωση και μετά να λαμβάνονται αποφάσεις. Δεν γίνεται, ε, είναι απαράδεκτο να έχουμε πρώτα δημοσίες στο αποτέλεσμα και μετά να κάνουμε εμείς τη συζήτηση. Δεν έχω επιβεβαίως, προσπαθεί η γραμματεία, το ξέρω. Αλλά μέχρι στιγμής δεν έχω ακούσει τίποτα. Και επίσης είναι σημαντικό, κατά την άποψή μου, οι επόπτες να εξετάσουν και τον κίνδυνο μετατόπισης, μετεγκατάστασης κάποιων επιχειρήσεων σε παράγοντες που δεν είναι εντός εντολής, ε, εντός παιδιόρμοδετών της Τραπεζικής Ένωσης. Έχουμε πιο αυστηρούς κανόνες για την εποπτεία των τραπεζών, έχουμε τις ασφάλειες, αλλά έχουμε και τη σκιώδη τραπεζική. Και θα πρέπει κατά την άποψή μου η Ευρωπαϊκή ε, Αρχή Τραπεζών, η EBA, αλλά και η ΕΚΤΑ e θα πρέπει να αναφέρουν και για τη διάσταση του φαινομένου αυτού μετατόπισης, μετακατάστασης πίσω και να μας δώσουν και προτάσεις. Γιατί δεν είναι δίκαιο το πεδίο ανταγωνισμού και πώς μπορούμε αυτό να το διορθώσουμε. Τέλος. Υπάρχουν προβλήματα υλοποίηση ό,τι αφορά την Τραπεζική Ένωση. Αναφέρατε αρκετά από αυτά τα προβλήματα. Εγώ σε ό,τι αφορά το SRB ε, έχω μια πιο αρνητική εκτίμηση σε σχέση με αυτήν που εσείς ε, περιλαμβάνετε στην έκθεσή σας. Υποτίθεται ότι θα έπρεπε να αναφέρει τακτικά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, για την εξέλιξη της κατάστασης. Δεν ξέρω αν υπάρχουν τέτοιες εκθέσεις. Τις αναφορές εγώ δεν τις έχω δει πάντως και κατά δεύτερον το μηχανισμό στήριξης, το backstop, δεν λειτουργεί σωστά. Αυτός ο μηχανισμός που έχει συμφωνήσει το Συμβούλιο. Τι σημαίνει ότι αν ε, είναι αφαιρέγγια μια τράπεζα και ζητά περισσότερα, απαιτούνται περισσότερα χρήματα, θα πρέπει να επαναχρηματοδοτηθεί από άλλα κράτη-μέλη. Αυτό είναι προκυκλικό, είναι σαφές. Και δεν ήταν αυτή η προσέγγιση μας, η δραματευτική ομάδα. Τέλος. Και με την οδεσία επίπεδου 2 βλέπουμε προβλήματα. Υπάρχουν καθυστερήσεις έχουμε προβλήματα στην υλοποίηση. Και γι' αυτό βέβαια δεν φταίνε οι επόπτε, είναι σαφέ. Φταίνε οι νομοθέτε. Και ιδίω οι κομισιόν. Η υλοποίηση λοιπόν πρέπει να είναι ένα ζήτημα που θα το αναφέρουμε στην έκθεση. Σα ευχαριστώ και πάλι και προσβλέπω και εγώ στη συνεργασία μα. Μάρκο Βάλιν επόμενο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαστε σε κάπως διαφορετική γραμμή κύματος, ε, σε άλλο μήκο κύματο, γιατί ε, το ενιαίο τραπεζικό σύστημα θεωρούμε ότι θα είναι πολύ ευάλωτο και δεν θα μπορεί να εγγυηθεί την αντιμετώπιση σημαντικών ε, σοκ στο τραπεζικό σύστημα. Γιατί όπως είπαν και ορισμένοι συνάδελφοι από την ΚΟΕ και από τους πράσινους, ε, είναι σημαντικό να θεσπίσουμε μια, ε, έναν διαχωρισμό ανάμεσα στην υγιή τραπεζική δραστηριότητα και την ε, λιγότερο βιώσιμη τραπεζική δραστηριότητα που μπορεί δηλαδή να προκαλέσει συστημικά σοκ όπως ας πούμε και το σκαιό, τη σκιώδη τραπεζική όπου δεν υπάρχουν ε, ρυθμίσεις ε, και θα ήταν καλύτερο στην έξεση ίσως να το περιορίσουμε καλύτερα. Ορισμένα παραδείγματα για το πώς η Τραπεζική Ένωση έχει αποδειχθεί ανεπαρκής. Αν αρχίσουμε από το διαφορετικό timing ανάμεσα στο ενιαίο σύστημα εποπτείας και στο ενιαίο σύστημα εξυγίανσης. Έπειτα η διαφορά του συνόλου των τραπεζών που μπαίνουν στο SSM και εκείνων που μπαίνουν στο SRM. Επίσης, οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την σύγκρουση συμφερόντων. Κάτι ακόμα, όπως ε, με την Political Review είδαμε πως ότι τιμωρήθηκαν οι τράπεζες που χρησιμοποίησαν τραπεζικά μέσα για να χρηματοδοτήσουν την πραγματική οικονομία, ενώ οι τράπεζες οι οποίες εμπεριέχουν κάποια προϊόντα που δεν είναι πολύ σαφή ε, και που ενδεχομένως εμπεριέχουν συστημικό κίνδυνο, δεν ε, υπέστησαν καμία επίπτωση. 0,1 ας πούμε η Deutsche Bank ενώ ε, δημιουργεί και άλλο ένα ταμείο το οποίο θα ε, δημιουργείται άλλο ένα ταμείο που θα είναι έτοιμο σε 8 χρόνια. Πλήρησαν επάρκεια ήδη από την ε, διάσωση των Ιταλικών τραπεζών που έγινε την περασμένη εβδομάδα και όπως εκείνες της Φεράρα αυτά αντιστοιχούν την αναφορά στο ενίο ταμείο εξυγίανση για τα πρώτα τρία χρόνια σε οκτώ τελικά και αυτές οι τράπεζες αντιπροσωπεύουν μόνο το 1% των Ιταλικών καταθέσεων. Δηλαδή ένα πολύ μικρό κομμάτι. Θέλω να καταλάβω, για, μάλλον για να καταλάβετε πόσο ευάλωτο είναι αυτό το σύστημα και πόσο δεν μπορεί να εγγυηθεί τη σταθερότητα. Ας προτάξουμε πιο συγκεκριμένα και φιλόδοξα προγράμματα, διαχωρισμό, να εξουδετερώσουμε το συστημικό κίνδυνο και να δημιουργήσουμε ένα τραπεζικό σύστημα το οποίο να μπορεί να προστατευτεί. Γιατί έτσι δυστυχώ θα είναι ευάλωτο το μέσο και στην πρώτη διακύμαση, στο πρώτο σοκ όπω εκείνο του 2009, θα πληρώσουμε όλες τι συνέπειε. Σα ευχαριστώ. Δεν βλέπω κάποιον από την e ΙΕΝΕΦ. Κυμπερβάν Μπερές. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ κύριε Σεγιωτά για αυτή την βάση συζήτηση. Ε, πιστεύω πως είναι μια σημαντική φάση για την Επιτροπή μας για να δούμε πώς λειτουργεί η ε, Τραπεζική Ένωση έχοντας υπόψη μας όλα όσα για παράδειγμα μας λέει ε, ο Ντάνιελ Χιλ όταν έρχεται εδώ για την ανάγκη να συνεχίσουμε να εναρμονίζουμε ή να μειώνουμε τις διαφορές που υπάρχουν στις εθνικές διατάξεις που στόχο έχουν μια εποπτεία κοινή. Εγώ πιστεύω πως οριζόντια σε ένα τέτοιο θέμα θα έπρεπε να ευνοήσουμε μια αξιολόγηση όσον αφορά τον αντίκτυπο της λειτουργίας της προστιθέμενης αξίας των όσων έχουμε ήδη ε, συστήσει για να εξοπλίσουμε τους Ευρωπαίους όταν θα χρειαστεί να συζητήσουν τις συνθήκες ε, έναρξης ισχύω του ΤΙΛΑΚ. Γιατί είμαστε σε μια φάση όπου έχουμε συγκεντρώσει διάφορα πολύ θετικά στοιχεία για μας, αλλά βρίσκω πως αυτό το μέσο που είναι η μελέτη αντικτύπου που χρησιμοποιείται σε ένα σωρό άλλους τομείς, έχω την εντύπωση ότι για τη δική μας επιτροπή μόλις που τολμάμε να το χρησιμοποιήσουμε. Και πολλοί διερωτώνται για το κατά πόσο το τυλάκα μάλλον πώς θα συνδεθεί το τιλάκ με τα όσα ήδη έχουμε κάνει. όσον αφορά τις δυνατότητες δηλαδή του χρηματοπιστωτικού συστήματος να πληρεί τις ε, ε, προδιαγραφές του. Θα πρέπει επίσης να γνωρίζουμε πώς όλα αυτά που θα πρέπει να αρχίσουν να ισχύουν 1η Πρώτου 2016 θα τεθούν σε εφαρμογή. Σημειώνω ότι δεν έχετε πιέσει για τις ημερομηνίε. Μήπως θα πρέπει να υπενθυμίσουμε αυτές τις προθεσμίες. Να εξασφαλίσουμε δηλαδή πως όλα θα είναι εντάξει και να συνεχίσουμε τη δέσμευση που έχουν αναλάβει οι κυβερνήσεις και έπειτα για τον τρίτο πυλώνα Φαντάζομαι πως θα υπάρχουν πολλές τροπολογίες. Ταυτόχρονα δεν θα μπορέσουμε μέσα σε αυτή την έκθεση να προβλέψουμε τη συζήτηση που θα έχουμε επί τη βάση της πρότασης της Κομισιόν της Ιδίας. Και σε αυτή τη φάση, για αυτόν τον τρίτο πυλώνα, το βασικό είναι να θυμίσουμε ότι αυτός ο τρίτος πυλώνας είναι αναπόσπαστο τμήμα της Τραπεζικής Ένωσης και των δεσμεύσεων που αναλήφθησαν από τους όσους συμφώνησαν να προχωρήσουν για τους δύο άλλους πυλώνες με επιτυχία. Και ίσως και να θυμίσουμε ότι η εμπειρία μας έχει δείξει σε σχέση με τους δύο προηγούμενους πυλώνες ότι το να καθυστερήσουμε την νομοθεσία μας οδηγεί στο να την εφαρμόσουμε σε πιο χαοτικές συνθήκες από ό,τι αν είχαμε προβλέψει. Και άρα λοιπόν θα πρέπει να δείξουμε βούληση να κλείσουμε και με την πρόταση της Κομισιόν και ε, να έχουμε ένα πλαίσιο, ένα χρονοδιάγραμμα ώστε η συζήτηση για τον τρίτο πυλόν να μπορέσει και αυτή να ολοκληρωθεί. Thank you. Uh, Ευχαριστώ. Δεν βλέπω κάποιον άλλον ομιλητή. Οπότε καταρχήν να σας ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις και τους συναδέλφους ε, για τις ε, παρεμβάσεις για τις συμβολές σας. Ε, πραγματικά προσβλέπω στη συνεργασία μαζί σας στη διαδικασία τροπολογιών και συμβιβαστικών. Θέλω να τονίσω για μια φορά ακόμα τα όσα είπε και ο Σφένο, ότι δηλαδή και εγώ αυτό προσπαθώ να κάνω. Να κάνω έκκληση σε όλους. Θα έχουμε πολλές ευκαιρίες να συζητήσουμε τα βασικά θέματα πολιτικής και συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις, οπότε δεν πιστεύω ότι χρειάζεται να κάνουμε αυτή την τακτική εργασία που κάνουμε, όπου συγκρίνουμε τις γενικές μας απόψεις. Η προστιθέμενη αξία αυτής της έκθεσης είναι κατά τη γνώμη μου να προσπαθήσουμε να ελέγξουμε όλα όσα μπορούμε να ελέγξουμε, τη δομή δηλαδή που θεσπίζουμε, όπως είπε και ο Σβέν, και ζητώ από τους συναδέλφους αν μπορούν να εστιάσουν από αυτό, γιατί υπάρχουν φυσικά πολλά να πούμε. Είχα και περιορισμό χώρου, οπότε δεν μπορούσα να ε, συμπεριλάβω όλα τα θέματα και οι τροπολογίες από αυτόν είναι πρόσδεκτες. Πιο συγκεκριμένα, η προστασία του τραπεζικού πλουραλισμού είναι κάτι το οποίο τονίζω στην έκθεσή μου και είμαι ευτυχής που συμφωνείτε με αυτό. Φυσικά θα μπορούσαμε περαιτέρω να το διευκρινίσουμε και να το συνδέσουμε με το θέμα που ανέφερε ο Σέν Γίγκολτ για την αναλογικότητα πολλά ίσως στοιχεία θα μπορούσαν να βελτιωθούν ώστε να εξασφαλίσουμε την προστασία του πλουραλισμού ενώ ταυτόχρονα θα εξασφαλίσουμε και ένα ισότιμο ε, πεδίο αλλά και ένα πραγματικό ε, επίπεδο εποπτείας. Αυτό συνδέεται και με ένα θέμα για το οποίο ε, άκουσα και τον κύριο Βάλη που το επικρίνει αλλά είναι κάτι που υπάρχει στην έκθεση. Παράγραφος 21 συγκεκριμένα λέει ότι υπάρχει ανεπαρκής δυνατότητα μέτρησης ε, για διάφορους κινδύνους εκτός από τον πιστοτικό κίνδυνο. Συμφωνώ λοιπόν μαζί σας ότι θα πρέπει να πούμε στον SSM ότι θα πρέπει να είναι σε θέση να μετρήσει όλες τις μορφές κινδύνου. Τώρα, αν αυτό απαιτεί ή όχι διαχωρισμό των τραπεζών και πάλι αυτό είναι μια συζήτηση πολύ χρήσιμη, σημαντική και την κάνουμε σε έναν άλλο τομέα, αλλά δεν νομίζω πως είναι εδώ κατάλληλος ο χώρος, γιατί είναι ένα άλλο θέμα. Δεν πρόκειται για εποπτεία τραπεζών. Βεβαίω ο καθένα είναι ελεύθερο να καταθέσει σχετικέ τροπολογίε, αλλά εγώ νομίζω πω είναι λίγο άσκοπο γιατί εδώ έχουμε ένα νομοθετικό φάκελο για ένα θέμα και είναι άσκοπο να μπούμε και να συζητήσουμε για το ίδιο θέμα στην έκθεση πρωτοβουλία. Το ίδιο ισχύει και για το ΕΝΤΙΣ, όπως συμφωνώ με την Περβάνος Περές, η γνώμη μου είναι, και από ό,τι κατάλαβα δεν συμφωνείτε όλοι με αυτό, είναι ότι ένας κοινός μηχανισμός καταθέσεων είναι σημαντικό στοιχείο της ε, Τραπεζικής Ένωσης και είναι μια γενική αρχή. Και τώρα έχουμε σχετική νομοθετική πρόταση πώς αυτό θα εφαρμοστεί. Και δεν είναι απαραίτητο να κάνουμε την ίδια συζήτηση λοιπόν σε αυτή την έκθεση και πρέπει να πω στο συνάδελφο Βάστορτ ότι δεν εφευρίσκω εγώ την πρόταση για το backstop το να πάμε πίσω είναι απαραίτητο 50 εκατομμύρια. Αυτό αναφέρθηκε στις δηλώσεις του ΕΚΟΦΗΝ στην ανακοίνωση της Επιτροπής για την Τραπεζική Ένωση. Το γεγονός ότι η Τραπεζική Ένωση μπορεί να απαιτήσει ένα κοινό backstop δεν είναι δική μου εφεύρεση. Και είναι ε, νομίζω σκόπιμο να το θυμίζουμε αυτό σε μια έκθεση για την Τραπεζική Ένωση. μπορεί κανείς να πει ότι θα μπορούσαμε να μην το έχουμε. Εάν λειτουργεί καλά το σύστημα εποπτείας δεν θα χρειαστεί να το χρησιμοποιήσουμε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει. Θα μπορούσαμε ίσως αυτό να το αναπτύξουμε περαιτέρω ε, στις τροπολογίες ότι αυτό θα πρέπει να γίνει με τον ε, ESM. Όσον αφορά το bridge financing, συμφωνώ με τις επικριτικές παρατηρήσεις και υπάρχουν ε, βεβαίως επικρίσεις. Μπορούμε, πρέπει να καλωσορίσουμε το γεγονό ότι γίνεται σχετική συζήτηση και μπορεί να γίνει και συμφωνία για το bridge financing. Πάντω, ανάμεσα σε δύο επιλογέ που περιλαμβάνονται στην περίφημη δήλωση του ΕΚΟΦΗΝ, πιστεύω πω η επιλογή του ESM θα ήταν πιο αποτελεσματική ώστε να εξασφαλίσουμε το bridge financing που είναι διαφορετικό από το backstop. Bridge financing είναι πώς θα πάμε μέχρι το 55 όταν το ταμείο δεν είναι έτοιμο, ενώ το backstop είναι αν χρειάζεται να ξεπεράσουμε Με χαρά βλέπω ότι τα όσα περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση της Κομισιόν προχωρούν πάνω κάτω προς την ίδια κατεύθυνση. Φοβούμαι ότι ο τρόπος με τον οποίο ορίζεται ο μηχανισμός είναι και ε, έχει στόχο να μην είναι τελικά πλήρως αποτελεσματικός αυτός ο μηχανισμός και αυτό μπορεί να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα. Τώρα, για την πλήρη εφαρμογή του PRB και της διακυβερνητικής ε, συμφωνίας, από ό,τι φαίνεται προκύπτει συγκεκριμένη προθεσμία, Έχουμε ένα ενίο ταμείο εξυγίασης και η, τα, η συμφωνία σχετική ε, μένει να κυρωθεί. Για τα παρατηρήσει της Συρβή Γκουλάρ συμφωνώ μαζί σας ότι ιδιαίτερα το θέμα της ε, χρηματοπιστωτικής ε, ε, του χρηματοπιστωτικού κατακαιρματισμού είναι σημαντικό και θα πρέπει να αναπτυχθεί καλύτερα και όντως υπάρχουν ορισμένα καλά στοιχεία το πακέτο OND για να μπορέσουμε να υπερβούμε τα στοιχεία του χρηματοπιστωτικού κατακαιρματισμού, ας πούμε απαιτήσεις ε, και απαιτήσει κτλ. Είναι πολύ σημαντικό. Συμφωνώ επίσης ότι θα πρέπει ο SSM να φτάσει στη σωστή ισορροπία ανάμεσα στους κανόνες και τη διακριτική ευχαίρεια σε επόπτης δεν μπορεί αυτομάτως να λειτουργεί ως αυτόματος πιλότος με βάση κάποιους κανόνες αλλά θα πρέπει, κανόνες, αλλά θα πρέπει με διάλογο και κοινή κατανόηση να γίνεται η εποπτεία με βάση τους κανόνες που έχουμε εγκρίνει. Γιατί τόσο τελική παρατήρηση Είπατε ότι 10 χρόνια στη Γερμανία κάναμε να φτιάξουμε τη γενική εποπτεία. Το γεγονός ότι εμείς ένα χρόνο καταφέρουμε αυτό το αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να κάνει την αξιολόγησή μας πολύ θετική, βεβαίως. Δεν είναι τέλειο, αλλά πιστεύω ότι στην έκθεσή μου θα βρείτε μια σωστή ισορροπία όσον αφορά την εκτίμηση του καλό αποτελέσματος και του εκ νέου καθορισμού διαφόρων στοιχείων όπου θα πρέπει να υπάρξουν περαιτέρω βελτιώσεις και διατυπώνω και κάποιες επικρίσεις φυσικά και θα εξετάσουμε στενά τις τροποποιήσεις και θα συνεργαστούμε για να γίνει η συμφωνία όσο γίνεται πιο γρήγορα. Το τίλακ είναι επίσης άλλο ένα ευαίσθητο σημείο που το αναφέρατε. Φυσικά θα το αντιμετωπίσουμε, αλλά είναι καλό που σε αυτή την έκθεση ορίζουμε κάποια σημεία. Είναι περίπλοκο και το να αντιμετωπίσουμε την ευρωπαϊκή ιδιαιτερότητα είναι πολύ σημαντικό για το πώς θα υπάρξει συντονισμός, πώς θα οριστεί στο πλαίσιο της συμφωνίας και βέβαια, συμφωνώ ότι θα έχουμε πλήρως τα δικαιώματά μας ως συν ε, ε, νομοθέτες όταν θα ξεκινήσει η μεταγραφή. Νομίζω πως εδώ μπορώ να σταματήσω. Σας ευχαριστώ και πάλι για τις παρατηρήσεις σας και προσβλέπω τη συνεργασία μαζί σας και στις τροπολογίες σας. Οι ε, προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι η 10 Δεκεμβρίου στις 5 το απόγευμα. Η εξέταση των τροπολογιών στις 11 Ιανουαρίου, η ψηφοφορία εδώ στις 25 Ιανουαρίου και μετά θα δούμε για την Ολομέλη. Εδώ λέει Μάρτιο, αλλά θα δούμε α, μήπως και γίνει και νωρίτερα. Σας ευχαριστώ όλους πολύ λοιπόν και τώρα περνάμε στο επόμενο σημείο. Έκθεση, έκτα, ετήσια έκθεση. Ο εισηγητής είναι ο κύριος Μαριάς, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σήμερα θα συζητήσουμε τις ε, τροπολογίες οι οποίες έχουν ε, κατατεθεί. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές αλλά και, τους, ε, και τη Γραμματεία ε, και όσους συμμετείχαν στην προσπάθεια να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε ε, συμβιβαστικές τροπολογίες. Διότι είναι αλήθεια ότι έχουν κατατεθεί 283 τροπολογίες. Ήδη έχουμε κάνει τρεις συναντήσεις με τους σκιώδεις εισηγητές, τη Γραμματεία και τους Συμβούλους και θα έλεγα ότι έχουμε καταλήξει ε, στο 80% περίπου να συμφωνήσουμε στη διαμόρφωση συμβιβαστικών τροπολογιών. Έχουμε 17 συμβιβαστικές τροπολογίες. Ε, από αυτές υπάρχουν, ε, φαντάζομαι, από ό,τι έχουμε συζητήσει, τρεις-τέσσερες ε, ε τροπολογίες που έχουν ιδιαίτερα προβλήματα και θα ήθελα να ακούσω τις απόψεις των εισηγητών στα ζητήματα αυτά. Υπάρχουν επτά αυτόνομες ε, παρενθέσεις, ε, παρεμβάσεις μάλλον και τις οποίες θα δούμε σε επίπεδο ψηφοφοριών. Είναι 7 παράγραφοι οι οποίοι θα συζητηθούν και επίσης το πρωί με τα ε, recitals λίγος πολύ τα έχουμε συμφωνήσει. Ε, αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα να μπορούμε σήμερα να συζητήσουμε και να καταλήξουμε όσο μπορούμε σε κάποιο κείμενο που ε, και βεβαίως εκφράζει το πνεύμα της ε, έκθεσης αλλά να λάβει υπόψη και τις ε, παρατηρήσεις των συναδέλφων. Να επισημάνω ότι σύμφωνα με την πρόταση που είχα διαμορφώσει ως εισηγητής ήθελα να μείνω στο χρονοδιάγραμμα το οποίο είχαμε δηλαδή να ψηφιστεί το report στα τέλη Δεκεμβρίου του 2015. Γι' αυτό άλλωστε είχα καταθέσει έγκαιρα το report με βάση τις ε, προτάσεις και το χρονοδιάγραμμα της Γραμματείας. Ο κύριος Δράγκη βεβαίως μας ενημέρωσε ότι υπάρχει διαθεσιμότητα δικιά του με βάση την ατζέντα για να γίνει η συζήτηση στην Ολομέλεια και η ψήφιση τον Φεβρουάριο του 2016. Επομένως ε, αυτό που συζητήσαμε και δέχτηκαν και οι, άλλοι σκιώδεις συζητητές είναι να μην έχουμε αύριο την ψηφοφορία επί των ε, τροπολογιών αλλά να πάει σε μια μεταγενέστερη ε, ημερομηνία. Οι ημερομηνίε, κύριε Πρόεδρε, τι οποίε έχουμε, ε, πρακτικά είναι δύο. Η μία περίπτωση είναι η 11η Ιανουαρίου 2016 και άκουσα από εσά ότι θα έχουμε συνεδρίαση στις 11 Ιανουαρίου και θα συζητήσουμε και το report το οποίο παρουσιάστηκε πριν λίγο. Η άλλη περίπτωση ε, εφόσον δεν συμφωνήσουν οι συντονιστές και αυτό θα μπορούσαμε να το δούμε μετά το τέλος της συζήτησης ε, υποχρεωτικά θα είναι η 7η Δεκεμβρίου που σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνουμε μια πολύ συντονισμένη προσπάθεια ούτως ώστε να καταλήξουμε και να έχουμε ε, την ψηφοφορία την άλλη εβδομάδα. σε κάθε περίπτωση τα κεντρικά σημεία τα οποία έχουν, έχει έκθεση νομίζω τα συζητήσαμε την προηγούμενη φορά. Εγώ θα μείνω σε τρία-τέσσερα σημεία. Το πρώτο αφορά τις πολιτικές λιτότητας και είναι δεδομένο ότι οι πολιτικές λιτότητας επέτειναν την κρίση, δεν έδωσαν καμία λύση στα βασικά προβλήματα όπως είναι η αντιμετώπιση της ανεργίας και βεβαίως δεν αντιμετώπισαν και την κρίση χρέους που, υπάρχουν, ε, που υπάρχει σε ορισμένα κράτη και κυρίως ε, στην Ελλάδα όπου το χρέος πλέον δεν είναι διαχειρίσιμο. Το δεύτερο θέμα που φύγει ε, η έκθεση ε, νομίζω είναι η αξιοποίηση του κανονισμού 472 του 2013 που δίνει τη δυνατότητα να εξετάσουν τα κράτη-μέλη για ποιο λόγο έχει φτάσει το χρέος σε τόσο ύψος ε, και ποιες είναι οι αιτίες που οδήγησαν ουσιαστικά στο να φτάσουμε σε αυτά τα αποτελέσματα υπερβολικών χρεών σε διάφορα κράτη-μέλη. Το τρίτο σημείο το οποίο ε, τέθηκε και έγινε συζήτηση και νομίζω θα ακούσω και τις απόψεις των συναδέλφων, είναι να υπάρξει ένα follow-up από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις αποφάσεις που έλαβε το Φεβρουάριο του 2014 για τον έλεγχο της λειτουργίας της Τρόικας και βεβαίως μέρος της Τρόικας όπως ξέρετε όλοι είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εδώ υπάρχει ένα θέμα που το ζητάει η έκθεση να υπάρξει μια ε, ένας τρόπος λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας όπως διαμορφώθηκε και από τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στο ζήτημα αυτό. Επιθυμούμε να υπάρχει διαφάνεια στις σχέσεις Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ένας δημοκρατικός διάλογος και μια λογοδοσία δημοκρατική απέναντι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπως το εξέφρασε και στην τελευταία συνάντηση που είχαμε σε αυτήν εδώ την αίθουσα και ο κύριος το θέμα της ρευστότητα νομίζω ότι είχαμε ένα σημαντικό διάλογο με τους συναδέλφους. Αναφέρεται η έκθεση και ε, στην ε, αγορά στοιχείων ενεργητικού που επιχειρεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με στόχο καταρχάς να ε, φέρει τον πληθωρισμό κοντά στο 2% στις ε, δυνατότητες που πρέπει να υπάρξουν για ρευστότητα στην οικονομία, ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να δανειοδοτηθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να μην υπάρχει απόκληση μεταξύ της ρευστότητας που παρέχεται σε πολύ μεγάλες επιχειρήσεις και στις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, θα έλεγα λοιπόν ότι αυτά είναι τα κεντρικά σημεία τα οποία επεξεργάζεται η έκθεση. Έχω αφήσει εκτός συζήτησης και τελειώνω κύριε Πρόεδρε τα σημεία που είναι επίμαχα για να ακούσω πλέον τις απόψεις των συναδέλφων και κλείνοντας τη συζήτηση να ε, πω και εγώ τις δικές μου απόψεις και τα συμπεράσματα με βάση τις τοποθετήσεις των ε, σκιωδών εισηγητών. Σας ευχαριστώ. Thank you. Uh, on the voting I understand. Ευχαριστώ. 7η Δεκεμβρίου είναι μόνη δυνατή μέρα για να συζητήσουμε την έκθεση αυτή με τον πρόεδρο Ντράγκη. Όσο κατάλαβα και εσείς το γνωρίζετε αυτό. Οπότε θα πρέπει να προσπαθήσουμε να τα καταφέρουμε. Να κάνουμε τη συζήτηση στο τέλος ε, όσον αφορά αυτό το θέμα για να μπορέσουμε να συζητήσουμε πρώτα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, να ευχαριστήσω τον εισηγητή και τους κοιόδης εισηγητές αλλά και τη γραμματεία για την επικοδομητική στάση όσον αφορά την... τις συμβαστικές προτάσεις. Πρέπει να συνεχίσουμε λοιπόν με αυτό το επικοδομητικό πνεύμα και να συμφωνήσουμε σε τροπολογίες που θα βρουν ευρύτατες ε, Πλειοψηφίε. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να καταφέρουμε να μα ακούσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εγώ υποστηρίζω την δομή που έχει έκθεση και θεωρώ πω πολλέ συμβαστικέ τροπολογίε πηγαίνουν σε σωστή κατεύθυνση. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένο με τι ισορροπημένε απόψει που διαμορφώνονται όσον αφορά την κατάσταση τη Ευρωπαϊκή οικονομία, την πολιτική ποσοτική χαλάρωση, τον εποπτικό ρόλο τη κεντρική τράπεζα και την καθημερινή τη λειτουργία. όμω πρέπει να γίνει περισσότερη δουλειά στις συμβαστικές προτάσεις που αφορούν τις μεταρρυθμίσεις και την εξυγίαση των δημοσίων οικονομικών σε πολλά κράτη-μέλη και όσον αφορά τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Τρόικας προφανώς πρέπει να συνεννοηθούμε στις επόμενες συναντήσεις των σκιωδών. Όμως είμαι πεπισμένος πως με την διάθεση που υπάρχει θα μπορέσουμε να βρούμε κάποιες συμβαστικές τροπολογίες που θα τις υποστηρίξει μια μεγάλη πλειοψηφία. Συμφωνώ με την πρόταση του εισηγητή να ψηφίσουμε αργότερα όμως ε, αναμένω να ολοκληρώσουμε τις εργασίες μας τόσο των δυνατόν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Μαυρίδης. Thank you, Chairman. Um, I would like... Uh, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μαριά για την ποιοτική του έκθεση και τις ε, προσπάθειές του να καταλήξει σε κάποιες συμβαστικές λύσεις. Ε, και βεβαίω και τους συναδέλφους ε, και τη γραμματεία. Σχεδόν τα έχουμε καταφέρει, νότι, όχι ακόμα όμως, σχεδόν. Ω σοσιαλιστές και δημοκράτες εμείς ε, έχουμε κάποια σημαντικά ζητήματα τα οποία θα αναφέρω έτσι, σύντομα. Πρώτα απ' όλα. καθώς ε, την προηγούμενη εβδομάδα η Κομισιόν δημοσίευσε την ε, πρότασή τη για ένα ενιαίο σύστημα εγγύηση καταθέσεων, πρέπει να υπάρξει μια αναφορά στην έκθεση. Οι σοσιαλδημοκράτε, ε, επέμεναν εδώ και καιρό, οπότε η ανάγκη να προχωρήσουμε γρήγορα στην ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης, όπως συζητήσαμε πριν από λίγο, με ένα ενιαίο μηχανισμό εγγύησης καταθέσεων πρέπει να αναφερθεί και στην έκθεση. Δεύτερον, για τις συμβαστικές ε, προτάσεις για το υφιστάμενο κενό του ποσοστού χρηματοδότησης μεταξύ μικρομεσαίων επιχειρήσεων και μεγάλων επιχειρήσεων. Εμείς ε, θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει αναφορά στην ανάγκη να προωθηθεί η κοινωνική οικονομία διαφοροποιώντας ε, το ρυθμιστικό περιβάλλον μεταξύ κερδοσκοπικών και μη κερδοσκοπικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Επί τη ευκαιρία το είχα ξεκαθαρίσει αυτό κατά τη διάρκεια των συζητήσεων και να πω πως αύριο οργανώνω μία εκδήλωση και είστε όλοι προσκεκλημένοι για αυτό το ζήτημα ακριβώς. 4 η ώρα αύριο. Για το συγκεκριμένο αυτό ζήτημα λοιπόν για το ρυθμιστικό περιβάλλον κερδοσκοπικών και μη επιχειρήσεων. Μετά, για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Εμείς θεωρούμε πως είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό καθώς παραμένουν ακόμα τεράστιο πρόβλημα σε ολόκληρη την Ένωση. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, 10 κράτη-μέλη και 6 μέλη της Ευρωζώνης έχουν ποσοστά μη εξυπηρετούμενων δανείων πάνω από το 10% των συνολικών δανείων και ε, σε κάποιες χώρες φτάνουμε το 45%. Ένας μηχανισμός λοιπόν για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια πρέπει να υπάρξει σε κάποια προβληματικά κρατημέλη όπως στην Κύπρο, όπως έγινε σε Ισπανία και Ιρλανδία για να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα. Θεωρούμε πως πρέπει να στηριχθεί μια τέτοια τροπολογία και είναι σημαντικό να συμπεριληφθεί στην έκθεση. Τέλος, θεωρούμε, και δεν χρειάζεται νομίζω να πω πολλά γι' αυτό, είναι θέση των σοσιαλδημοκρατών πως οι πολιτικές λιτότητας δεν είναι η λύση για να αντιμετωπίσουν τα τη μελη το βάρος του χρέους. Όσον αφορά το χρόνο διάγραμμα για τις ψηφοφορίες, συμφωνούμε. Νομίζω εδώ πέρα δεν έχει υπάρχει πρόβλημα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον εισηγητή. Πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε υπόψη ε, και παρότι αναβλήθηκε το είπατε και εσείς η ψηφοφορία, θα τα καταφέρουμε. Υπάρχουν λοιπόν πράγματα που πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Πρόκειται για μια έκθεση που αφορά το έργο ενός άλλου θεσμικού οργάνου και δι της Δεν είναι και αμεληταίος αυτός ο φορέας, εφόσον είναι αρμόδιος ε, για την νομισματική πολιτική και έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα και αυτό το στοιχείο θα πρέπει να το έχουμε κατά νου. Θα πρέπει ταυτόχρονα να μπορούμε να εξηγούμε ανεξάρτητα και αυτόνομα τι πιστεύουμε, αλλά ταυτόχρονα να παραμένουμε σε μια συμβαστική γραμμή μεταξύ των πολιτικών ομάδων, γιατί είναι μια έκθεση από ένα θεσμικό όργανο για ένα άλλο θεσμικό όργανο, όχι ενό εισηγητή μια συγκεκριμένη πολιτική οικογένεια και επειδή ξέρουμε να, κάνουμε, να, να ερχόμαστε σε συμβιβασμό θα το πετύχουμε πιστεύω και αυτή τη φορά. Καλό θα ήταν να εστιάσουμε όμως πιστεύω στα ουσιώδη της έκθεσης ε, και να αποφύγουμε τη διασπορά. Ε, πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, θα έχει μια ισχυρή θέση εάν μπορεί με τοποθέτησή του να συγκεντρώσει μια ευρεία πλειοψηφία του επανσυνάδελφου του ΕΛΚ και πιστεύω ότι ίσως ε, ορισμένοι θα χρειαστεί αυτά που έχουν πει αυθορμήτως κάπως να τα μετριάσουν κατά κάποιο τρόπο. Η ομάδα Άλντε θα συνεισφέρει όσο μπορεί. Απλά να πω ότι πρέπει να έχουμε υπόψη μας γιατί ακριβώς πρόκειται δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι ουσιαστικά διακυβεύονται οι σχέσεις μας με την ΕΚΤ. Πρέπει να είμαστε αξιόπιστοι. Πρέπει να κάνουμε λογικές προτάσεις και με αυτόν τον τρόπο ενισχυόμαστε ως θεσμός. Δεν θα ε, ρυθμίσουμε τους λογαριασμούς μας, ούτε θέλουμε να εκφράσουμε μειονοτικές απόψεις. Ευχαριστώ. Thank you, um, Chair, and Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ τον εισηγητή <clears throat> και τους κοιόδης για την εργασία τους. Θέλω να αναγνωρίσω ότι ο εισηγητής ήταν εξαιρετικά ε, πρόθυμος να εξασφαλίσει όσο γίνεται ευρύτερη συνένεση. Δυστυχώς για αυτή την έκθεση που αφορά την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ο πολιτικός συμβιβασμός πολύ συχνά είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί, διότι ορισμένοι από εμά έχουμε πολύ διαφορετική άποψη για τον ρόλο που παίζει η έκτοτε στην εσωτερική οικονομική πολιτική τα τελευταία χρόνια. Και θα με έχετε ακούσει να το αναφέρω αυτό τακτικά εδώ σε αυτή την αίθουσα. Και επίσης γνωρίζετε πόσο, πολλά, πόσο πολύ πιστεύω ότι υπάρχουν διαρθρωτικά προβλήματα στη λειτουργία της ΕΚΤ και στη λογοδοσία της. Και, το Πολλές φορές έχω πει ότι η ΕΚΤ λειτουργεί υπό την πίεση διαφόρων μεγάλων πολυεθνικών και επίσης ε, πολύ συχνά καθορίζουν τη φορολογική τους πολιτική με βάση την προσέλκυση τέτοιων ομίλων, ιδιαίτερα όσον αφορά το εκτιμώντας F, ποσοτική χαλάρωση που δεν είναι απαραίτητο προβληματική, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με θετικό και προοδευτικό τρόπο και αν χρησιμοποιηθεί με αυτόν τον τρόπο μπορεί να είναι χρήσιμο χρήσιμη και να εξυπηρετήσει την πραγματική οικονομία. Μόνο όμω όταν υπάρχει πραγματική πολιτική βούληση για να γίνει κάτι τέτοιο και εγώ έχω πολλέ αμφιβολίε όσον αφορά το συγκεκριμένο, τη συγκεκριμένη συμβιβαστική, ενώ αναγνωρίζω ότι οι συγκητής και άλλοι έχουν ε, προσπαθήσει πολύ για να εξασφαλίσουν όσο γίνεται ευρύτερη συνένεση. Υπάρχουν αρκετοί τομεί όπου πιστεύω πρέπει να ε, το εξετάσουμε περισσότερο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μαριά για την έκθεσή του. Αυτό που θέλω να πω ε, καταρχήν είναι ότι πρέπει να αποφύγουμε αυτή τη φορά αυτή η έκθεση να είναι μια άσκηση ρουτίνας. Ε, θα ήταν σφάλμα, λεμόντας υπόψη τι έγινε πέρυσι σε σχέση με την ΕΚΤΑ και ότι και το δικαστήριο έπρεπε να διορθώσει κάποια ζητήματα, αυτά που έγιναν στην Ελλάδα. Ήταν μια έκθεση ρουτίνα. Υπάρχουν ε, σημαντικά ζητήματα, ουσιώδη ζητήματα που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση και θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μαριά γιατί τις είχε συμπεριλάβει πολλέ από αυτέ τι βασικέ θέσει ε, στο αρχικό σχέδιο έκθεση ε, και ήμασταν σύμφωνοι. Τώρα βέβαια χρειάζεται να γίνει μέγιστη προσπάθεια και να βασίζεστε σε εμά, τη δική μα πολιτική ομάδα, για να μην υπάρξει ε, κάπως πιο ήπια διατύπωση, να μην ε, μετριαστεί ε, η το, να μην μετριαστούν αυτά τα σημεία, γιατί πρέπει να παραμείνουν κατά την άποψή μα. Όπω για παράδειγμα, ότι έχουμε ένα ζήτημα νομικού πλαισίου σε ό,τι αφορά τη δράση τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, νομισματική διάλογη. Πολλοί από αυτού που γίνονται εδώ, σε αυτήν την αίθουσα και με τον Τράγκη κάποιες φορές ε, αφήνει και να εννοηθεί ότι από τις ε, ε, αποφάσεις του Δικαιωτικού Συμβουλίου πολλές φορές γίνονται με διακριτική ευχέρεια, πολύ μεγάλη διακριτική ευχέρεια και αυτό δεν είναι σωστό, όπως επίσης για το τι έγινε στην Ελλάδα. Η παράγραφος 25 για μένα είναι πάρα πολύ σημαντική. Αν δεν μπούμε τίποτα για το τι έκανε η έξι σχέση με την Ελλάδα, δεν έχει νόημα να συντάσσουμε τέτοιου είδους εκθέσεις. Ε, γιατί αυτό αφισβητεί, αυτό που έγινε δηλαδή, και βασικά στοιχεία ε, που αφορούν τη λειτουργία της τράπεζας και εμείς νομίζω ότι πρέπει να αποφανθούμε και θα ήταν ε, σφάλμα μας να διαγραφεί, να απαλληφθεί αυτή η παράγραφος 25. Πρέπει να δούμε τι έγινε με πολλές αποφάσεις που ελήφθησαν για την Ελλάδα. Ότι είχε υπάρξει συντονισμός, είχαν γίνει συναντήσεις και στο πλαίσιο της Ευρωομάδας, του Eurogroup. Μα πού είναι τελικά η ανεξάρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ε, απέναντι σε τέτοιες ε, καταστάσεις. Αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να τα αφηνεύσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πρέπει να αποφαίνεται από αυτόν. Και ε, κάποια άλλα ζητήματα που θεωρώ πολύ σημαντικά. Πρώτον, εμείς είχαμε πει ότι ήταν πολύ κακή ιδέα το SSM να είναι υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο αποπτικός μηχανισμός. Το είδαμε και τους τελευταίους μήνες δημιουργήθηκε σύγχυση μεταξύ του τι είναι επόπτης ε, και ε, τι είναι ο φορέας που εκτελεί. Τελικά ήταν ένα mission impossible αυτό που έγινε. Κύπρος, Ελλάδα, έχουμε πολλά παραδείγματα. Επίσης, σε ό,τι αφορά τα μη συμβατικά μέτρα εμπορική πολιτικής. Ε, καλό είναι και το αναφέρει η έκθεση και χαίρομαι γι' αυτό ότι φυσικά ήταν απαραίτητα αυτά τα μη συμβατικά μέτρα ε, της νομισματικής πολιτικής, ε, συγγνώμη, νομισματικής, όχι εμπορικής πολιτικής, ε, είδαμε τι αντίκτυπο μπορεί να έχουν αυτά όμως τα μέτρα αν διατηρηθούν μακροπρόθεσμα και αυτό θα πρέπει να το αναφέρει η έκθεση. Εδώ θα σταματήσω. Είναι κάποια από τα σημεία αυτά που σας είπα, τα οποία θα ήθελα να περιλαμβάνονται, αλλά κυρίως το μήνυμα που θέλουμε να δώσουμε είναι ότι δεν είναι μια έκθεση ρουτίνας, είναι μια σημαντική χρονιά, εξαιρετική χρονιά και πρέπει να αναφέρουμε τα ουσιώδη και ένα μπράβο στον κύριο Μαριέ γιατί τα αναφέρει πολλά από αυτά τα σημαντικά. Thank you, Marco Valli. Ευχαριστώ Μαρκο Βάλλη και εγώ ευχαριστώ τον εισηγητή γιατί ήταν πολύ δύσκολο να ε, βρούμε συμφωνία σε μία τόσο ε, δύσκολη έκθεση γιατί έχουμε πολλές διαφορετικές πολιτικές ιδεολογίες στον οικονομικό τομέα. Είναι πάντοτε δύσκολο να βρεθούν οι συμβιβαστικές και όταν βρεθούν είναι πράγματα τα οποία ποτέ δεν ικανοποιούν όλους απολύτως. Στο εσωτερικό λοιπόν της έκθεσης υπάρχουν στοιχεία σημεία για την οικονομική διακυβέρνηση, για ολόκληρο το πακέτο των διορθωτικών μεταρρυθμίσεων, το ΕΦΣΥ, την, και την Ένωση των Κεφαλαιογορών. Ε, δεν τα βλέπουμε αυτά με πολύ θετικά, γιατί ακριβώς στις συμβιβαστικές έχουν τονιστεί πολιτικές θέσεις που ακολουθούν διαφορετική πορεία από τις δικές μας θέσεις. Όμως θα πρέπει να πω την αλήθεια, υπάρχουν μέσα σε αυτή την έκθεση πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, τα οποία μπορούμε να στηρίξουμε. Με αρχή γενομένης από το γεγονός ότι οι πρόσφατες μετρήσεις εκτάκτων των πολιτικών ήταν ανεπαρκής και ε, στην έκθεση αυτή το αναφέρουμε γιατί δεν επιλύθηκε το πρόβλημα της ε, πίστοσης ούτε της πραγματικής οικονομίας. Ε, λύθη ίσως το πρόβλημα κάποιων τραπεζών. Αλλά και αυτό θα φανεί. καλή είναι η συμβιβαστική που κάνει σωστή επικρίση στο σύστημα του ευρώ και αναφέρεται στο γεγονό ότι οι φορολογικές προσαρμογές και οι πολιτικές λιτότητες δεν συνέβαλαν παρά στην τελμάτωση και στην ύφεση. Έπειτα πολύ καλές είναι οι παράγραφοι που αφορούν το διαφάνεια και τη μεγαλύτερη δημοκρατική νομιμότητα, ιδιαίτερα όσον αφορά το ρόλο της ΕΚΤ. Εντό της Τρόικα είδαμε πως στη διάρκεια της ε, Ελληνική κρίση υπήρχαν ε, στοιχεία, υπήρξαν στοιχεία που έπρεπε όντως να τονιστούν. Υπάρχουν λοιπόν πολύ πιο ευρεία θέματα πολιτικού χαρακτήρα που είναι πολύ δύσκολο να βρούμε συνένεση και όπου δεν συμφωνούμε, αλλά για πολλά άλλα θέματα συμφωνούμε. Γιατί πραγματικά τονίζονται ζητήματα που μέχρι σήμερα δεν έχουν ποτέ εξεταστεί σε μια τέτοια έκθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρείω τον εισηγητή και βέβαια να του ευχηθώ καλό κουράγιο για την συνέχεια γιατί δεν θα είναι τόσο απλά τα πράγματα. Το ευρώ και η νομισματική πολιτική από ό,τι φαίνεται πως ε, είναι όπως και η μεταναστευτική κρίση άλλωστε κάποια σημεία στα οποία κάποιες ομάδες ε, ε, θέλουν ε, να μην συνεισφέρουν καθόλου επικοδομητικά. Οι ομάδες αυτές της ε, πλειοψηφίας οι οποίες δεν θέλουν να συνεισφέρουν επικοδομητικά στο μέλλον της Ένωσης. Έτσι όπως έχουν τα πράγματα λοιπόν δεν πάει αρκετά μακριά η έκθεση παρά το ότι υπάρχουν κάποιες καλές συμβαστικές προτάσεις ΕΛΚ, Σοσιαλδημοκράτες και Άλτε δεν θέλουν να δουν την ε, αλήθεια για τον ρόλο της Ευρωπαϊκής ε, Κεντρικής Τράπεζας και για το ότι παρανόμως ε, αγόρασε δημόσια χρέη. Αναφέρομαι εδώ πέρα στην τροπολογία 83. Βεβαίως μπορούμε να γνώμε την πραγματικότητα αλλά δεν μπορούμε ποτέ να γνώμε τις συνέπειες που έχει αυτό. Κάτι το οποίο από ό,τι φαίνεται οι συνάδελφοι δεν το αντιλαμβάνονται ακόμα. Βλέπουμε λοιπόν πως οι τροπολογίες του ΙΕΝΕΦ και του ΙΕΦΤΕΝΤΕ δεν είναι αυτές οι οποίες ε, δίνουν τον ε, τόνο και δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να στηρίξουμε τελικά την έκθεση αυτή, αλλά βεβαίως ε, υπάρχει ακόμα χρόνος και μπορεί τελικά να μπορέσουμε να έρθουμε πιο κοντά σας. Ευχαριστώ. Thank you, Σας ευχαριστώ, κύριε Σύκτης. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τους σκιώδεις συζητητές ε, για τις τοποθετήσεις τους και να πω έχουμε ορισμένα θέματα που πρέπει έτσι λίγο να τα βάλουμε σε μια σειρά. Πρώτα απ' όλα υπάρχει συμφωνία ως προς τη δομή της ε, έκθεσης και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το δεύτερο είναι ότι όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να πετύχουμε τις αναγκαίες συνενέσεις προκειμένου να μπορέσει αυτή η έκθεση να γίνει αποδεκτή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να ψηφιστεί. Και να ψηφιστεί μάλιστα με αυξημένη πλειοψηφία, διότι είναι μια έκθεση η οποία κρίνει στο μέτρο των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την ε, λειτουργία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε μια φάση η οποία ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, αφορού, υπήρχε η, το το ζήτημα της Ελλάδας αλλά και άλλα θέματα τα οποία απασχόλησαν την τράπεζα. Και ως εκ τούτου θα πρέπει να υπάρχει μια τοποθέτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στα θέματα αυτά διότι δεν είναι δυνατόν να έχουμε μια έκθεση ρουτίνας χωρίς να θίξει τα θέματα τα οποία πραγματικά απασχόλησαν ε, το 2014 την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Κατά την έννοια αυτή υπάρχει η παράγραφος 25 που αναφέρεται στον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας απέναντι στην Ελλάδα. Έχω ακούσει απόψεις από τους σκιώδεις εισηγητές, αλλά σε κάθε περίπτωση κατά την άποψή μου πρέπει τα θέματα να τεθούν. Βεβαίως ο στόχος είναι να έχουμε μια αυξημένη πλειοψηφία και στήριξη σε αυτή την έκθεση, ώστε να υπάρχει και το αντίστοιχο μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ιδίως σε θέματα οικονομικής διακυβέρνησης Ιδίω όσον αφορά τι σχέσει τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τη δημοκρατική λογοδοσία η οποία χρειάζεται να υπάρχει εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και επισημαίνω για άλλη μια φορά ότι σε αυτήν εδώ την αίθουσα πριν λίγε μέρε ο κύριος Δράγκη αναφέρθηκε ξεκάθαρα στις σχέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ότι ο ίδιος έρχεται εδώ σε αυτή την αίθουσα προκειμένου να μας ενημερώσει αλλά να αναλάβει ταυτόχρονα υπόψη και τις απόψεις των ε, Ευρωβουλευτών. Ε, υπάρχουν σημεία τα οποία φυσικά πρέπει να δει κανείς, το ρόλο της Τρόικας, το ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ως μέλος της Τρόικας, ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων που υπάρχουν στη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ως νομισματική αρχή, ως εποπτική αρχή και αυτά είναι θέματα τα οποία οπωσδήποτε η έκθεση πρέπει να τα θίξει. Και σαν πρώτη εισήγηση όταν έγραψα αυτή την έκθεση έθεσα τα θέματα αυτά με σαφήνεια, αποσκοπώντας πάντοτε στη συζήτηση και φυσικά στο να καταλήξουμε σε κοινέ θέσεις που όπως είπαν πάρα πολλοί δεν είναι εύκολο διότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, διαφορετικές ιδεολογίες, διαφορετικές κατευθύνσεις. Σε κάθε περίπτωση θα γίνει προσπάθεια να ενσωματωθούν οι διάφορες σκέψεις, να υπάρξουν οι κατάλληλοι συμβιβασμοί. Είναι δεδομένο ότι θα πρέπει να αναφερθούμε και στα κόκκινα δάνεια, όπως είπε ο συνάδελφος, ε, από το S&D διότι τα κόκκινα δάνεια είναι σημαντικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή και για την Ελλάδα και για την Κύπρο και για ορισμένες άλλες χώρες. Πρέπει να υπάρξει ρύθμιση, δεν πρέπει οι άνθρωποι να χάσουν τα σπίτια τους, να βγουν τα σπίτια ε, των ε, οικογενειακών στο σφυρί. Ε, αυτά τα θέματα νομίζω ότι θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε και παραμένω στη διάθεση των συναδέλφων. Τώρα κύριε Πρόεδρε απευθύνομαι σε εσά σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα. Ε, από ό,τι έχω πληροφορηθεί υπάρχει μια απόφαση των ε, coordinators να μην γίνει ψηφοφορία ε, στις 11 ε, Ιανουαρίου παρότι θα έχουμε συνεδρίαση. Ε, εάν θέλουμε και εγώ επιθυμώ να γίνει συζήτηση της εκθέσεως και να ψηφιστεί τον Φεβρουάριο σύμφωνα με το πρόγραμμα τότε έχουμε δύο θέματα τα οποία σας τα αναφέρω και μετά την συνεδρίαση μπορούμε να τα δούμε μαζί σας και με τη γραμματεία. Η μία περίπτωση είναι πράγματι να έχουμε την ψηφοφορία στις 11 Ιανουαρίου αφού θα γίνει η συνεδρίαση. Η δεύτερη περίπτωση είναι να την έχουμε την ψηφοφορία στις 7 Δεκεμβρίου. Ε, αυτό νομίζω ότι μπορούμε να το αφήσουμε ανοιχτό να το συζητήσουμε μαζί σας μετά την συνεδρίαση και να λάβουμε υπόψη και το τι λένε οι συντονιστές. Σε κάθε περίπτωση τελειώνοντας, εάν είναι να πάμε σε ψηφοφορία στις 7 Δεκεμβρίου, σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνουμε μια πάρα πολύ εντατική δουλειά ε, αυτή την εβδομάδα με τους σκιώδεις προκειμένου να διαμορφωθεί η voting list την 5η το απόγευμα. Γι' αυτό λοιπόν θα σας παρακαλούσα να λάβετε υπόψη το ενδεχόμενο να πάμε σε ψηφοφορία στις 11 Ιανουαρίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you. Uh, um, Εγώ σας ευχαριστώ. Δυστυχώς ε, είναι σαφής η απόφαση των συντονιστών που δεν μας επιτρέπει να ψηφίσουμε τον Ιανουάριο συγκεκριμένη ημερομηνία. Ένας γενικός κανόνας αυτός, δυστυχώς μπορούμε να τον αλλάξουμε. Επομένως, ε, όπως είπαμε, στην τελευταία συνεδρίαση των συντονιστών υπήρχε αναβολή κατά μια εβδομάδα, αλλά δεν μπορεί να επιμηκυνθεί αυτή η αναβολή. Είναι μια έκθεση για το 2014, την ψηφίσουμε το 2016. Δεν έχουμε άλλη ημερομηνία, ε, έχουμε και τον κύριο Τράγκη. Είναι σημαντικό νομίζω να είναι παρόν για την έκθεση αυτή, άρα θα πρέπει να γίνει 7 Δεκεμβρίου. Είμαι βέβαιος ότι από τεχνικής πλευράς είναι εφικτό το ίδιο και από πολιτικές πλευράς. Αυτή λοιπόν ημερομηνία 7 Δεκεμβρίου ψηφίζουμε. Σας ευχαριστώ πολύ όλους και όλες. Και δίνω τώρα στον Φάργκους Φέρμπερ την Προεδρία. Σας ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Έχουμε ακόμη δύο σημεία στην ημερήσια διατάξη που μέσα σε 25 λεπτά θα πρέπει να τα διεκπαιρεώσουμε. Ε, εκτός αν θέλουν να παραμείνουν οι διερμηνείς. Πάμε λοιπόν ε, στο 7 προς μια νομοθετική πράξη για την ενιαία ψηφιακή αγορά. Θα δώσω το λόγο στον Ρενάτο Σόρου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να τα πω γρήγορα. Γιατί λέτε ότι έχουμε καθυστερήσει. Ε, να τα πω στα Ιταλικά όμως καλύτερα. digital single market. Έχουμε να κάνουμε με την ενιαία ψηφιακή αγορά. Ci occupiamo adesso del digital single market e dare il parere della nostra comunità. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε γνωμοδότηση ως Επιτροπή για την ε, ενιαία ψηφιακή αγορά και θεωρώ πως είναι ένα από τα πιο σημαντικά προγράμματα και σχέδια της Επιτροπής μας αυτή τη θητεία. Η ενιαία ψηφιακή αγορά ασχολείται με το να μπορέσουμε και στον ψηφιακό τομέα να φτάσουμε σε μια ενιαία ευρωπαϊκή αγορά. Έχουμε λοιπόν ενιαία αγορά για ένα σωρό από τα πράγματα που ε, κατασκευάζουμε και πουλάμε, αλλά είμαστε, είμαστε πίσω όσον, άφερε, όσον αφορά τα άειλα αγαθά και αυτό μας κάνει να συνειδητοποιούμε και την καθυστέρηση με την οποία συχνά οι θεσμοί ε, αντιμετωπίζουν και επιλύουν ε, Ε, τα θέματα που απασχολούν τον κόσμο που αλλάζει τόσο γρήγορα. Εμείς έχουμε ε, μια, ε, τη γνώμη μας για όλα αυτά, αλλά και εμείς της Επιτροπής ΕΚΟΝ πρέπει να γνωμοδοτήσουμε γιατί έχουμε τη γνώμη μας όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη, την ανάπτυξη γενικότερα και την απασχόληση. Ε, καταλήξαμε νομίζω σε έναν καλό αριθμό συμβιβαστικών που ελπίζω πως ε, αύριο θα μπορέσουν να εγκριθούν με μεγάλη πλειοψηφία αν και ε, κάποια σημεία παραμένουν, παραμένει διαφωνία ή μάλλον κάποια σημεία θα έπρεπε να υπογραμμιστούν καλύτερα όπως για παράδειγμα η δυνατότητα να προωθήσουμε περαιτέρω την ε, εμπορία μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας των ε, πολιτιστικών αγαθών. 124 τροπολογίες περίπου κατατέθηκαν ε, μεγάλο ενδιαφέροντος τροπολογίες και μπορώ να τις συνοψίσω σε κάποιους τίτλους, ας πούμε, ανάπτυξη οικονομική. Είναι προφανές ότι η οικονομία έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια ότι η βιομηχανία ψηφιακή έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ γρήγορα και κάποιες φορές μάλιστα ε, με ηλικιώδεις ρυθμούς έχουν δημιουργηθεί νέες βιομηχανίες, νέα συστήματα. Κάποιες επιχειρήσεις έχουν φτάσει λόγω του αριθμού των συμμετεχόντων αλλά και λόγω του τζίρου των κερδών τους έχουν φτάσει στις πρώτες θέσεις στην παγκόσμια αγορά. Η Κομισιόν εκτιμά ότι μια ψηφιακή μετάβαση της ευρωπαϊκής οικονομίας και της ευρωπαϊκής κοινωνίας θα μπορούσε να επιφέρει ωφέλη περίπου 415 δις ετησίως, ένα τεράστιο νούμερο και αυτό είναι ωφέλη όσον αφορά, και ωφέλη όσον αφορά την απασχόληση 3,9 εκατομμύρια νέες θέσεις απασχόλησης, θέσεις απασχόλησης καλές, βιώσιμες και που αφορούν όχι μόνο τον τομέα της καινοτομίας, ε, της ε, startup, αλλά και την ψηφιακή μεταποίηση, στο πιο παραδοσιακό μεταποιητικό τομέα, αυτό που ονομάζεται μετάβαση προς μια ε, βιομηχανία 4,0. Επίση επαναλαμβάνω και αυτή τη μετάβαση, τη, μετάβαση στην ψηφιακή που θα πρέπει να συνοδευτεί από τα απαραίτητα κεφάλαια, να στηριχθεί από τα απαραίτητα κεφάλαια για την καινοτομία αλλά και για την μετάβαση και να συνοδευτεί επίση από στήριξη για την ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων. Δεν αρκεί να έχουμε ένα μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων που είναι σε θέση να γράφουν κωδικούς, άρα δηλαδή να κατακτήσουμε ειδικού, αλλά θέλουμε να υπάρξει μια πολιτιστική μετάβαση στην ουσία. Δηλαδή να κατακτηθεί ένα νέο είδος αλφαβητισμού από πλευράς κάθε Ευρωπαίου πολίτη. και να μπορέσουμε με κάθε τρόπο να στηρίξουμε τη δυνατότητα της δημιουργίας μιας μεγάλης ευρωπαϊκής υποδομής για υπερευρίας, υπερευρίας ζώνης. Είναι ανάγκη να προωθηθεί η σύγκληση των χωρών και των ευρωπαϊκών λαών και να μην δημιουργήσουμε, να μην προκαλέσουμε περαιτέρω ε, ρήξη, να καλύψουμε αντίθετα το ψηφιακό χάσμα. Οι πράσινοι μάλιστα τονίζουν ότι η πρόσβαση στο ίντερνετ θα έπρεπε να θεωρείται ένα κοινό αγαθό τεράστια σημασία, το οποίο θα πρέπει να ευνοείται με κάθε δυνατό τρόπο. Τονίζουμε και το θέμα των νέων θεμελιωδών δικαιωμάτων και προσθέτουμε ένα χάρτη δικαιωμάτων του ίντερνετ. Ε, η συζήτηση, ε, μάλλον ένα, μια άλλη δέσμη τροπολογιών αφορά την ανταγωνισμό. Γνωρίζουμε όλοι πως η Κομισιόν αντιμετωπίζει το θέμα της υπόθεση Google. Η Κομισιόν πρόσφατα ξεκίνησε μια πρωτοβουλία μια ευρεία διαβούλευση για να καταλάβουμε το ρόλο και τους κινδύνους που περιέχονται στις νέες μεγάλες ε, πλατφόρμες του ίντερνετ. Μάλιστα, αυτός ο ψηφιακός κόσμος ε, διανύει δύο νέα φαινόμενα που ίσως ο κόσμος ε, της παραδοσιακής μηχανίας δεν τα έχει αντιμετωπίσει. Δηλαδή το γεγονός ότι ε, πέρα από την ανάπτυξη μιας υπηρεσίας φτάνουμε να έχουμε περιθωριακό κόστος ε, ίσο με μηδέν. Οπότε μπορεί να όλοι οι ανταγωνιστές να συμμετέχουν Πρέπει να προστατευτεί λοιπόν για να παρακολουθεί το ανταγωνισμό, να ευνοηθεί η διαρκή παρουσία μεγαλύτερου ανταγωνισμού και για αυτέ τι νέε αγορέ είναι, τόσο, είναι πολύ σημαντικό αυτό και ίσω και μάλιστα εγώ πιστεύω πω οπωσδήποτε πρέπει να μεριμνήσουμε για την προστασία του ανταγωνισμού η οποία δεν ε, ε, γίνεται ακόμα με κατάλληλο τρόπο, θα πρέπει να ευαθυνθεί. Ε, κάτι ακόμα σημαντικό είναι η φορολόγηση. 28 διαφορετικά φορολογικά συστήματα, διαφορετικά συστήματα ΦΠΑ για παράδειγμα, δημιουργούν εμπόδιο στην ανάπτυξη. Ναι, και κλείνω. Δημιουργούν λοιπόν φραγμούς για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, που είναι μεγάλο κομμάτι της οικονομίας μας. Κάτι ακόμα σημαντικό. που ίσως να μην το έχουμε όμως καταλάβει πλήρως, είναι η οικονομία η οποία βασίζεται στα δεδομένα και τη χρήση αυτών. Αυτές είναι οι παρατηρήσεις μου. Εγώ ε, κλείνω έτσι. Υπάρχουν ενδιαφέρουσες συμβιβαστικές και ελπίζω πως αύριο θα έχουμε μεγάλη πλειοψηφία. Ε, ευχαριστώ όλους τους κοιόδους που εργάστηκαν με μεγάλη επιμέλεια και βούληση για εξέβρεση κοινών θέσεων σε αυτό το σημαντικό τομέα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Δίνω τον λόγο στους κύριους για το ΕΛΚ Καλπέλτ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Κύριο Πρόεδρε να ευχαριστήσω τον εισηγητή και για την διάθεση που είχε για συμβιβασμούς. Δεν θέλω τώρα να τα αναφέρω όλα αυτά, τα έχουμε συζητήσει. Θα ήθελα μόνο να αναφερθώ σε πιο προβληματικές συνδυαστικές προτάσεις. Ε, αυτή η ΕΦ, παραδείγματος χάρη για ένα αρμονισμένο ΦΠΑ. Οπωσδήποτε συμφωνώ με τον εισηγητή πως ε, η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση μπορεί να χαρακτηριστεί από μειωμένα εμπόδια και θεωρώ πως αυτό το οποίο ζητάει ο εισηγητής για ένα απλοποιημένο σύστημα ΦΠΑ στο διαδίκτυο είναι κάτι το υπερβολικό και δεν είναι ακόμα οικονομική πραγματικότητα. Δεν φαντάζομαι πως το ίδιο προϊόν έχει διαφορετικό ΦΠΑ ανάλογα με το είδος αγοράς. Αν γίνεται κάτι, αν αγοράζεται κάτι στο διαδίκτυο ή όχι. Γι' αυτό εμείς δεν υποστηρίζουμε αυτό το κομμάτι και δεν μπορούσαμε να συνεννοηθούμε μέχρι στιγμής που ε, να πείσω τον εισηγητή να αντικαταστήσει τη λέξη εναρμονισμένο με τη λέξη συντονισμένο. Εμείς χαιρόμαστε για το ότι καταλήξαμε σε μια πρόταση μετά από όλες αυτές τις ε, συζητήσεις ε, όσον αφορά και τους φραγμούς στην είσοδο στην ψηφιακή οικονομία. Συμφωνούμε ότι πρέπει να μειωθούν, αλλά Βεβαίως ε, κάποια πράγματα είναι προ όφελο του Ευρωπαίου πολίτη. Δεν μπορεί κάποιος να ανοίξει τράπεζα χωρίς ε, τις απαραίτητες εγγυήσει. Ε, το ίδιο ισχύει και για ταξιδιωτικά πρακτορία κτλ. κτλ. Είναι μεγάλος ο κατάλογος. Εν ολίγης, στηρίζουμε τις συμβαστικέ προτάσεις πλην τη συμβαστική πρόταση F και σε κάποιες περιπτώσεις ε, ζητάμε χωριστές ε, ψηφοφορίες. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω να το δεχτεί ο συγητής τις χωριστές ψηφοφορίες και να αντικαταστήσει όπως είπα τη λέξη εναρμονισμένο με το συντονισμένο στη συμβαστική πρόταση για να μπορέσουμε να τη στηρίξουμε και αυτήν. Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία. Ευχαριστώ. Όπως είπα έχουμε δύο εκθέσεις ακόμα ε? Ναι. και 15 λεπτά από το ECR δεν βλέπω την κυρία Σουίνμπερν. Φιλελεύθερου, δεν βλέπω τον κύριο Τόρβαλτς. Από τον Κούε όμω κάποιον βλέπω, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, θα ήμασταν τον πιο σύντομα. Θέλω να ευχαριστήσω και πάλι ε, εισηγητή Σκιώδη ε, και να πω ευθύ εξ αρχή ότι φυσικά οι ψηφιακέ υπηρεσίε ε, υπέρ του Περλόνους και τα λοιπά, αναγνωρίζουμε ότι θα πρέπει να διατίθενται πιο άμεσα, ιδίω σε μικρομεσαίες επιχειρήσει και πολύ μικρέ επιχειρήσει. αλλά υπάρχουν και κάποια ζητήματα για τα οποία έχω σοβαρέ ανησυχίε και σε ό,τι αφορά τι συμβαστικέ προτάσει όσο το τον πιο σύντομα για το D. Καλώ ορίζει νέο κεφάλαιο αγορών που είναι ένα συμπλήρωμα στην αγορά ψυχικών υπηρεσιών και στη σχετική στρατηγική κτλ για να τα πούμε μια πρόταση από προσανατολίζει και για το ε. Επίσης προβληματική συμβαστική πρόταση που λέει ότι το φορολογικό πλαίσιο που ισχύει δεν μπορεί να συνεχίσει να εφαρμόζεται δεδομένα των ιδιαιτεροτήτων τη ψηφιακή οικονομίας και ακούσαμε να λέει και ο εισηγητή ε, τι ζητήματα ε, προκύπτουν ε, με, διαφορετικού με διαφορετικούς 29 κτλ. Ε, δεν πρέπει να απονομευτεί όμω η φορολογική εθνική κυριαρχία με τέτοιου είδου εκθέσει. Είναι ένα τομέα, ο ψηφιακό τομέα, που έχει αναγκαστεί να υπερπηδήσει του κόσμου τα εμπόδια για να μπορούμε να πάμε στο γραφείο μας, να ανοίγουμε την οθόνη και να βλέπουμε στο σπίτι του, στην οικογένειά μας, εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά. Ή για να αγοράζουμε με δύο-τρία ε, πατήματα ενώ κουμπιού, ε, εισιτήρια για συναυλίες σε όλο τον κόσμο κτλ. Δεν νομίζω ότι αυτοί οι οποίοι ε, ενταργάζονται στον τομέα αυτό δεν θα μπορέσουν να περιπηδήσουν τα εμπόδια που έχουν να κάνουν στους φορολογικούς τελείς κτλ. Είναι γελία αυτά τα πράγματα. Δεν θα το στηρίξω λοιπόν αυτό. Δεν μου αρέσει η κατεύθυνση που παίρνει η έκθεση. Δεν θα μπορέσω να την υποστηρίξω. Ευχαριστώ πολύ. Μιχαλ για τους πράσινους. Ευχαριστώ. Εμεί μπορούμε να στηρίξουμε την έκθεση, είμαστε ικανοποιημένοι. Πραγματικά προσπάθησε να βρει συμβαστικές λύσεις ο εισηγητής, κατά την απόψή μου. Βλέπουμε εδώ πέρα πως έγιναν προσπάθειες να υπογραμμιστεί ότι το ίντερνετ και η εσωτερική αγορά είναι μια υποδομή για την κοινωνία και βοηθούν τη συνολική οικονομική ανάπτυξη. Αυτό αναφέρεται σε πολλά σημεία και δεν είναι μόνο πλέον έκτημα για κάποιους λίγους. Πηγαίνει σωστή κατεύθυνση Τρεις προτάσεις έχουμε ακόμα, θα τις στείλουμε γραπτές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Μάρκο Βάλλη, δεν το βλέπω όμως. Μπάρμπαρα Κάπελ για το ENF, ούτε αυτήν την βλέπω. Η κυρία Περές ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στρέφουμε στον εισηγητή κυρίως, στο ΕΛΚ όμως. Σε ό,τι αφορά τη συμβαστική ΕΦΑ. Το ΕΛΚΑ δεν θα στηρίξει από ό,τι κατάλαβα αυτή τη συμβαστική πρόταση που όμως υπερβαίνει και τα δέοντα. Με ποια έννοια. Ποιο θέμα πραγματεύεται αυτή η συμβαστική τροπολογία. Το αν θα αντιμετωπίσουμε με τον ίδιο τρόπο, με ισότιμο τρόπο, ένα πολιτισμικό αγαθό, αν είναι ψηφιακό ή αν είναι σε έντυπη μορφή. Λέμε ότι θέλουμε να προωθήσουμε μια ψηφιακή οικονομία Πώς λοιπόν τιμωρούμε τα πολιτιστικά αγαθά που βρίσκονται σε ψηφιακή μορφή. Συμβαστική F λάθος ε, υποστηρίζει ή μάλλον πολύ σωστά λέει ότι τα κρατη μπορούν να έχουν μικρότερο φορολογικό για αυτά τα πολιτιστικά αγαθά. Όμως ποιο είναι το πρόβλημα. Το δικαστήριο θεωρεί ότι ένα βιβλίο, από τη στιγμή που είναι ηλεκτρονικό, e-book, δεν αποτελεί πολιτιστικό αγαθό. Επομένως, Έχουμε μια δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εναρμονίσει και να επιτρέψει μια μείωση ε, του ΦΠΑ στα ηλεκτρονικά βιβλία, στα e-books. Η Κομισιόν δεσμεύτηκε γρήγορα να καταθέσει πρόταση για τη μείωση του ΦΠΑ στα e-book. Πούμε, μια διατύπωση πολύ μετριοπαθή που δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα που δημιουργήθηκε τι αποφάσει του δικαστηρίου. Κρίμα, κρίμα. Ελπίζω με τη στήριξη του ΕΛΚ λοιπόν μέχρι αύριο να μπορέσουμε να διορθώσουμε αυτή τη συμβιβαστική ΕΦ και να βρούμε μια διατύπωση που θα είναι πιο ισχυρή και θα έχει και σχέση με την πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Αλλά νομίζω πως η ε, ώρα για <laughs> διαπραγματεύσει είναι πολύ λίγη, γιατί αύριο ψηφίζουμε. Ο εισηγητής θέλει να πάρει το λόγο για 1,5 λεπτό maximum. No, Io interverrò Όχι. 30 δευτερόλεπτα μόνο. 30 δευτερόλεπτα μόνο, Πρόεδρε. Να σας εξηγήσω ότι μιλάμε για την ενιαία ψηφιακή αγορά για 16 λεπτά. Αν αυτή είναι η προσοχή που αξίζει αυτή, αυτό το θέμα και αυτό δίνει η, αυτή η Επιτροπή σε ένα τέτοιο ζήτημα, ε, τότε καλή τύχη. Με συγχωρείτε, λέει ο πρόεδρο. Δεν, δεν παραβίασα εγώ το χρονοδιάγραμμα. Είχαμε τη συζήτηση για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που τράβηξε λίγο παραπάνω. Περιμένω να το σέβεστε, λέει ο κύριο Σιγητής. Τέταρτη φορά ήταν ε, κοιτάξτε, υπήρχε χρόνος που είχε προβλεφθεί στην ημερήσια διάταξη. Ακόμα και αν δεν σε ενδιαφέρει το θέμα. Ο πρόεδρος, ε, επιτρέψτε μου να πω δύο λόγια. Κοιτάξτε, ε, είχαμε καθυστέρηση 20 λεπτών από τη συζήτηση για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δεν μπορώ, δεν έφταιγα εγώ, ήταν δική μου ευθύνη, μου έδωσε την Προεδρία ο πρόεδρο. Αλλά και οι διερμηνεί κάποια στιγμή πρέπει να σχολάσουν. Αυτό πρέπει να λύσω. Και αυτό προσπάθησα να κάνω. Να μην κατηγορείτε εμένα όμως, ε, δεν είμαι εγώ υπεύθυνο. Λοιπόν, ψηφοφορία αύριο. Περνάμε στο σημείο 8 ε, της έκθεση για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ο κύριος Παπαδημούλης δεν είναι εδώ, αλλά ο κύριος ε, Κάρτη θα παρουσιάσει την έκθεση σε 2,5 λεπτά. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Παπαδημούλης συζητά συγγνώμη, δεν πρόλαβε να πάρει το τρένο σήμερα από το Παρίσι. Μάλλον το τρένο είχε πρόβλημα στο δρομολόγιο. Ήθελε να ευχαριστήσει τους ηγητές για τη συνεργασία τους. Συνεργάστηκαν πάρα πολύ καλά τις προηγούμενες εβδομάδες. Προσπάθησαν λοιπόν να καταλήξουν και προσπάθησε ο κ. Παπαδημούλης να σεβαστεί όλες τις απόψεις, να τις ενσωματώσει στις συμβιβαστικές προτάσεις και θεωρεί πως κατάφεραν να το κάνουν αυτό. Η έκθεση αυτή είναι αποτέλεσμα δύο πολύ επικοδομητικών συνεδριάσεων των ε, εισηγητών και υπήρχε ένας αρκετά μεγάλος βαθμός ε, συνένεσης. Η γνωμοδότηση καλωσορίζει το ότι περιλαμβάνεται το 6,93% στο πλαίσιο του δανεισμού την αύξηση αυτή κατά 6,93% στο δανεισμό της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και θεωρεί πως θα πρέπει να επανεξεταστεί η αύξηση κεφαλαίου της ε, τράπεζας. Δυστυχώς το 2013 οι συνολικές επενδύσεις μειώθηκαν σε σχέση με την εποχή προκρίσης και υπάρχει μια ανισορροπία επενδύσεων και θεωρεί πως ε, εξακολουθεί να είναι μεγάλη πρόκληση εξευρεστές ενεργασίας. Υπάρχει επίσης πρόβλημα πρόσβασης ε, στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ζητά την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να ξαναδεί το πρόγραμμά της ε, των επενδύσεων και να επενδύει σε έργα τα οποία έχουν μεγάλη οικονομική και κοινωνική σημασία και θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε χώρες που έχουν υψηλή ανεργία και κενό στις επενδύσεις για να προωθηθεί η κοινωνική συνοχή. Η έκθεση τονίζει την ανάγκη να λειτουργεί η ΕΦΣΑ με τρόπο διαφανή σύμφωνα με τα κριτήρια του κανονισμού της θεωρούμε πως θα πρέπει επίσης να δοθεί ιδιαίτερος ρόλος στην εντοχή της αγοράς εργασίας ειδικά εκεί όπου υπάρχουν κενά επενδύσεων λόγω του περιβάλλοντος υψηλού κινδύνου. Για τα θέματα φορολογίας συζητείται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να εγκρίνει μια πιο επίκαιρη και υπεύθυνη πολιτική φορολογίας και να μην συνεργάζεται με εταίρους που είναι αποδεδειγμένα αρνητικοί και να λάβει υπόψη τον κίνδυνο της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος και κάποια άλλα πράγματα κύριε Πρόεδρε αν μου επιτρέπετε ζητάει η τράπεζα να αξιολογήσει τις ΣΔΙΤ όσον αφορά το αποτέλεσμα στις θέσεις εργασίας και την προσθέμενη αξία για την κάθε οικονομία και κοινωνία. Ε, επειδή ο χρόνος πιέζει δεν θα πω τίποτα άλλο. Ε, και πάλι ο εισηγητής ευχαριστεί όλους τους σκιώδες για την διαδικασία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Περνάμε τώρα στους σκιώδες. Τόμας Μάν για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ. Δεν φταίει ο πρόεδρος, να το πω και εγώ, για την καθυστέρηση. Ε, έχουμε έναν κατάλογο εδώ πέρα που δεν έχει μεγάλη σχέση με την πραγματικότητα. Από το α μέχρι το ω. Κοίταξε, υποτίθεται πως ε, συνεργαζόμαστε όλοι μαζί και όχι μόνο η γκουε και η Πράσινη. Θα ήθελα να μπορέσουμε να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες, αλλά δεν γίνεται να δουλέψουμε έτσι. Ως ε, υποστηρίξαμε κάποιες ε, συμβαστικές ε, προτάσεις γιατί ήταν αρχικά τελείως αρνητική η έκθεση. Έχει αλλάξει πράγματι η οικονομική κατάσταση, αυτό είναι αλήθεια. Ε, πράγματι υπήρχαν σημάδια οικονομικής ανάκαμψης, ναι. Αλλά αν δεν μπουν αυτά τα πράγματα στην έκθεση θα πρέπει να την καταψηφίσουμε. Πρέπει να αλλάξουν λοιπόν κάποια πράγματα γιατί Υπάρχουν στοιχεία που δεν έχουν ούτε μία σχέση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αλλά με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που θα ήθελε να γράψει μια έκθεση ο συγγητή, επίση μιλάτε για συγκεκριμένε χώρε ότι έχουν έλλειψη επενδύσεων, μα και αυτό δεν έχει σχέση με την εντολή τη έκθεση. Γι' αυτό σε πολλά σημεία ζητήσαμε χωριστέ ψηφοφορίε και χαίρομαι που συμφωνούν μαζί μα και οι άλλε ομάδε. Οπότε αύριο θα έχουμε πάρα πολλέ χωριστέ ψηφοφορίε. Αλλιώ δεν γίνεται να συμφωνήσουμε την έκθεση. Ευχαριστούμε κύριε Μαν. Μαρία Ζωά Ροντρίγκε για τους Σοσιαλδημοκράτες. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομη. Να πω ότι η ομάδα μας υποστηρίζει τις, τις συμβιβαστικές που προτείνεται και θα ήθελα να θυμίσω ότι εισήγαμε προφορικές τροπολογίες όσον αφορά την, ε, όσον αφορά την αναφορά στους φορολογικούς παραδείσους. που προτείνουμε να εντοπίζονται όχι μόνο από τον ΩΣΑ, αλλά και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό μόνο. Σας ευχαριστώ. ECR, Stanislav, Όζοκ. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, θα προσπαθήσω να είμαι όσο γίνεται πιο σύντομος. Ε, δεν χρειάζεται να με μαλώσετε με το σφυρί. Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τη δουλειά τους μέχρι στιγμής. Ε, θέλουμε να στηρίξουμε την ε, ε, έκθεση. Συμβιβαστικέ Α, Β και Γ δικοτοπτήσουν την οικονομική πραγματικότητα της Ένωσης αλλά και του κόσμου γενικότερα. Θα πρέπει να υπογραμμίσουμε το ρόλο των ε, βιώσιμων ιδιωτικών επενδύσεων για τις μικρομεσαίες, το F και το G δεν μπορούμε να το στηρίξουμε διότι υπάρχει πρόβλημα περαιτέρω σύγκληση. Όπως έχει πει ο συνάδελφος, καλωσορίζουμε την των ψηφοφορία ε, και θα μπορέσουμε έτσι να υιοθετήσουμε σωστέ θέσει. Σα ευχαριστώ εξ ονόματο των φιλελευθέρων. Ευχαριστώ για του φιλελεύθερου κ. Σάιξατ. Άλλον συνάδελφο αντικαθιστώ, αλλά δεν έχει σημασία. Α, για του φιλελεύθερου δεν βλέπω. Τώρα λοιπόν περνάμε στου πράσινου. Τώρα έχετε το λόγο. Ναι, ναι, συγγνώμη που σα είπα ελεύθερο. Ναι. Ίσως να μπορώ να πω και κάτι Quest Να πω ότι η Μόλι δεν μπορούσε να είναι εδώ. Στηρίζει τι συμβασικέ προτάσει ε, που έχουμε καταρτήσει. Είναι καλέ οι προτάσει για τους φορολογικούς παραδείσου αλλά και τα σχετικά με την πράσινη μετάβαση. Οι επενδύσεις δηλαδή να πηγαίνουν στα κοινωνικά ομόλογα και στα πράσινα ομόλογα. Τα στηρίζουμε αυτά. Βέβαια, έχουμε για αύριο μια προφορική τροπολογία γιατί πιστεύουμε ότι δεν είναι επαρκώ επαρκώς σαφή τα ονόματα ε, Volkswagen. Δεν θα πρέπει να τη δανείζει η ΕΚΤΑ αφού φαίνεται ότι κάνουν ε, κατάχρηση των ε, χρημάτων που παίρνουν, θα κάνουν μια προφορική τροπολογία. Μα ανησυχεί επίση ε, ότι έχουν ζητηθεί κάποιε χωριστέ, μάλλον κατά τμήματα ψηφοφορία, για του φορολογικού παραδείσου και τι και επενδύσει, επενδύσεις. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να παραμείνουν στην έκθεση, ιδίω αν θέλουμε να μιλήσουμε για πράσινε επενδύσει. την ίδια μέρα που έχουμε την έναρξη τη διάσκεψη για το κλίμα στο Παρίσι τέτοιου είδου συμβασμοί πρέπει να παραμείνουν. Αλλιώ θα ξανασκεφτούμε τι θα ψηφίσουμε. Μέχρι στιγμή τη στηρίζουμε την έκθεση με αυτέ τι συμβαστικέ προτάσει και ευχαριστούμε και τον εισηγητή για τη δουλειά του. Ο πρόεδρο, ευχαριστώ πολύ. Η FDD Μάρκο Βάλλη. Σα ευχαριστώ πολύ σύντομα. Να πω ότι συνεργάστηκα πολύ καλά με τον εισηγητή της ΓΟΕ και μπορέσαμε να πετύχουμε καλές συμβαστικές, ειδικά όσον αφορά την αύξηση των επενδύσεων στην έρευνα και την ανάπτυξη της ε, ΕΤΕΠ και τις επενδύσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν πρόβλημα δανεισμού λόγω της έλευσης επενδύσεων από πλευράς του παραδοσιακού τραπεζικού τομέα. Συμφωνούμε επίσης ε, για την παράγραφο που ξαναπαναξετάζει τις δυσκολίες ε, στις χώρες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, δηλαδή χάσμα ανεργίας ε, και μεγάλων επενδύσεων. Και επίσης το κομμάτι που μιλάει για τις ε, τους φορολογικούς παρανδύσους. Είναι απαραίτητο η Τράπεζα Επενδύσεων να έχει έναν ορίζοντα ανοιχτό προς ε, τι αρχέ τη ε, κοινή λογική, δηλαδή να μην χρηματοδοτεί επιχειρήσει που λειτουργούν σε αυτέ τι χώρε και που να μην χρηματοδοτεί παρά μόνο έργα βιώσιμα. Για την υποδομή, για την έφηση, όσον αφορά τέτοιου είδου χρηματοδοτήσεις θα πρέπει να προσέχουμε να είναι υποδομές που είναι φιλικές ε, προς το περιβάλλον και να μην επενδύουμε σε αυτοκίνητα ας πούμε που εξακολουθούν να ρηπαίνουν με διοξείδιο του άνθρακα. Ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω την κυρία Κάπελ από το ΕΦΕΝ και δεν βλέπω να ζητά κανεί άλλο το λόγο. Να σας ενημερώσω μόνο πως έχουμε μια, ένα νέο κατάλογο ψηφοφοριών σύμφωνα με τις συστάσεις κάποιων συναδέλφων και έχουν μοιραστεί ε, απόψε ε, στις 4 περίπου. Ελπίζω θα τα βρείτε λοιπόν στα γραμματοκιβώτιά σας. Θέλετε να ξαναπάρτε λόγο να σας ευχαριστήσω εσάς, τους κοιόδες και τους διερμηνείς για την ε, υπομονή τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε αύριο. τέλος συνεδρίασης. 10 και μετά θα έχουμε ψηφοφορίες. Ευχαριστώ και τις υπηρεσίες μετάφρασης.